Αλλάξαμε. Ε, η κανονικά η αλλαγή στην έναρξη των συνεδριάσεων για το απόγευμα έπρεπε να ισχύει από τη νέα κοινοβουλευτική θητεία. Γιατί βλέπω ότι δεν ε, συνηθίσαμε όλοι στο 2,5. Πολλοί νομίζουν ακόμη ότι ξεκινάμε στις 3 και έρχονται με το πάσο τους. Γι' αυτό χρειάστηκε να καθυστερήσουμε κάπως κι εμείς περιμένοντας να έρθουν όλο και περισσότεροι βουλευτές, αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Οι α, μας ζήτησαν να μας διαβάσουν πάλι ένα μήνυμα, γι' αυτό παρακαλώ φορέστε τα ακουστικά σας για να ακούσουμε το μήνυμα των δερμηνέων. Βρισκόμαστε στην τρίτη εβδομάδα κινητοποιήσεων λόγω τη εργασιακή διένεξη με τη διοίκηση για τι συνθήκε εργασία μα. Σε ορισμένε καμπίνε έχουν επιστρατευτεί όλοι οι διερμηνεί και είναι υποχρεωμένοι να εργαστούν.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 δημόσια μας συνεδρίαση. Έχει ήδη ανάψει πρώτη διαφάνεια. Έχουμε μαζί μας ε, τον Επίτροπο Αντριού και τον καλωσορίζουμε θερμότατα στην ε, συνεδρίαση της Επιτροπής. Ε, είχαμε πολύ καιρό να σας δούμε κύριε Αντριού Δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά που σας είχαμε στην Επιτροπή. Χαίρομαι πάντως που μας ήρθατε και πάλι. Ποιο είναι το θέμα της σημερινής ανταλλαγής απόψεων. Δεν είναι μόνο ένα, είναι πολλά και διάφορα. Έχουμε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Θα μιλήσουμε για την υγεία των φυτών, για την υγεία των ζώων, την καλή μεταχείριση των ζώων, την ασφάλεια των τροφίμων, ε, τα νέα μέτρα φυτοπροστασίας ε, και της καταπολέμησης των επιβλαβών οργανισμών των φυτών, το θέμα της προστασίας των, των ζώων κατά τη μεταφορά, το νέο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά, για τον οποίο μάλιστα η συγγετής μας είναι ο κύριος Ντόρφμαν από τους συντηρητικούς μεταρρυθμιστές. Ε, και αυτό γίνεται σε συνεργασία με τις Επιτροπές Μεταφορών και περιβάλλοντος, αν θυμάμαι καλά. Μάλιστα έγινε προσπάθεια να συσταθεί και ειδική εξεταστική επιτροπή. Τελικά καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι εμείς είμαστε η αρμόδια επιτροπή και πιο γρήγορα θα διεκπαιρεώσουμε το ζήτημα. Πάντως όλοι είμαστε υπέρ υψηλών προδιαγραφών ε, για την καλή μεταχείριση των ζώων και κατά τη μεταφορά και καλό θα ήταν. Να μην έχουμε ε, μεταφορά των ζώων σε μακρές αποστάσεις, μακρές αποστάσεις από το σφαγείο. Πάντως θα πρέπει να βελτιώσουμε τις συνθήκες ε, για τη μεταφορά των ζώων. Είπαμε θα μιλήσουμε και για την ασφάλεια των τροφίμων, τη σχέση με τις τρίτες χώρες. Όπως ξέρετε, μια αντιπροσωπεία της ε, Επιτροπής μας μετέβη στη Βραζιλία και εκεί είχαμε επαφές ε, και με την ε, Γενική Διεύθυνση Υγείας, την οποία ευχαριστούμε θερμά γιατί κάποιοι, κάποια μέλη της Γενικής Διεύθυνσης Σάντε συμμετέχουν τακτικά και μας ενημερώνουν και στις συνεδριάσεις μας. Οπότε κύριε Επίτροπε θα σας δώσω πρώτα το λόγο για να μας κάνετε την παρουσίαση, μετά θα δώσω το λόγο στους συντονιστές για σχόλια και ερωτήσεις και μετά τις απαντήσεις σας στους συντονιστές θα έχουμε γενική συζήτηση με τους υπόλοιπους βουλευτές. Επειδή έχουμε ήδη μείνει λίγο πίσω στο χρόνο, σας θέλω παρακαλώ να προχωρήσουμε αμέσως. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη. Αυτή η διάλογη είναι σημαντικές συζητήσεις και γόνιμες. Μας επιτρέπουν να μετρήσουμε την πρόοδό μας και να προβληματιστούμε για σημαντικά θέματα ε, τα οποία ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της ε, προηγούμενης χρονιάς. Πολύ δε περισσότερο αυτές οι συζητήσεις ε, είναι απόδειξη της συνεργασία μας προς ένα κοινό στόχο, να διατηρήσουμε τις, τα υψηλότερα δυνατά επίπεδα ανθρώπινης υγείας, υγείας των ζώων και των φυτών, ευημερία και ευζοία των ζώων και ασφάλεια των τροφίμων. Σα ευχαριστώ που με καλέσατε. Θέλω να αναφερθώ επί ευκαιρία σε διάφορα θέματα που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα την Επιτροπή σα, του Ευρωπαίου πολίτε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επειδή όμως έχετε συζητήσει αυτό το θέμα πρόσφατα, θα ήθελα να αρχίσω ευστώντας στην προσοχή ε, στο πρόσφατα εγκριθέντα εφαρμοστικό κανονισμό για εθελοντικές ενδείξεις προέλευσης στην επισήμαση των τροφίμων. Ποιος είναι ο στόχος αυτής της νέας νομοθεσίας. Είναι απλός. Εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες για την προέλευση του βασικού συστατικού δεν θα εξαπατούν τον καταναλωτή. Είναι σαφή τα κριτήρια ε, τα οποία εξασφαλίζουν ίσους κανόνες για τον κλάδο και βελτιώνουν την κατανόηση των καταναλωτών. Όπως γνωρίζετε, τα κράτη-μέλη έχουν κοινοποιήσει εθνικά μέτρα για δεσμευτική και υποχρεωτική σήμανση σε σχέση με την προέλευση για κάποια συστατικά ορισμένα. Κράτη-μέλη θα στείλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκθεση για τη λειτουργία και αντίκτυπο αυτών των μέτρων σε εσωτερική αγορά. Στη συνέχεια θα τα αξιολογήσει όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κατά πόσο έχουν πραγματικό αντίκτυπο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυστηρή νομοθεσία για την ασφάλεια ε, των τροφίμων και την υγεία των ζώων και των φυτών. Ε, ωστόσο, έχουμε και ε, νοσήματα των ζώων και των φυτών. Και πολλοί αγρότες όπως και εσείς ε, ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να γίνει ε, και παίρνουν τα μέτρα τους. Εμείς όμως θα πρέπει να έχουμε μία απάντηση συντονισμένη στατηγική όσο και ταχεία. Στην περίπτωση της ξυλέλα ε, έχουν υιοθετηθεί αυστηρά μέτρα και στη συνέχεια ενημερώθηκαν ανάλογα με τις εξελίξεις για να προστατεύεται η επικράτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε όμως παρόλα αυτά να έχουμε ταχύτερες διαδικασίες παντού σε όλα τα κράτη-μέλη. Αντίστοιχα, η συνεχιζόμενη και έμονη παρουσία της αφρικανικής πανόλης του χείρου είναι πολύ σοβαρή απειλή παντού σε όλα τα κράτη-μέλη για τη χειροτροφία και όχι μόνο για τα κράτη που πλήττονται από τα συγκεκριμένα κρούσματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει αυστηρές ε, ρυθμίσεις για το περιορισμό της μεταφοράς ζώντων χείρων και των προϊόντων τους και συνεχίζονται συζητήσεις και σε διεθνές επίπεδο για να ε, διαβεβαιώσουμε και και να καθησυχάσουμε τους εμπορικού μας εταίρους. Επίσης, οι τοπικές κοινωνίε θα πρέπει να συμμετέχουν με ανοιχτό και ειλικρινή διάλογο με όλους τους ενδιαφερομένους για να γίνονται ε, καλά και ομαλά οι έλεγχοι και στι δύο περιπτώσεις. Ε, ιδιαίτερα όταν έχουμε κάποια μέτρα τα οποία δεν είναι δημοφιλή, όπως η αποκοπή τη ουρά των χειριδίων. Ε, είναι πολύ σημαντικά επίσης ε, τα θέματα αυτά και θα πρέπει να ενημερώνονται και οι κυνηγοί, ιδιαίτερα για την Αφρικανική Πανόλη του Χείρου. Πρόσφατα ε, είδαμε το Μάρτιο στη Σόφια την συνεδρίαση που οργάνωσε η Βουλγαρική Προεδρία. Δεν γνωρίζουν σύνορα οι επιδημίες ούτε οι επιζώτιες. Γι' αυτό είναι δική μας ευθύνη και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ημών ως μελών της Επιτροπής σας να ενημερώνεται το κοινό ότι είναι για το κοινό καλό αυτές οι ε, αντιδράσεις. Αλλιώς θα έχει σοβαρές επιπτώσεις αυτό για τη γεωργία, την υγεία των ζώων και την οικονομία μας. Η αφρικανική πανόλη του χείρου λοιπόν θα πρέπει να ελεγχθεί και είναι σημαντικό αυτό και υπάρχει χώρος για βελτίωση. Άλλο παράδειγμα, η απάτη στα τρόφιμα. Πέρυσι είχαμε την κρίση του Φιπρονίλ που χρειάστηκε να ελέγξει και να δοκιμάσει όλα τα συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, τα διδάγματα που αντλήσαμε μα δείχνουν ότι είναι πιο ισχυρά τα συστήματα προστασίας τροφίμων και αποτελεσματικά από ό,τι στο παρελθόν. Ποιε είναι λοιπόν οι αλλαγέ που γίνονται. Συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε το σχέδιο δράση που εκπονήθηκε μετά την Υπουργική Διάσκεψη. Οι υπηρεσίε Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι ομόλογοι στα κράτη-μέλη έχουν ε, συστήσει τρία δίκτυα για ε, διοικητική βοήθεια και συνεργασία, ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τρόφιμα και ζωοτροφές και για την απάτη στα τρόφιμα. Σε ένα ενιαίο σύστημα ε, ηλεκτρονικών υπολογιστών, σε μια εφαρμογή που ολοκληρώνεται όπως έχει σχεδιαστεί στα τέλη του 2018. Επίσης αναθεωρήθηκε η νομοθεσία για να υποστηρίξει αυτές τις αλλαγές με ένα νέο σύνδεσμο στον νέο κανονισμό για τους επίσης επίσημους ελέγχους. Εμείς συζητούμε ένα ε, σχέδιο κειμένου από τον Απρίλιο με τα κράτη-μέλη. Κανένα σύστημα δεν είναι ε, άψογο. Προβλήματα θα υπάρχουν και χρειάζονται πάντα βελτιώσεις, αλλά οι συγκεκριμένες πρόνοιες συνιστούν σημαντική βελτίωση. Προ, πριν προχωρήσω θέλω να πω δύο λόγια για τον πρωταγωνιστικό ρόλο που διαδραματίζουν τα κράτη-μέλη στην ακαιρεότητα του συστήματος ασφάλειας των τροφίμων. Ας πούμε πώς χρησιμοποιούν το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και τα υπόλοιπα. Ε, αυτό είναι βασική ε, ευθύνη των κρατών μελών. Η άλλη πλευρά του νομίσματος είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ε, εξασφαλίζει την ταχεία ε, και απρόσκοπτη ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Βεβαίως χρειάζεται Επίσης, ένας πρωταγωνιστικός ρόλος των κρατών ε, μελών για την πολυπόμενη παρακολούθηση, για την ταχεία και αποτελεσματική συνέχεια που δίνουμε για να ανταποκρινόμαστε σε κινδύνους. Χρειάζεται συλλογική λοιπόν, προσπάθεια αξιότιμοι βουλευτέ. Οι δικέ μα προδιαγραφέ για τα τρόφιμα και την ασφάλειά του ε, αφορούν και του διεθνεί εταίρου που θέλουν να εξάγουν προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται και σε αυτού. Θέλω να σα διαβεβαιώσω και πάλι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει ό,τι μπορεί για να προστατεύει την υγεία των Ευρωπαίων πολιτών. Και αυτό κυρίω ε, αφορά και το κρέα από τη Βραζιλία. Όταν ξέσπασαν τα σκάνδαλα ε, με τα κρέατα στην Βραζιλία, ε, αμέσως ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Βραζιλία να επιβάλλει αυστηρά μέτρα έτσι ώστε να είναι ασφαλείς εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα ενισχύθηκαν και οι εισαγωγικοί έλεγχοι ε, στα σύνορά μας. Η αρμόδια Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΤΕ έχει κάνει ήδη δύο ελέγχους στη Βραζιλία από πέρσι και αυτό τον καιρό τελειώνει έναν έλεγχο για ε, κατάλοιπα ε, κτηνιατρικών προϊόντων σε προϊόντα ζωικής προέλευσης από τη Βραζιλία. Στις 8 Μαΐου απαγορεύσαμε 20 εταιρείε να, ε, από να εξάγουν προϊόντα κρέατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές που ενέχονται στην απάτη. Επανειλημμένα τόνισα στο Βραζιλιάνο ε, αρμόδιο υπουργό ε, ότι είναι υποχρεωμένοι να ελέγχουν τι εξάγουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και φυλασσόμεθα να λάβουμε και περαιτέρω μέτρα αν χρειαστεί. Αντίστοιχα, έχουμε και μια εξυγχρονισμένη συνολική συμφωνία με το Μεξικό, όπου προτείνεται ένα ευρύτατο κεφάλαιο που αφορά υγειονομικά και φυτο θέματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ελέγξει σε βάθος τη δυνατότητα και την ικανότητα των μεξικανικών συστημάτων να εξασφαλίζουν ε, ότι εξάγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο βόλιο κρέα το οποίο ανταποκρίνεται στι προδιαγραφέ μα. Αυτό σημαίνει ε, να εγγυηθούν ότι ποτέ δεν έχουν χρησιμοποιηθεί αυξητικές ορμόνες και άλλοι αυξητικοί παράγοντες κατά την εκτροφή. Και αυτό θα γίνει πριν ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση για να επιτραπεί αυτό το εμπόριο. Και μια που συζητούμε τα θέματα του εμπορίου, θα ήθελα να τονίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει ό,τι μπορεί έτσι ώστε να εξασφαλίσει καλύτερη πρόσβαση στην αγορά ε, ε, των ευρωπαϊκών τροφίμων στην Κίνα. Ε, υπάρχει η αρχή της περιφεροποίησης που είναι πάρα πολύ μεγάλη προτεραιότητα για μένα και συνεργάζομαι με τους επιτρόπους Χόγκαν και Ελμάνστρομ για να πείσω την Κίνα να ε, προσχωρήσουν στις διεθνείς προδιαγραφές ε, στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων. Συναντήθηκα με τον αρμόδιο υπουργό 27 Μαΐου, τον Κινέζο, για να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Πρόσφατα ο επίτροπο Χόγκαν πήγε στην Κίνα και ζήτησε ε, πρόσβαση στην αγορά για βόλιο κρέα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ο αντιπρόεδρος Κατάινεν θα μεταβεί την άλλη εβδομάδα σε ένα υψηλού επίπεδου οικονομικό διάλογο με την Κίνα. Προτίθεμαι και εγώ να μεταβώ εκεί για να πείσω του αρμόδιου υπουργού για το πόσο στιβαρό είναι το σύστημά μα και πόσο ασφαλεί τα προϊόντα μα. Όταν ανέλαβα το άξιμα μου ε, υπήρχαν τότε 12 δράσεις που εκκρεμούσαν από τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ευημερία των ζώων. Και χαίρομαι που βρίσκομαι στην ευτυχή θέση να σας ενημερώσω ότι κάθε μία από αυτές ε, ολοκληρώθηκε. Τρεις από αυτές τις δράσεις ήταν καθοριστική σημασίας για να βελτιωθεί η εφαρμογή της κοινοτική της ενωσιακής νομοθεσίας. Μία σύσταση για την ευημερία των χείρων εγκρίθηκε το 2016, κατευθυντήριες γραμμές για τη μεταφορά των ζώων Λοιπόν δημοσιεύτηκαν το 2017 μία μελέτη για τις βέλτιστες πρακτικές για την προστασία των ζώων τη στιγμή τη σφαγή, ολοκληρώθηκε το 2017. Επιπλέον η Επιτροπή ενέκρινε έξι εκθέσει. Μία εξ αυτών αφορά στις επιπτώσεις ε, ε, στην ευημερία των ζώων μετά από δράσεις τη ευρωπαϊκή Ένωση. Φαίνεται λοιπόν ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο για μα η ευημερία των ζώων και η έκθεση επισημαίνει ότι υπάρχει προστιθέμενη αξία από τα ε, προϊόντα που τοποθετούνται στην αγορά μετά από την εφαρμογή υψηλών προδιαγραφών ευημερία των ζώων. Υπάρχουν και άλλε πέντε εκθέσει που αφορούν παρεμφερή τεχνικά θέματα. Πρέπει εδώ να αναφέρω ότι συστήσαμε το 2017 την ε, πλατφόρμα ευημερία των ζώων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Μάρτιο αυτού του έτους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όρισε, καθόρισε το πρώτο κέντρο ε, Ευρωπαϊκή Ένωση για την ευημερία των ζώων. Και τώρα θα αναφερθώ σε κάτι που είναι καθοριστική σημασία για όλους μας. Όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα νέο πρόγραμμα ευρωπαϊκό ε, δράσης για τη μικροβιακή αντοχή. Ε, έχουν γίνει πάρα πολλές συγκεκριμένες προτάσεις και η ε, τελευταία έκθεση θα δημοσιευτεί, θα επικαιροποιείται. Προσβλέπω λοιπόν στην ε, γνωμοδότηση, στην έκθεση πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το πρόγραμμα δράση. Η αντιμετώπιση τη ε, αντιμικροβιακών ουσιών είναι καθοριστική σημασία. Γνωρίζω ότι υπάρχουν διαπραγματεύσει για την, για την αντιμικροβιακή εντοχή και η μικροβιακή εντοχή και για, τις, για τα ε, ζω, φαρμακούχες ε, ζωοτροφές, ε, οι, κανονισμοί είναι καθοριστική σημασία, ολοκληρώθηκαν από τον μήνα και είναι καθοριστική σημασία. Θέλω να συγχαρώ του συζητητέ για το θέμα που παρουσίασαν σχετικά με τις φαρμακούχες ζωοτροφές. Υπάρχει ένα ολόκληρο σώμα δικαίου και παράλληλα πρέπει να επισημάνουμε ότι κανένα σύστημα δεν είναι επαρκές. Εμείς ε, θεωρούμε ότι θα πρέπει να αναζητάμε μια νέα διαδικασία για βελτίωση. Τον Απρίλιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τις προτάσεις για τη διαφάνεια και την βιωσιμότητα της ε, αξιολόγησης κινδύνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στην αλυσίδα διατροφής. Έχοντας πάντα αυτό κατά νου, η πρόταση δεν σημαίνει ότι παραγωνίζεται το σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε άλλο προκύπτει μια στοχευμένη αναθεώρηση του γενικού κανόνα για τα τρόφιμα και κάποιες τομεακές νομοθετικές παρεμβάσεις. Παρουσίασα την πρόταση στα κράτη-μέλη στο πλαίσιο του Συμβουλίου Αγκριφής και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Απρίλιο. Θέλω να υπογραμμίσω ότι μέσα από μια σειρά διαβουλεύσεων υπήρξε ενημέρωση για την πρόταση της Επιτροπής και θέλω να επισημάνω και τις ε, ανοιχτές διαβουλεύσεις για το κοινό που μέσα από ένα ερωτηματολόγιο που έτρεξε για περίπου 8 εβδομάδες. Βασίζεται σε τέσσερα, τέσσερις πυλώνες ε, η πρόταση. Πρώτον, ότι οι πολίτες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στην ενημέρωση από την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας Τροφίμων. Δεύτερον, να υπάρχει η ποιότητα των ε, μελετών που είναι απαραίτητε. Σε τρίτον, να συμπεριλαμβάνονται και τα κράτη-μέλη στη δομή της ΕΨΑ, να υπάρχουν επιστημονικά πάνελ, χωρίς όμως να απαγορεύουν τα ανεξάρτητα πάνελ της ΕΦΣΑ. Και τέλος, ε, νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό ε, θα ενισχυθεί η επικοινωνία ανάμεσα στην ΕΦΣΑ, τα κράτη-μέλη, τους άμεσα εμπλεκόμενους και την κοινή γνώμη. Στόχος μας είναι να εγκριθεί αυτή η πρόταση μέχρι την άνοιξη του 2019 η υποστήριξη του Κοινοβουλίου και αυτή τη Επιτροπή είναι καθοριστική σημασία αν θέλουμε να επιτύχουμε το στόχο μα. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, σα ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σα και α ξεκινήσουμε τώρα με μία ελπίζω επικοδομητική ε, συζήτηση, ερωτήσει και απαντήσει για να μπορέσουμε να ανταλλάξουμε απόψει. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Όπως ε, συνήθως θα δώσω το λόγο για δύο λεπτά στους συντονιστές. Δύο λεπτά στον κάθε συντονιστή λοιπόν. Ο Άλμπερτ Ντες είναι ο πρώτος ομιλητής. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ και σας ε, κύριε Επίτροπε. Ανδρικάητης ε, που μας ενημερώσατε. Δυστυχώς δεν μπορούσα να έρθω νωρίτερα από την αρχή της ομιλίας σας, αλλά γνωρίζω ότι εσείς ως ε, Επίτροπος κάνετε πάρα πολύ καλή δουλειά και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Παρακολουθώ την εργασία σας ε, εκ του και αυτό που με χαροποιεί ιδιαίτερα είναι ότι εσείς προσπαθείτε πάντα να λαμβάνετε υπόψη σας ε, τα συμφέροντα της γεωργίας και το γνωρίζω αυτό από τότε που είσαστε Επίτροπος. Αναφερθήκατε σε μία σειρά από ε, θέματα που αφορούν στη μικροβιακή αντοχή. Εγώ είδα λίγο τα στατιστικά δεδομένα στη Γερμανία και νομίζω ότι μπορεί κάτι να γίνει αν ληφθούν τα σωστά μέτρα. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι το 2011 στη Γερμανία είχαμε κατανάλωση ε, αντιβιωτικών 1.600 τόνους στη Γερμανία κατέτος. Και ε, Πέντε χρόνια αργότερα μόνο 850 τόνους. Δηλαδή μειώθηκε η χρήση κατά 900 τόνους με την εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω ε, να ε, συγκεντρώσετε και περισσότερα στοιχεία όσον αφορά την ε, ιατρική που αφορά στους ανθρώπους. Οι γεωργοί καταγράφουν ακριβώς πότε δίδουν αντιβιωτικά στα ζώα, αλλά αυτό δεν συμβαίνει στην περίπτωση των ανθρώπων. Και θα ήθελα να καταγράφετε και εκεί ακριβώς σε ποιον χορηγούν τα αντιβιωτικά, ποιος τα λαμβάνει, έτσι ώστε οι κατηγορίες να μην αφορούν μόνο τους γεωργούς. Γιατί έχουμε την εντύπωση ότι εμείς περιορίζουμε τα αντιβιωτικά αλλά στις ε, θεραπευτικές αγωγές ανθρώπων, εκεί διευρύνονται. Όσον αφορά στο εμπόριο, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, δηλαδή τον Οκτώβριο του 2010 στο Στρασβούργο, στην Ολομέλεια, αποφασίσαμε ότι οι εισαγωγέ γεωργικών προϊόντων θα επιτρέπονται μόνο εφόσον καλύπτονται οι δικέ μα προδιαγραφέ για την προστασία του καταναλωτή και την προστασία των ζώων. Να ισχύουν ελάχιστε προδιαγραφέ. Και αυτή η πρόταση εγκρίθηκε με ονομαστική ψηφοφορία ε, και πλειοψηφία 2 τρίτων. Νομίζω αυτό μπορείτε κάθε φορά να το επικαλείστε οποτεδήποτε συνάπτονται εμπορικέ συμφωνίε. Κατά την εισαγωγή προϊόντων, να εισάγουν υπάρχονται προϊόντα όπου δεν λαμβάνονται υπόψη οι δικέ μα προδιαγραφέ, αυτό σημαίνει απλά στρέβλωση του ανταγωνισμού. Τελειώνω να σα πω ότι πραγματικά εμπιστεύομαι την εργασία σα. Κύριε Αντριέ, ευχαριστώ. Και ζητώ και εγώ συγγνώμη από τον Επίτροπο γιατί δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω την παρουσίαση, αλλά συνεργαζόμαστε στενά, οπότε παρακολουθώ τους ή ε, το περιεχόμενο των εργασιών, αλλά και γνωρίζω τις προκλήσεις. Σας ευχαριστώ που φαίνεται να λαμβάνετε υπόψη προκλήσεις. Ε, εξού και οι βελτιώσεις που προτείνετε στις νομοθετικές διατάξεις για τα τρόφιμα, που είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Στην Επιτροπή Αλίας είχαμε μια σημαντική ανταλλαγή πληροφοριών ε, και συζήτηση και εδώ συζητούμε τα θέματα της φυτοπροστασίας ε, και τη χρήση φυτοφαρμάκων και υπάρχει κάποια βελτίωση κατάσταση. Πάντως η, η, αναθεώρηση της Γενικής Ομοθεσίας ε, για τα τρόφιμα έχει ουσιαδή σημασία γιατί η κοινωνία έχει φέρει και πάλι τη γεωργία στο επίκεντρο τη συζήτηση. Υπάρχει μια μεγάλη συνειδητοποίηση. Αντιλαμβανόμαστε ότι η γεωργία δεν είναι πια μια συνηθισμένη οικονομική δραστηριότητα, γιατί έχει άμεση σχέση με, την, με τα τρόφιμα, Γεωργία, και με την ανθρώπινη υγεία. Ε, ε, έχει, έχουμε συνειδητοποιήσει πια αυτή την αλληλεπίδραση, κάτι που μας υποχρεώνει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και αυστηροί στις εργασίες μας, γιατί είναι ε, μην αντιστρέψει αυτή τη διαδικασία τη επιρροή που έχει η γεωργία και στην υγεία των ανθρώπων μέσα των τροφίμων αλλά και στο περιβάλλον. Οπότε είμαστε μάρτυρες ε, και συμμέτοχοι μια ρηξικέλευτη αλλαγή. Θα πρέπει λοιπόν να παρακολουθήσουμε όλε αυτέ τι αλλαγέ, ε, συνοδεύοντα τις με τα απαραίτητα νομοθετικά μέτρα. Θα ήθελα τώρα να σα θέσω κάποιες ερωτήσεις για να διευκρινίσουμε συγκεκριμένα θέματα. Το ζήτημα της διαφάνειας είναι πολύ σημαντικό. Σε ποιο βαθμό οι προτάσεις σας ε, θα βελτιώσουν τη διαφάνεια των επιστημονικών μελετών που απαιτούν τη βάση για την αξιολόγηση των κινδύνων. Δεύτερη συναφής ερώτηση. Πρόσβαση του κοινού σε όλα τα δεδομένα. Είναι σημαντικό το θέμα της δημόσιας πρόσβασης. Είπατε ότι θα το σκεφτείτε. Ε, υπάρχουν ακόμη κάποιες εμπιστευτικές πληροφορίες και ποιες είναι αυτές τι απόρριτε πληροφορίες υπάρχουν, τι ελέγχου θα μπορούσε να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εξετάσει τη συμμόρφωση των εργαστηρίων και των μελετών με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Αυτό είναι μείζον ζήτημα. Ε, δεν μπορώ να αναφέρω διεξοδικά όλα τα σημεία. Κάνω μία σύνοψη. Πώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να βελτιώσει τη διακυβέρνηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλεια Τροφίμων, της, του ΕΦΣΑ. Χρειάζεται περισσότερα μέτρα ε, και μέσα για καλύτερη διακυβέρνηση. Πώς θα το εξασφαλίσετε. Σε ό,τι αφορά την ανακοίνωση επίσης, τελευταίο θέμα. Κύριε Επίτροπε, πώς πρόκειται να βελτιώσετε την επικοινωνία με το κοινό για την καλύτερη αξιολόγηση των κινδύνων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ. Η κυρία Μάκιντάιρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και τον Επίτροπο για την παρουσίαση που μας έκανε. Μας μιλήσατε για την σημασία που έχει ε, η παροχή ασφαλών τροφίμων στους Ευρωπαίους πολίτες. Και μας είπατε πως θα μεριμνήσετε ώστε να μην ε, χρησιμοποιούνται αυξητικές ορμόνες ή άλλοι αυξητικοί παράγοντες στο εισαγόμενα κρέατα. Επίσης, μιλήστε για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την ε, καλή μεταχείριση των ζώων για την ευζοία. Εσείς πώς εφαρμόζετε τις προδιαγραφές της καλής μεταχείρισης των ζώων στο κρέας και κυρίως ε, το εισαγόμενο κρέας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί φυσικά μας είναι προσφυλές το θέμα των ε, προδιαγραφών της καλής μεταχείρισης των ζώων και τα, τη στηρούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα πρέπει και το εισαγόμενο κρέας να πληρεί τις ίδιες υψηλές προδιαγραφές. Δεύτερη ερώτηση που τη προκάλεσε τα σχόλια του κυρίου Ντες, που πολύ εύστοχα μίλησε για τη σημασία που έχει η μικροβιακή αντοχή και η ανάγκη να αντιμετωπιστεί. Διερωτώ με, κύριε Επίτροπε, μιλήσατε με την ο, ειδική ομάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την ΝΑΤΖ, που ασχολείται με τη συμπεριφορά των καταναλωτών ε, δηλαδή με την ανάγκη να πείσουμε του καταναλώτε να κάνουν το σωστό χωρί να του αναγκάζουμε νομοθετικά να το κάνει. Γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αντίστοιχη εμπειρία. Σε ό,τι αφορά τη συνταγογράφηση αντιβιωτικών για του ανθρώπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω τη διαδικασία αυτού του NADS, αυτή τη ειδική ομάδα, μειώνεται ο αριθμό τη συνταγογράφηση αντιβιωτικών κατά 2 εκατομμύρια μέσα σε ένα χρόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, Μήπως θα μπορούσατε να μιμηθείτε το παράδειγμα του Ηνωμένου Βασιλείου και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μειωθεί έτσι έμεσα και όχι νομοθετικά η χρήση των αντιβιωτικών. Η κυρία Μίλλερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, Εχθές είχαμε την ευκαιρία στην Επιτροπή ΠΕΣΤ να το συζητήσουμε μαζί σας αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Και πάλι μιλήσατε για το γενικό πλαίσιο της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και η πρόταση που καταθέσατε τώρα πραγματικά επιφέρει διαφάνεια και τελικά καλύτερη επικοινωνία. Και θα πρέπει να υπάρξει καλύτερη επικοινωνία. Αυτό το αναγνώρισαν όλοι. Τώρα για την Αφρικανική Πανόλη των Χείρων. Οι ε, αγρότες ε, ανησυχούν πάρα πολύ. Ελπίζω όλα να πάνε κατευκήν, έτσι όπως τα σχεδιάζουμε. Δεν είμαι καθόλου εύκολη. Ε, τα προληπτικά μέτρα δεν ξέρω αν τηρούνται. Το θέμα της ευζοίας των ζώων μας απασχολεί εδώ και καιρό και την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο στη διακομματική ομάδα, το Intergroup, το σχετικό, ήρθαμε αντιμέτωποι με δύσκολα στοιχεία ε, και για τη μεταφορά ζών των μόσχων. Σας έκανα μια ερώτηση. Δεν θα πρέπει να επιτρέπονται εκτός της Ευρώπης μεταφορές ε, ζών, ζών των ζών προς φαγή μην στέλνουμε ζωντανά τα ζώα, το κρέας να εξάγουμε, γιατί δεν ξέρουμε τι γίνεται μετά τα σύνορα. Και ακούω από τη Νέα Ζηλανδία ότι έχουν ένα πάρα πολύ αυστηρό νόμο προστασίας των ζώων, όπου απαγορεύεται η σφαγή ε, χωρίς αναισθησία, μόνο με αναισθητοποίηση και μετά εξάγεται το κρέας. Αυτός είναι ο σωστός ε, δρόμος και ο σωστός τρόπος και θα πρέπει να είναι ο δικός μας στόχος. Ε, για την ε, αντίσταση των ε, μικροβίων στα αντιβιωτικά είναι καλό το σχέδιό σας, αλλά μια που είμαστε και στα παραγωγικά ζώα, να κάνουμε μια διάκριση ανάμεσα στα αντιβιωτικά για τα παραγωγικά ζώα και τα αντιβιωτικά για τα κατοικίδια ζώα συντροφιάς. Γιατί ε, δεν ξέρουν οι κτηνίατροι οι οποίοι κουράρουν ζώα συντροφιά, ε, γάτε, σκύλου κτλ. Αν θα πρέπει και αυτοί να δίνουν στοιχεία και να τηρούν μητρό για το πώ χρησιμοποιούν τα αντιβιωτικά. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Σας άκουσα σε αρκετές περιπτώσεις να ομιλείτε και προσπαθήσατε να μας καθησυχάσετε σχετικά με το κρέας, με αυτά που έρχονται από τη Βραζιλία, κυρίως όσον αφορά στα επιπρόσθετα προϊόντα που έρχονται από τη Βραζιλία. Δεν νομίζω ότι πείσατε κανέναν εδώ. Αλλά λέτε βέβαια συνέχεια τα ίδια και τα ίδια. Έχουμε ακούσει 100% ε, έλεγχη στα ζώα, μικροβιολογική έλεγχη. Υπάρχει μία έκθεση και φαντάζομαι θα την έχετε διαβάσει όπου στη Βραζιλία κατέστη σαφές ε, ότι δεν εφαρμόζεται τα ίδια στάνταρτ όπως ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, στα σφαγεία δεν τηρείται αρχείο για τα ζώα που σφαγιάζονται μεμονωμένα μόνο σε αυτά που σφαγιάζονται ομαδικά. Ως εκ τούτου δεν μπορούμε να ιχνηλατήσουμε πίσω το κρέας, να φτάσουμε στην ε, κτηνοτροφική μονάδα όπου εξετράφει το ζώο. Και ερωτώ, αυτή η ιχνηλασία τι νόημα έχει να υπάρχει εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την αρχή, τη στιγμή ε, που ε, δεν εφαρμόζεται και εδώ ζητάτε και τελευταία λεπτομέρεια ακόμα και τον, ε, το χρώμα του εσώρουχου ενό Γεωργού αλλά έχουμε περιπτώσεις όπου δεν ισχύουν όλα αυτά βέβαια και θα τα έχετε ακούσει έχουν ληφθεί επανειλημμένα φοβάμαι όμως ότι ισχύουν επίσης όλα αυτά είναι φάρσα. Τι νόημα έχει να εφαρμόζονται εδώ συγκεκριμένε προδιαγραφέ όταν εισάγεται κρέα από άλλε περιοχέ που δεν πλησιάζουν καν στι δικέ μα. Και όσον αφορά την εφημερία των ζώων, τι θα κάνετε, θα παρακολουθείτε τα ζώα στη Βραζιλία για να δείτε πώ το συμπεριφέρονται, θα βάλετε chips στα ζώα, κάμερε, πώς θα γνωρίζετε ότι εκεί εφαρμόζονται οι ίδιες προδιαγραφές όπως εδώ. Η απάντηση είναι ότι δεν ε, θα γνωρίζετε αν εφαρμόζονται αυτές οι προδιαγραφές. Εμείς συνεχίζουμε να τα λέμε, αλλά φοβάμαι ότι δεν μας ακούτε πια. Και εγώ θα ξεκινήσω με τη Βραζιλία γιατί πήγαμε ως Επιτροπή Επιτόπου και πρέπει να σας πω κραν πόρο απέχουμε από το να εφαρμόζονται οι δικέ μα οι προδιαγραφέ στη Βραζιλία. Παρ' όλα αυτά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει να διαπραγματεύεται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, αγνοεί και συνεχίζει να διπραγματεύεται και με τη Μερκοσούρ, σαν να μην υπάρχει κανένα απολύτω αποτέλεσμα. Αυτό πρέπει όμω να μου το εξηγήσετε. Για το Μεξικό μιλάμε για προδιαγραφέ που δεν μπορούν να ε, τηρηθούν με τι δικέ μα. Και ανεξάρτητα από αυτό, στη συγκεκριμένη περίπτωση τη Βραζιλία, ε, πρέπει να πούμε ότι είχαμε μία μακρά σε βάθο συζήτηση για τη γλυφοσάτη, αλλά οι ποσότητε χρήση τη γλυφοσάτη στη Βραζιλία είναι 10 φορέ πιο μεγάλε και ακριβώ Δυστυχώς αυτή η σόγια εισάγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να τα πω ξεκάθαρα πρέπει να εφαρμόζουμε παντού τα ίδια μέτρα και δύο σταθμά. Πάω στα ε, φυτοφάρμακα. Ένα πράγμα που με εκπλήσει είναι το εξής. Ε, ε, απαγορεύτηκαν τα νοικοτινοειδή, ε, αυτό το δέχτηκαν όλοι και τώρα ακούμε ότι ορισμένες χώρες λένε ότι ενδεχομένως ε, να υπάρχουν κάποιες έκτακτες καταστάσεις για τα νοικοτινοειδή στη Ρουμανία, ακόμα ίσως και στο Βέλγιο μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Τι γίνεται, πώς ταιριάζει αυτό. Είτε θα πούμε ότι απαγορεύουμε από την αγορά, είτε θα πούμε ότι μπορούμε να έχουμε κατεξαίρεση περιπτώσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν ε, ισχυρίζει ότι όλα αυτά είναι επικίνδυνα, πρέπει να φροντίσει ώστε να εξαφανιστούν από την αγορά. Και κάτι άλλο. Ε, πώ μπορούμε να ε, είμαστε σίγουροι ότι αυτή η πρωτοβουλία για τη διαφάνεια τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που είναι ένα βήμα προ τα εμπρό, πώ μπορεί να εφαρμόζεται και στι λεπτομέρειε. Γιατί οι εταιρείε θα μπορούν να πούν ότι πρόκειται για επαγγελματικά, επιχειρηματικά, μυστικά και έτσι ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλεια Τροφίμων δεν ξέρω αν θα μπορεί να ελέγξει κατά πόσο εφόσον τα έγγραφα που θα έχουν κατατεθεί είναι ε, σωστά ή όχι. Για να το κάνει αυτό χρειάζεται περισσότερα χρήματα και μεγαλύτερο και περισσότερο προσωπικό. Κάτι άλλο, ο κανισμός ε, για τα φάρμακα εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία. Νομίζω όμως, όπως είπε και ο κύριος Ντές, δεν θα πρέπει να μιλάμε μόνο για τους τόνους ε, που χρησιμοποιούνται, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η χρήση. Να το κοιτάμε και αυτό. Και συμφωνώ απόλυτα και στην περίπτωση του ανθρώπου θα πρέπει να περιστεί η χρήση των αντιβιωτικών. Νομίζω ότι από αυτού του σημείου ε, συμφωνούμε όλοι. Ο κύριος Άγνιο, ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, εγώ ασχολούμαι με την πτυνοτροφία και αυτή την κατεύθυνση έχουν και οι ερωτήσει μου. Καταρχήν για τη μικροβιακή αντοχή, την οποία ανέφεραν και οι Κατά τη γνώμη μου αυτό είναι το μείζον πρόβλημα που έχουμε στη Γεωργία αυτή τη στιγμή είναι να προσπαθήσουμε να σταματήσουμε την υπερβολική χρήση φαρμάκων αντιβιωτικών, ώστε να μην λαμβάνουν τα αθεκτικά βακτηρίδια, να μην περνάνε στου ανθρώπου. Γιατί να μην έχουμε λοιπόν ε, καμία ε, ταψηλή επιχορήγηση για την βιοασφάλεια, γιατί όλοι γι' αυτό μιλάνε, βιοασφάλεια. Μόνο έτσι θα μειώσουμε τον αριθμό των ασθενειών, αλλά χρειαζόμαστε ε, υποδομή που είναι δαπανηρή. Γι' αυτό χρειάζεται μια πλουσιοπάροχη επιδότηση. Επίσης έχουμε άγρια πτηνά που είναι, έχουν ανθεκτικότητα σε κάποια προβλήματα. Εμεί έχουμε τη γενετική ικανότητα αυτά τα βασικά ανθεκτικά γονίδια να μεταφέρουμε στα κατοικίδια μα και στα, ε, στα πτηνά. Ε, και αν οι, οι κτηνοτρόφοι αποφασίσουν να καταργήσουν τα αντιβιωτικά, να ξέρουν ότι αν αντιμετωπίσουν πρόβλημα θα έχουν ένα δίκτυο ασφαλείας για να μπορέσουν να αντικαταστήσουν τα χαμένα πτηνά. Επίσης, η γρήπη των πουλερικών. είπαμε ότι κάποια στελέχη της γρήπης μπορούν να, να μεταδοθούν και στον άνθρωπο και εκεί μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Επίσης, κάποια άγρια πτηνά που προσβάλλονται από την γρήπη των πουλερικών τελικά αναρώνουν, άρα έχουν ανθεκτικά γονίδια. Αυτά δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και να τα μεταφέρουμε και στα εξημερωμένα πτηνά. Ε, επίσης, ε, τα πουλιά, τα πτηνά ελευθέρας βοσκήσεως είναι πιο επιρρεπή στην ε, γρήπη των πουλερικών, μια κυκλοφορούν ελεύθερα. Οπότε θα πρέπει να προβλέψουμε κάποιες ε, αντισταθμίσεις για να περιορίσουμε ίσω την επαφή με τα άγρια πτηνά. Και από πού θα έρθουν όλα αυτά τα κονδύλια. 40% του προπολογισμού του γεωργικού προπολογισμού αφορά κλιματικέ δράσει. Κατά τη γνώμη μου, είναι σπατάλη χρημάτων. Νομίζω ότι ένα μεγάλο τμήμα, μεγάλο μερίδιο αυτού του γερικού προπολογισμού θα πρέπει να πηγαίνει σε δράσει αυτέ που σα παρουσίασα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Όπως είχαμε συμφωνήσει, μετά τον πρώτο γύρο των συντονιστών, θα δώσω το λόγο στον Επίτροπο για να σχολιάσει τι παρατηρήσει και να απαντήσει σε ερωτήσεις και θα ακολουθήσει δεύτερο γύρος ερωτήσεων με του υπόλοιπου ευρωβουλευτές. Ευχαριστώ. Είπατε για την ΚΑΠ και το 40% του γεωργικού προπολογισμού και πού πηγαίνει. Μα εναπόκειται στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμφωνήσουν για τα ποσοστά και τις αναλογίες, ε, ανάλογα με τις ανάγκες και την πραγματικότητα. Δεν είναι βέβαια τόσο εύκολο κάτι τέτοιο. Και οι απλοποίηση μερικέ φορές δημιουργούν πολλά προβλήματα. Α είμαστε σαφεί και συνεπεί. Και να ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση του κύριου Ντες. Αναφερθήκατε σε ένα πολύ καλό παράδειγμα και μας παρουσιάσετε ένα γερμανικό παράδειγμα με τη μειωμένη χρήση αντιβιωτικών. Τώρα πολλά κράτη-μέλη κάνουν κάτι παρόμοιο. Και αυτό αποτελεί καλό παράδειγμα ότι τα μέτρα μας και οι διατάξεις μας ε, στο σχέδιο δράσης για την ενιαία υγεία, One Health, αποτέλεσαν ισχυρό εργαλείο για τη μείωση της χρήσης των αντιβιωτικών. Τώρα έχουμε και νέους μηχανισμούς και νέα εργαλεία στα χέρια μας. Έχουμε πια πολλές δυνατότητες ε, να περιορίσουμε τη χρήση φαρμάκων. Έχουμε τους δύο κανονισμούς για τα κτηνιατρικά φάρμακα και τις φαρμακούχες ζωτροφές ε, που διεκπαιρεώθηκαν αυτές τις μέρες, αλλά αναφερθήκατε και στην ανθρώπινη υγεία. Όταν υιοθετήσαμε το σχέδιο δράση για τη μικροβιακή εντοχή, το συνοδεύσαμε με κάποιε κατευθυντήριε γραμμέ για τη σωστή χρήση αντιβιωτικών για τον άνθρωπο. Αυτό έγινε πέρυσι. Επίσης, έχουμε πολλά εργαλεία για ταχύτατους διαγνωστικούς ελέγχους. Γιατί θα πρέπει να εξοπλίσουμε, να εφοδιάσουμε τους παθολόγους μας ε, μέσω στα διαγνωστικά εργαλεία για να μπορούν αμέσω να αποφασίζουν αν πρόκειται για ιό ή βακτηρίδιο. Και υπάρχουν πολλά κονδύλια που αφιερώνονται σε αυτό το σκοπό. Είχαμε μάλιστα θεσπίσει και ένα βραβείο ε, για όσους προτείνουν ε, νέα διαγνωστικά εργαλεία ώστε να βοηθήσουμε τους παθολόγους μας, τους γενικούς μας παθολόγους, να κάνουν πιο γρήγορα τη διάγνωση, γιατί αν πρόκειται για ιό ή για μικρόβιο. Επίσης, ε, γιατί, για τον εμβολιασμό. Είδατε τις συστάσεις του Συμβουλίου με το νέο πλαίσιο δυνατοτήτων για τη βελτίωση το, της δυνατότητας εμβολιασμού. Προκειμένου να καλυφθεί το θέμα της εποχιακής γρήπης. Αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα. Τα εμβόλια μερικές φορές μας βοηθούν να περιορίσουμε τον αριθμό των νοσούντων. Γιατί πολλές φορές ε, κάποιοι που κολλάνε γρήπη ή έχουν κάποια λίμωξη ή με κάποια φλεγμονή μετά χρησιμοποιούν αντιβιωτικά και έτσι εντείνεται η μικροβιακή αντοχή. Θα πρέπει λοιπόν με, τον εμβολιασμό να αποτρέψουμε το να νοσήσει κανεί. Και χρειαζόμαστε κάποιου αυστηρού δείκτε νοσοκομιακού ελέγχου και ελέγχου στη χρήση των αντιβιωτικών. Να χρησιμοποιούνται αντιβιωτικά μόνο μετά από συνταγογράφηση. Έχουμε πολλού μηχανισμού πια, πολλά εργαλεία, ώστε να αποφύγουμε την κατάχρηση των αντιβιωτικών στον άνθρωπο. Και θα συνεχίσουμε ε, προς την κατεύθυνση αυτή για να περιορίσουμε την χρήση των αντιβιωτικών. Επίσης, ε, ζητήσαμε από τα κράτη-μέλη να οριστικοποιήσουν τα εθνικά σχέδια δράσης τους μέχρι τα τέλη του έτους για να εξασφαλίσουμε μία ε, συνοχή και συνέπεια μεταξύ του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης και των Εθνικών Σχεδίων Δράσης. Και έτσι να αναπτύξουμε κάποιες κοινέ προσπάθειες ε, και πολύ συνεκτικές στον τομέα αυτό. Αναφερθήκατε και στη Γενική Νομοθεσία για τα τρόφιμα. Τη διαφάνεια και τις μελέτες, τις επιστημονικές μελέτες που χρησιμοποιούνται Ε, για την αξιολόγηση του κινδύνου και πώς θα εξασφαλίσουμε δημόσια πρόσβαση αυτών των επιστημονικών μελετών. Και επίσης ε, το θέμα της διακυβέρνησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Τροφίμων είναι πολύ σημαντικό και τις ανάγκες ενίσχυσης της επιστημονικής ικανότητας ε, του ΕΦΣΑ και την ανάγκη να ελέγχουμε και τα εργαστήρια που κάνουν τις δοκιμές. Επίσης, μας καταδείξατε την αλληλεπίδραση μεταξύ ε, της γεωργίας, ε, της παραγωγής τροφίμων, της ε, υγείας των ανθρώπων και στη κοινή γεωργική πολιτική και στην μεταρρύθμιση της ζητούμενο είναι ασφαλή τρόφιμα και ζητούμε από τα κράτη-μέλη να έχουν διατροφικές πολιτικές ιδιαίτερα για τα παιδιά και τους εφήβους. Θέλουμε σωστές πολιτικές διατροφής, περιεκτικές, ολιστικές και κατάλληλα σχέδια διατροφής σε εθνικό επίπεδο, ώστε να καταναλώνουμε ασφαλή τρόφιμα και μάλιστα σε κοινωνικά προσιτές τιμές. Αυτό είναι μείζον ζήτημα και σίγουρα θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Τώρα εναπόκειται στα κράτη-μέλη να κινηθούν προς, την, προς αυτή την κατεύθυνση με τέτοιες σωστές πολιτικές διατροφής. Σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε όλες οι μελέτες και οι συναφείς πληροφορίες που υποβάλλονται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας Τροφίμων για ε, ε, αξιολόγηση κινδύνου να είναι δημόσια προσιτές ε, και μάλιστα αυτόματα και από, την πρώιμη φάση της διαδικασίας. Βέβαια, την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών θα την εξασφαλίσουμε υπό όρους όμως και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, σε περιορισμένες περιπτώσεις. Τώρα έχουμε ένα νομικό πλαίσιο, την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και κάποιες επιπλέον προϋποθέσεις σε τομεακές νομοθεσίες. Αλλά αυτή τη στιγμή ο ΕΦΣΑ έχει και έναν θετικό κατάλογο κριτήριων και έτσι είναι πολύ πιο εύκολο τώρα να εφαρμόζει πολύ πιο σαφή κριτήρια για το απόρριτο, για τον απόρριτο χαρακτήρα των μελετών και ο ΕΦΣΑ μπορεί να αξιολογεί όλα τα έγγραφα και κατόπιν να επαληθεύει την κατάσταση. Και αν κάτι δεν ευθυγραμμίζεται με τα κριτήρια ε, και δεν χρειάζεται να πληρείται η εμπιστευτικότητα, γίνεται δημόσια προσιτή η σχετικά επιστημονική μελέτη, που μάλιστα θα είναι και προσιτή σε ηλεκτρονική μορφή και το θέμα της αποκλειστικότητας και προστασίας δεδομένων ή προστασίας πνευματικών δεδομένων θα πρέπει όλα αυτά να καθορίζονται πολύ σαφέστερα, ιδιαίτερα στις ε, ε, τομεακές νομοθεσίες και προτείνονται αναθεωρήσεις σε οκτώ τέτοιες τομεακές νομοθεσίες, ώστε να έχουμε μια πιο συνεπή και συνετή προσέγγιση. Και φυσικά κάτι τέτοιο καλύπτει όλη την τροφική αλυσίδα, όχι μόνο τα φυτοφάρμακα. Η διαφάνεια θα πρέπει να καλύπτει όλη την αλυσίδα, όλη την τροφική αλυσίδα και όλους τους ετούντες. Είτε παράγουν φυτοφάρμακα, είτε παράγουν πρόσθετα ε, που περιλαμβάνονται στα τρόφιμα, είτε κάτι άλλο. Είναι σημαντικό όλα αυτά να γίνονται με το σωστό και διαφανή τρόπο. Και επίσης ε, για την πρόσβαση στα δεδομένα. Ε, καταρχήν, ε, θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση σε μη επεξεργασμένα δεδομένα ε, με επιφύλαξη των εξαιρέσεων και ο πλήρης δημόσιος έλεγχος εξαρτάται και γίνεται μάλλον με τη βάση της παροχής των μη επεξεργασμένων δεδομένων, raw data. Σε ό,τι αφορά τη διακυβέρνηση, φυσικά προσπαθούμε να βελτιώσουμε τη διακυβέρνηση, μια και πια στο Διοικητικό Συμβούλιο θα έχουμε και εκπροσώπους των κρατών μελών, εκπροσώπους των μη κυβερνητικών οργανώσεων, του κλάδου, αλλά και εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, οι εκπρόσωποι αυτοί θα αφορούν περισσότερο θέμα της αξιολόγησης και όχι της διαχείρισης του κινδύνου. Και εδώ θα έχουμε κριτήρια. Και θα ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις για την ε, συμβατότητα ή σύγκρουση συμφερόντων. Θέλουμε να αποφύγουμε οπωσδήποτε σύγκρουση συμφερόντων η ασυμβατότητα. Και επίσης στο νέο πολίτες δημοσιονομικό πλαίσιο θα προβλέψουμε επιπλέον χρηματοδότηση 62,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο θα αφιερώνουμε στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας Τροφίμων. Τώρα εξαρτάται από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τους συνομοθέτες αν θα δεχτούν την πρόταση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πάντω ε, σίγουρα με το επιπλέον αυτό κονδύλιο θα βελτιώσουμε την οικονομική δυνατότητα της ΕΦΣΑ, ε, του ΕΦΣΑ μάλλον, και την δυνατότητα να προσλάβει επιπλέον προσωπικό. Και μπορεί έτσι να προσλάβει και επιπλέον επιστήμονες. Όχι μόνο από τα πάνελ στα οποία συμμετέχουν ε, εκπρόσωποι των κρατών μελών, αλλά και εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Η κυρία Μακεντάιρ ρώτησε πώς θα εφαρμόσουμε τις ε, δικές μας υψηλές προδιαγραφές ε, ευζοίας και στα εισαγόμενα προϊόντα. Στα εισαγόμενα προϊόντα από τρίτες χώρες. Καταρχήν, χάρη στις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο Παγκόσμιο Οργανισμού Υγείας των Ζώων. Τώρα έχουμε τέτοιες υψηλές προδιαγραφές ευζοίας παγκοσμίω. Φυσικά δεν είναι ίσως τόσο υψηλές όσο οι δικές μας οι κοινοτικές οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές, αλλά σίγουρα έχουν αναβαθμιστεί οι προδιαγραφές ε, στον Παγκόσμιο Οργανισμό ε, Υγείας των Ζώων. Και δεν είναι εύκολο να επιβάλλουμε το ίδιο υψηλό επίπεδο προδιαγραφών, αλλά σίγουρα συμβάλαμε στη βελτίωση και αναβάθμιση αυτών των προδιαγραφών παγκοσμίω. Επίσης, ε, προσφέρουμε αρρωγή στις χώρες Μέση Ανατολής ε, και καταρτίζουμε εμπειρογνώμονες ε, για τα, για τα πρότυπα και τις προδιαγραφές μας. Έχουμε ειδικά προγράμματα για τις χώρες αυτές. Κυρίως για τη μεταφορά ζώων που πηγαίνουν προς χώρες μέσης της Εγγύης και Μέσης Ανατολής. Έτσι συμβάλλουμε στην αναβάθμιση των προδιαγραφών αυτών και στις χώρες της ΕΕ. και Μέσης Ανατολή. Επίσης έχουμε διμερείς εμπορικές συμφωνίες με τρίτες χώρες. Στις εμπορικές αυτές συμφωνίες έχουμε ειδικά κεφάλαια για την ευζοία, για την καλή μεταχείριση των ζώων. Ο κύριος Χόισλινγκ αναφέρθηκε στη Συμφωνία Μερκοσούρ. Πολύ καλό παράδειγμα. Και στη συζήτηση η Μερκοσούρ συμφώνησε να συμπεριλάβει στη συζήτηση και θέματα μικροβιακής αντοχής και καλής μεταχείρισης των ζώων. Γιατί ε, η εμπορική συμφωνία δεν είναι μία μονοσήμαντη συμφωνία, είναι αμφίδρομη συμφωνία. Και δεν θα πρέπει φυσικά να απαγορεύσουμε ε, τις αγωγές από όλες τις τρίτες χώρε μέχρι ότου ανοίξουν την αγορά του ε, στα δικά μας προϊόντα. Φυσικά χρειάζεται απλούστευση. Και ίσως θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα προγράμματα κατάρτισης για να έχουμε πιο ασφαλή τρόφιμα. Και τέτοια προγράμματα έχουμε κάθε χρόνο. Και στέλνουμε τους ειδήμονές μας σε τρίτες χώρες για να συνεργαστούν με τους, τους ε, εθνικούς εμπειρογνώμονες των τρίτων χωρών για να αναπτύξουν και τα δικά τους πρότυπα και τις προδιαγραφές για την ευζοία. Επίσης, τα μηνύματά μας θα πρέπει να τα διαδώσουμε στην κοινωνία μας, στους γεωργούς και κτηνοτρόφους μας, για να δουν ότι πραγματικά κάνουμε πολλά στις διμερείς μας σχέσεις με τις τρίτες χώρες, τις εμπορικές μας συμφωνίες. Δεν είναι ότι Μπορεί Είναι εύκολο να με βλέπετε στον κακό της ιστορίας, αλλά δεν είμαι μόνο εγώ. Θα πρέπει να αναλάβουμε και εμείς τις ευθύνες ε, ε, τις ευθύνες μας και να βοηθήσουμε τους εταίρους μας τρίτες χώρες να αντιληφθούν την περιπλοκότητα του ζητήματος καλής μεταχείρισης των ζώων. Η κυρία Μακεντάιρ επίσης ε, αναφέρθηκε ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο και το πώς καταπολεμούν την αντίσταση των μικροβίων στα αντιβιωτικά. Ε, και πολλές άλλες χώρες σας μιμούνται. Είναι πραγματικά πολύ καλό. Τώρα έχουμε το δίκτυο Ενία υγεία One Health που απαρτίζεται από εκπροσώπους όλων των κρατών μελών και συζητούμε εκεί πολλά θέματα που έχουν να κάνουν με την υγεία και την διάδοση βελτίστων πρακτικών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και με ε, μεγάλη επιτυχία το δίκτυο. Η κυρία Μούλερ ρώτησε τι γίνεται με την αφρικανική πανόλη του χείρου και με την ευζοία των ζώων κατά τις μεταφορές ζών των ζώων. Μάλιστα. για την Αφρικανική Πανόλη του Χείρου. Ξέρετε ότι έχουμε επίμονη παρουσία της ε, νόσου αυτής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Ε, ε και ε, Εστονία, Πολωνία, Τσεχική Δημοκρατία, Ουγγαρία και Ρουμανία έχουν ανοιχνεύσει ε, τέτοια κρούσματα είτε στους ε, χείρους που εκτρέφονται σε χειροτροφία είτε σε αγριογούρουνα. Ε, έχουμε πραγματικά πολλά μέτρα, αν μου επιτρέπετε... Το μεγαλύτερο θέμα εκεί είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Δεν είναι μόνο ο αγριόχειρος. είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να, ε, και πολύ δύσκολο να έχουμε αποτελέσματα αν δεν υπάρχει ανθρώπινη αντίδραση. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Στέλνουμε ομάδες ελεκτών εκεί, βοηθούμε, ανανεώνουμε τη στρατηγική μας για την ευζοία των ζώων κάθε τρεις μήνες και ζητούμε από τον Οργανισμό Ασφάλειας Τροφίμων, ΕΦΣΑ, να δούμε πώς μπορούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ελέγξουμε το μηχανισμό των αγριοχείρων και με ποιες μεθόδους δεν αρκεί το κυνήγι, μπορεί να βρούμε και νέες μεθόδους. Και τώρα περιμένουμε από την ΕΦΣΑ να μας απαντήσει ή να μας συμβουλεύσει. Και βεβαίως έχουμε και μέτρα βιοασφάλειας και αυστηρά τα οποία εφαρμόζουμε μπορείτε αν θέλετε να σας στείλουμε όλα τα στοιχεία και τις λεπτομέρειες για τις δραστηριότητες αυτές, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό το νόσημα. Και συνεργαζόμαστε πάρα πολύ με τους γειτονές μας, Ουκρανία, ε, Μολδαβία, Λευκορωσία και Ρωσία, γιατί η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη. Αν δεν μπορείς να εναρμονίσεις τις στρατηγικές σου, είναι πάρα πολύ δύσκολο να σταματήσεις τη διάδοση ενός τέτοιου νοσήματος. Και πραγματικά έχουμε μεγάλες δράσεις. Το καλοκαίρι θα πάμε στη Λευκορωσία για να συζητήσουμε με τους αρμόδιους και υπηρεσιακούς παράγοντες και για την ε, μεταφορά ζών των ζώων. Γνωρίζετε Ναι, ναι, ξέρω. Ε, είπατε και για την αναισθητοποίηση στα σφαγεία. Κάποιοι μας ζητούν να σταματήσουμε να εξάγουμε ζώντα ζώα. Δυστυχώ is, Δυστυχώς αυτό είναι αδύνατο. Είναι αδύνατο αυτό. Δεν υπάρχει κανένας οικονομικός λόγος για να γίνει αυτό. Καλύτερο είναι να έχεις προδιαγραφές και πρότυπα και να τις στηρείς και να ζητούμε από όλους τους ενεχομένους να τηρούν τους ίδιους κανόνες και να έχουμε και πάρα πολύ αυστηρούς ελέγχους ε, για τις μεταφορές. Ξέρουμε ότι το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, διότι έχουμε εξαγωγές πολλές ζών των ζών και ζητούμε από όλα τα κράτη-μέλη να συνεργάζονται για να δούμε πώς μπορούμε να ε, προγραμματίζουμε ε, τις ε, δραστηριότητες τις εξαγωγικές με τους μεταφορείς για να μην προκαλούνται προβλήματα σε σημεία όπως είναι το καπιτάν Αντρέπ στην Βουλγαρία σε διαβάσεις συνοριακές. Και Χαίρομαι πολύ για την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την αναισθητοποίηση. Είναι πάρα πολύ σαφής ε, η κατάσταση και μπορούμε να ακολουθήσουμε για να δούμε πώς μπορούμε και πάλι να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να ε, εφαρμόσουν αυτή την απόφαση ε, του Δικαστηρίου για την σφαγή των ζώων όταν πρόκειται για κάποιες θρησκευτικέ μορφές και κανόνες σφαγής. Πώς να το πω τώρα, πώς να το διατυπώ. για θρησκευτικούς λόγους τα σφάζουν αλλιώς, χωρίς αναισθητοποίηση. Ε, είμαστε σε μόνιμο διάλογο με τα κράτη-μέλη για αυτό το θέμα. Βεβαίως, ε, έχουμε ελέγχους, έχουμε εκθέσεις, έχουμε μελέτες, έχουμε συμβουλές που παρέχονται. Και βεβαίως όλα αυτά τα θέματα αφορούν ε, την πλατφόρμα για την ευζωία των ζώων και εκεί συζητούνται. Ο κύριος Φλάναγκαν. Ε, μας ρωτήσατε για τη Βραζιλία. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Το σύστημα εισαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, έχει πάρα πολύ ε, αυστηρούς ελέγχους. Στις 8 Μαΐου ε, αποφασίσαμε να βάλουμε σε μαύρη λίστα 20 επιχειρήσεις από τη Βραζιλία. Αυτό είναι άλλη μία απόδειξη της ισχυρής βούλησης και δέσμευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προστατεύει τον Ευρωπαίο καταναλωτή. Θα διατηρήσουμε τους ελέγχους, θα τους αυξήσουμε μάλιστα, θα εξακολουθήσουμε να μπλοκάρουμε οποιαδήποτε νέα προσθήκη επιχείρηση ή περιφέρεια στις εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν γίνει έλεγχοι πρόσφατα και οι έλεγχοι μας ε, αποτελούν τη βάση για να πάρει ε, θεμητά όποια μέτρα και ε, όποια 11 μέσα έχει στη διάθεσή της να εκμεταλλευτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά έχουμε και ε, διεθνείς υποχρεώσεις ε, και με τεκμηρίωση έχουμε προβεί σε αυστηρά μέτρα κατά της Βραζιλίας. Βεβαίως είμαστε σε μόνιμη και διαρκή επαφή για να βελτιώνεται η δυνατότητα της Βραζιλίας να παρέχει περισσότερη διαφάνεια ε, για να υπάρχει επίσημο σύστημα ελέγχου στη Βραζιλία. για τα ε, ε, παρασιτοκτώνα, μάλλον τα ζυζανιοκτώνα, τα φυτοφάρμακα, το γλυφοσάτι, ότι χρησιμοποιεί περισσότερη η Βραζιλία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ γίνεται λόγος για εκτίμηση κινδύνου, για ε, δραστικές ουσίες, για να δούμε αν είναι καρκινογόνες ή όχι. Αλλά για τα φυτοφάρμακα, αυτό είναι στα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν μέτρα που δεν θα επιτρέπουν Ε, κατάχρηση ε, φυτοφαρμάκων. Ε, δεν θα το συζητήσουμε εμείς με το Μερκοσούρ για τις συμφωνίες μας, τις εμπορικές, με βάση τους κανόνες του εμπορίου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο βέβαια κάθε φορά να εισάγουμε τέτοια μέτρα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε πολλά προβλήματα με τα φυτοφάρμακα και τώρα προτείνουμε να απαγορευθούν τέσσερα φυτοφάρμακα, μάλλον όλα τα φυτοφράγματα που είναι τοξικά για τον άνθρωπο. Τα κράτη-μέλη δεν συμφωνούν αυτή τη στιγμή για το TICAT Ή... Χρησιμοποιούμε κάποια ε, λιπάσματα ή το χαλκό στη βιολογική γεωργία αντί για φυτοφάρμακα που και αυτό είναι προβληματικό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνει μεγάλη συνέπεια όταν κάνει λόγο για έλεγχο φυτοφαρμάκων κτλ. Κύριε Άγνιου, η προσέγγιση σας είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι πάρα πολύ καλό να δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιούμε καλύτερα τις σύγχρονες τεχνολογίες για τους ενδημικούς βυρούς. Ε, συγγνώμη. Ε, γιατί έχουμε αποδημητικά πτηνά ε, άγρια πτηνά που έρχονται από το Βόρειο Πόλο ξέρω εγώ και ε, μεταδίδουν την γρήπη των πτηνών και πρέπει να δούμε τι πρέπει να κάνουμε και τι μπορούμε να κάνουμε για τους ιούς αυτούς εκεί που ενδημούν. Εκεί χρειάζεται βέβαια νέα τεχνολογία, νέα έρευνα και νέα ε, μέσα και εργαλεία και ζητήσαμε από τους συναδέλφους της έρευνας και ανάπτυξης να επιληφθούν και να το κοιτάξουν. Ε, για να μπορέσουν οι επιστήμονες να μας βοηθήσουν ε, να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τέτοια φαινόμενα. Και τα εμβόλια κατά της νόσου αυτής, της γρήψης των πτηνών, δεν είναι εύκολο. Η απάντηση δεν είναι να περικοπούν τα κονδύλια στην ε, κοινή γεωργική ε, πολιτική. Έχει να κάνει και με την κλιματική αλλαγή. Δεν συμμερίζομαι τη δική σας άποψη, κύριε Άγνιο. Περνάμε τώρα στην, στο δεύτερο γύρο της συζήτησης. Η ε, κυρία Πετήρη είναι η πρώτη που ζήτησε το λόγο. Ή μάλλον πρώτα η μαλλον πρωτα Αγγιλέρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Επίτροπε. Πάρα πολύ εκτενείς ήσασταν σε πολλά θέματα. Κανένα δεν αποφύγατε. Θέλω να σας πω το εξής. Ε, ξέρω, θα υπάρξει τριμερής διάλογος, ε, θα έχουμε πολύ καλή ε, νομοθεσία για τις φαρμακούχες ε, ζωοτροφές, για την αντίσταση στα αντιβιωτικά. Ε, είμαστε ικανοποιημένοι και ελπίζω και στους δύο τριμερείς διαλόγους να ευοδοθεί αυτή η προσπάθεια και να εγκριθεί η πρόταση. Επειδή δεν έχουμε χρόνο, θέλω να αφαιρθώ σε αυτό. Έχουμε ένα σύστημα ελέγχου των εισαγωγών και είναι σημαντικό να είναι άκαμπτο και αυστηρό. Αλλά ε, στην περίπτωση των εσπεριδοειδών, ο κλάδος ε, έχει την αντίθετη αίσθηση. Ε, στη Νότια Αφρική υπάρχει πρόβλημα. Ε, έχουν αυξηθεί εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό σημαίνει, εσπεριδοειδών, ότι παρά τις ασθένειες που έχουν εξεσπάσει στη Νότια Αφρική, εξακολουθούμε να εισάγουμε τέτοια προϊόντα, εσπεριδοειδή και μεταδίδεται αυτή η ασθένεια και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτό. Και τελειώνω λέγοντας ότι θεωρώ πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και ε, σωστή την ε, πρότασή σας ε, για τη διαφάνεια και την εκτίμηση κινδύνου στη διατροφική αλυσίδα, να ενισχυθεί η ΕΦΣΑ, ο Οργανισμός για την Ασφάλεια Τροφίμων, πολύ καλά εργάζεται, αλλά να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια για να μην αμφισβητεί ο κόσμος τη δράση της. Είπατε κάτι και συμφωνώ Χρειάζονται νέοι πόροι, βεβαίω. Αυτά τα 62 εκατομμύρια που είπατε έτσι όφησαν να είναι και πιο διαφανής και πιο αποτελεσματικός. Αλλιώς δεν θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστώ τον κύριο Επίτροπο, τον κύριο Ντρουκάτη για όλα αυτά που μα είπε, αλλά και για το ότι ο συνήθω έρχεται εδώ, είναι Σε Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη δουλειά που έκανε για την Ξυλέλα. Μιλήσαμε για το θέμα αυτό την προηγούμενη εβδομάδα. Πρέπει απλά να επιταχύνεται. Θα αναφερθώ λιγάκι στο σημερινό θέμα. Του τελευταίους μήνε βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλέ επιμαχε θέσει που αφορούν στην αξιολόγηση των ευαίσθητων ουσιών. Δηλαδή κυρίως ε, γενετικά τροποποιημένοι ε, οργανισμοί, γλυφοσάτη ή ε, κάποιες αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, στην υγεία από διάφορες ενδοκρινείς ουσίες. Όλα αυτά ενέχουν τον κίνδυνο ότι δεν θα υπάρχει πλέον η ίδια αντικειμενικότητα στις μελέτες που χρησιμοποιεί ο Οργανισμός Ασφάλειας Τροφίμων. Οι πολίτες θέλουν μεγαλύτερη διαφάνεια και γι' αυτό εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον Επίτροπο το εξή. Πολλέ από αυτές τι μελέτε πληρώνονται από αυτόν που ζητάει να γίνει μελέτη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει μήπως να αλλάξει αυτή την αρχή του ποιο δηλαδή θα πληρώνει, αν θα πληρώνει ο ετών αυτός που ζητάει την ε, αξιολόγηση. Με τον τρόπο αυτό νομίζω ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια, κάτι το οποίο επιθυμούν διακαώ οι πολίτε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, και εγώ θα ήθελα να σε ευχαριστώ και εσάς και τους συνεργάτες σας ε, για τη δουλειά που κάνετε. Εγώ έχω μια πολύ ευθεία ειλικρινή ερώτηση. Γνωρίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δρομολογήσει μία έρευνα που αφορά ε, στην ε, σήμανση που χρησιμοποιείται στην Αγγλία. Θεωρούμε ότι αυτή δεν είναι μία σωστή ρύθμιση, γιατί όσον αφορά το κόκκινο, το κίτρινο, το πράσινο, αυτή η σήμανση δεν είναι σωστή θέλουμε να ενημερώσουμε τον πολίτη. Ε, δεν θέλουμε από εκεί να εξαρτάται η δική του απόφαση για αγορά ή όχι ενός προϊόντος. Ε, βέβαια κάνατε ένα βήμα προς τα μπρος ε, και θέλω να το αναγνωρίσω, αλλά γνωρίζουμε ή θέλω να ξέρω, μήπως θεωρείτε κι εσείς ότι θα πρέπει να υπάρξει κάποια αλλαγή που να αφορά στην προέλευση των πρώτων υλών, κάτι το οποίο μεταξύ άλλων το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το ζήτησε στην Ολομέλεια. Και νομίζω ότι αυτό αφορά οκτώ ε, χώρες ε, οι οποίες έχουν δρομολογήσει αυτήν ακριβώς ε, την κατεύθυνση, δηλαδή να είναι υποχρεωτική η αναγραφή προέλευσης των πρώτων υλών. <laughs> Η κυρία Ράς Γκαρσία, ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ανταλλαγή απόψε, κύριε Επίτροπε. Σε ό,τι αφορά προηγούμενη ερώτηση, για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουμε λόγω εισαγωγών από τρίτες χώρες. Η αναθεώρηση του κανονισμού του 2015 για την καταπολέμηση των επιβλαβών οργανισμών στα φυτά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε υποσχεθεί ότι μέσα σε δύο χρόνια θα καταρτήσει ένα κατάλογο των προϊόντων, μάλλον των απαγορευμένων ουσιών. Τι γίνεται, εκπονήθηκε αυτός ο κατάλογος, έχετε κάποια νέα στοιχεία. Επίσης, έχω μια ερώτηση για την ξυλέλα φαστιδιώσα. Δεν πρόκειται να παραιτηθούμε. Τι γίνεται, τι γνωρίζει για την προέλαση της ε, ασθένειας αυτής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τι μέτρα πρόκειται να θεσπίσετε για να αποφύγετε εξάπλωση της ε, αρρώστιας αυτής του επιβλαβούς οργανισμού ξυλέλα για να μην οδηγηθούμε σε ε, ανεπανόρθωτη βλάβη. Τέλος, οφείλω να ομολογήσω ότι είμαι απογοήτευσε ιδιαίτερα η ανικανότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αντιληφθεί πόσο σημαντικό είναι το θέμα της άμυνας στα τρόφιμα, food defense. Εδώ και καιρό ζητούμε ε, νομοθετικές διατάξεις για να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, ε, αγροτροφικές ε, για να μπορέσουν να εξάγουν στην Ιαπωνία, τον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πέρασε ε, πάνω από ένα χρόνο και δυστυχώ ε, εισακούστηκε το αίτημά μα. Ελπίζω στην επόμενη κοινοβουλευτική θητεία ε, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη δική τη θητεία να λάβει υπόψη αυτό το αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το food defense, την άμυνα στα τρόφιμα. Ο κύριο Ερντό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, φαντάζομαι δεν θα σας ε, ε, παραξενεύσει ούτε θα σας ε, εκπλήξει που θα σας μιλήσω για το μέλι που είναι το τρίτο πιο νοθευμένο προϊόν στην ευρωπαϊκή αγορά. 20% του εισαγόμενου μελιού από την Κίνα είναι νοθευμένο και ο κύριος Δεκάστρο το επισήμανε. Και αν δεν αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα στην ίδια την οδηγία, δεν πρόκειται να το επιλύσουμε. Κύριε Επίτροπε, σκοπεύετε μέχρι το τέλος της θητείας σας να αναθεωρήσετε τη σχετική οδηγία, να αλλάξουν οι νομοθετικές διατάξεις για να αποτραπούν τέτοια φαινόμενα νόθευσης προϊόντων. Κυρία Πετήρη, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Μήπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκέφτεται να συμπεριλαμβάνει και μία επισήμανση της ημερομηνίας σφαγής στα προϊόντα κρέατος. Για παράδειγμα, στην Κροατία έχουμε κρέας που εισάγουμε από άλλα χώρα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα κρέας που είναι κατεψυγμένο χρόνια ολόκληρα και δεν αποκλείεται να έχει μολυνθεί σε μερικές περιπτώσεις και με σαρμονέλα. Καλό θα ήταν λοιπόν στη σήμανση των προϊόντων κρέατος να αναφέρεται και η ημερομηνία της φαγής. Έτσι θα προστατεύσουμε τους καταναλώτες και θα διενεργήσουμε πιο αποτελεσματικό έλεγχο. Επίσης, ε, μία ερώτηση για τον έλεγχο εισαγόμενων οποροκυπευτικών από τρίτες χώρες σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται φυτοφάρμακα που απαγορεύονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας είπατε ότι τα κράτη-μέλη έχουν την ε, δυνατότητα να ελέγξουν τέτοιου είδου εισαγόμενα οποροκυπευτικά στα σύνορά τους και αν ε, θεωρήσουν ότι δεν πληρούνται οι προδιαγραφές να απαγορεύσουν τις σχετικές εισαγωγές. Αυτό έκανε η Κροατία, αλλά ε, δυστυχώς γίναμε στόχος ε, επικρίσεων και τελικά ανακλήθηκε το σχετικό μέτρο. Έχουμε όμως καθήκον να φροντίσουμε για την ασφάλεια των καταναλωτών και το δικαίωμά τους ε, να καταναλώνουν ασφαλή τρόφιμα και επίσης να μην υπόκειται σε του ανταγωνισμού η γεωργή μας, ο κύριος Χαϊτεμα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ με αυτό που προτείνετε σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό ασφάλεια τροφίμων, ότι θέλετε να δαπανίσετε περισσότερα χρήματα, αλλά για να πω και το λιγότερο που θα πω είναι ότι έτσι θέλει το πρόβλημα, ίσως μόνο τα συμπτώματα και με ανησυχεί ιδιαίτερα, γιατί το πρόβλημα πάει πολύ πιο βαθιά. Ε, βλέπουμε το χάρη ε, πολλέ μελέτε ε, που λένε ότι οι χημικέ ουσίε είναι καλέ ή κακέ, ή είναι επικίνδυνε ή όχι, αλλά από τη στιγμή που εγκρίνονται ασκείται κριτική. Και αν δεν εγκρίνονται δεν ασκείται καμία κριτική. Αυτό θεωρώ ότι είναι φαρισμένο. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί να μην κατηγορούμε τους ε, επιστήμονες για την αξιολόγησή τους γιατί είναι υποκριτικό το να αποδίδουμε την ευθύνη στους επιστήμονες ότι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους και όταν, παραδείγματος χάρη, ε, προκύπτει μια γνωμοδότηση που λέει απαγορεύεται μια χημική ουσία, σιωπή, μετά δεν ακούγεται τίποτα για την επιστήμη. Εξάλλου, αυτό δεν είναι μόνο ε, το υπευθυνότητα, το φταίξιμο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και το Κοινοβουλίο. Εμείς ως πολιτικοί θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί να μην αποδίδουμε ευθύνε στους επιστήμονες γιατί αν δεν έχουμε επιστήμονες τότε υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και τότε θα πρέπει να κάνουμε πολιτικές συζητήσεις για χημικές ουσίες. Δεν ξέρω τι ξέρουν οι συνάδελφοι αλλά εγώ τουλάχιστον δεν είμαι τοξικολόγος. Ε, δεν τα καταλαβαίνω μερικέ φορές ούτε καν ε, τις χημικές ονομασίε τίποτα. Αν λοιπόν του αρνηθούμε του επιστήμονε, μιλάμε για πλήρη καταστροφή. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι ε, η αύξηση του προπολογισμού του ΕΦΣΑ είναι καλή προσπάθεια για να ενισχύσουμε την δυνατότητα αξιολόγηση ε, κινδύνου. Σε ό,τι αφορά την Αφρικανική Πανόλη των Χείρων, όταν ε, είχαμε κρούσματα στην Εστονία, ήμουν τότε υπουργό. Και μας είπατε ήδη τι κάνατε, τι μέτρα λάβατε μέχρι στιγμής για την αντιμετώπιση Αφρικανικής Πανόλης των Χείρων. Αλλά μήπως θα μπορούσατε να σταθείτε λίγο περισσότερο στην κτηνιατρική πτυχή αυτού του φαινομένου και πόσο επιτυχεί ήταν η κτηνιατρική αντιμετώπιση της ε, επιζώτιας. Υπάρχει καμία ελπίδα να βρεθεί ε, είτε εμβόλιο είτε θεραπευτική ε, αγωγή για την αντιμετώπιση της αφρικανικής πανόλης των χείρων. Ευχαριστώ επίση του συναδέλφου που διοργάνωσαν πριν από δύο μέρε μια εκδήλωση, ένα σεμινάριο για την Αφρικανική Πανόλη των Χείρων. Ευχαριστώ. Κύριο Χόισλινγκ. Ε, κύριε Επίτροπε, ζητώ συγγνώμη που επανέρχομαι, αλλά δεν απαντήσατε στο ερώτημά μου και συγκεκριμένα στα νέο νοικοτινοειδή. Ε, τρία, τρεις ουσίες απαγορεύσαμε. Τώρα, ε, τα κράτη-μέλη που ζητάνε κάποια κατεξαίρεση ρύθμιση, εγώ είχα την εντύπωση ότι η απαγόρευση είναι απαγόρευση. Αλλά από ό,τι ακούω τελικά είναι μάλλον θέμα των κρατών μελών να ζητάνε την αδειοδότηση μιας ουσίας. Εγώ είχα την εντύπωση ότι ισχύει γενικά μια απαγόρευση, αλλά δεν μειώθηκε η συνολική ποσότητα των νεονικοτινοειδών. Όλοι πιστεύουν ότι δεν χρησιμοποιούνται πια, αλλά δεν ισχύει αυτό. Αν ε, κάποια κράτη-μέλη χρησιμοποιούν αυτές τις ουσίες, διερωτάται κανείς τελικά Μέχρι πού φτάνει μια απαγόρευση, τι γίνεται με το θέμα των απαγορεύσεων. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Επίτροπε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να σας υποβάλω ερώτηση και για όλα αυτά που μας είπατε σχετικά με την πανόλη των χείρων. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι, περισσότερο μία ρητορική ε, ερώτηση. Τα δικά σας τα προγράμματα ποια είναι, πότε θα έχει πάψει να ισχύει πλέον αυτή η κατάσταση που υπάρχει τώρα, γιατί δεν είναι τώρα τέσσερις οι χώρες, είναι έξι χώρες όπου παρουσιάζεται σε ένταση αυτό το φαινόμενο. Ίσως λοιπόν θα πρέπει να γίνει κάτι σαφέστερο, να καταδείξουμε στα κράτη-μέλη ε, μία λύση και θα ήθελα να αναφερθώ και στην πρόταση που κάνετε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή διεξάγονται διαπραγματεύσεις. Ε, προσπαθούμε να δούμε ε, πώς ε, θα μετακινούνται καλύτερα τα προϊόντα και όχι μόνο αυτό, αλλά ε, τα πλεονάσματα μια χώρας ε, να χρησιμοποιούνται ίσω κάπου αλλού για την προστασία του περιβάλλοντος. Τελικά θέλω να ρωτήσω τι γίνεται με τι ε, τιμέ των τροφίμων. Μήπω και εκεί δεν πρέπει να γίνουν κάποιες προσπάθειες. Μήπω δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι προδιαγραφέ προστασία τη υγεία, αλλά και παραγωγή. Γιατί αν τελικά έχουμε μία αγορά θα πρέπει να έχουμε και ενιαίε προποθέσει. Στην Ευρώπη ε, γίνονται τεράστιες επενδύσεις για ποιοτική παραγωγή και εισάγονται ε, προϊόντα που έχουν παραχθεί με αθέμητο ανταγωνισμό. Κύριε Επίτροπε, ε, δεν άκουσα την παρουσίαση. Θα κάνω περισσότερο σχόλιο και όχι τόσο ερώτηση. Νομίζω ότι το θέμα της, του προγράμματος για την υγεία είναι πολύ σημαντικό λόγω της κλιματικής αλλαγής. Είχα μία ε, ένα τηλεφώνημα που με ανησύχησε πάρα πολύ και ένα από τα πράγματα που με ανησυχεί είναι ότι δεν θέλουμε στην Ευρώπη να απαγορεύουμε ε, κάποιες ζωές, αλλά ενδεχομένως μερικές φορές κάποιες χημικές ουσίες πρέπει να τις επιτρέπουμε. Η αναλογικότητα είναι σημαντική. Ε, για το θέμα των τσιγάρων. Εκεί, ναι, να τα απογορέψουμε, αλλά σε κάποιες άλλες περιπτώσεις να έχουμε και κάποιο απόθεμα κάποιων χημικών ουσιών για να αντιμετωπίσουμε προβλήματα που πραγματικά υπάρχουν. Ευχαριστώ. Δύσκολο είναι να είμαστε λακωνικοί με τέτοια πληθώρα ερωτήσεων που καλύπτουν τόσο μεγάλο φάσμα και είναι και τόσο περίπλοκες. Ας ξεκινήσουμε από την κυρία Γκιλέρα. Μιλήσατε για τις ε, σημαντικές ε, προδιαγραφές και τις, την ενίσχυση των προτύπων στη νέα νομοθεσία και μάλιστα ιδιαίτερα για τα εισπεριδοειδή. Έχουμε λάβει σχετικά μέτρα για τρίτες χώρες που έχουν εντοπιστεί επιβλαβείς οργανισμοί και συνεχίζονται οι συζητήσεις. Και το ίδιο ρώτησε και η κυρία Ράς Γκαρσία, τι γίνεται με τον κατάλογο με τις απαγορευμένες ουσίες. Φυσικά συζητούμε τα κράτη-μέλη την υποχρέωσή τους να μας παρουσιάσουν αυτό το κατάλογο των απαγορευμένων ουσιών. Συνεχίζονται ακόμη συζητήσει με όλους τους ε, ενδιαφερόμενους, που είναι 28 προς το παρόν ακόμη. Ε, δεν είναι εύκολα τα πράγματα, αλλά προσπαθούμε να το καταφέρουμε. Για την ξυλέλα φαστιδιώσα. Κύριε Καπούτο, μας ρωτήσατε για την ξυλέλα, τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς, τους ενδοκρινικούς ε, μετα... Ε, διαταράκτες και το πόσο γλυφοσάτη είναι τέτοιος ενδοκρινικός διαταράκτης. Δεν ε, υπάρχουν σχετικές αξιολογήσεις για τους μη, κυβερνητικ... μη, μη γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς και τη γλυφοσάτη. Και ο μεγάλος αριθμός αιτήσεων που, που ετησίως λαμβάνει η ΕΦΣΑ είναι καλό παράδειγμα της ικανότητας του ΕΦΣΑ να αντιμετωπίσει αυτά τα θέματα. Η συντριπτική πλειοψηφία των ετούντων δεν αφορούν επίμαχα θέματα, ούτε ε, απαιτούν ε, παρέμβαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχει μεγάλος αριθμός μελετών που στηρίζει την εφαρμογή τέτοιων θέμα των τέτοιων ουσιών. Μιλήσατε για το οικονομικό μοντέλο. Υπάρχει εγγενής δυσκολία ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο ΕΦΣΑ ή οι δημόσιες αρχές θα επιλέξουν το συγκεκριμένο εργαστήριο με διαγωνισμό, με ανοιχτέ διαδικασίες και τι ποσό θα καταβάλουν για την διεξαγωγή των μελετών. Δεν είμαστε έτοιμοι προς το παρόν να τροποποιήσουμε το χρηματοοικονομικό μοντέλο, που είναι πολύ περιπλοκό ήδη. Πάντως, για το θέμα της σήμανσης, συμφωνώ μαζί σας, κύριε Ντεκάστρο, ότι ήρθε επιτέλους η ώρα να συζητήσουμε αυτά τα θέματα της επισήμανσης. Ίσως θα μπορούσαμε να οργανώσουμε σχετικές συζητήσεις ε, για τη πιθανότητα μιας πανευρωπαϊκής σήμανσης. Ε, ε, να έχουμε το Made in EU με επιμέρου αναφορά ε, της χώρας, Γερμανία, Λιθουανία, αλλά με το πανευρωπαϊκό σύστημα ευρωπαϊκό προϊόν, made in EU. Τώρα έχουμε την 25η επέτειο της ενιαίας μας αγοράς. Ιδανική ευκαιρία λοιπόν να συζητήσουμε και αυτά τα θέματα της σήμασης. Είμαστε έτοιμοι για ένα πανευρωπαϊκό σήμα μαζί με την χώρα προέλευσης, γιατί θα θέλαμε να αναφέρεται και χώρα προέλευσης, πέραν του σήματος του ευρωπαϊκού προϊόντος, αλλά σε ένα ενιαίο πλαίσιο, όπως και για το ευρώ. Το κάθε ευρώ ε, έχει και ε, ένα, μια, ένα εθνικό σύμβολο, παρόλο που το ευρώ είναι ενιαίο νόμισμα. Είναι σημαντικό κάτι αντίστοιχο να έχουμε και στα σήματα, να έχουμε ένα πανευρωπαϊκό σήμα το ευρωπαϊκό προϊόν με αναφορά και τη συγκεκριμένη χώρα προέλευση. Νομίζω ότι είναι ιδανική στιγμή να συζητήσουμε και αυτά τα θέματα. Η κυρία Ραν Καρσία ε, επίση ε, έθεσε παρόμοια θέματα. Τα απάντησα όμω για το μέλι, κύριε Ερντό, για το μέλι και την οθεία του μέλιου. Όντως είναι πρόβλημα η νοθεία στο μέλι. Είναι πολύ επιρρεπές αυτό το προϊόν και το στην οθεία. Είχαμε πολλές συζητήσεις και ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι να αντιμετωπιστεί αυτή η νοθεία. Απλώς θα πρέπει να ενισχυθούν οι έλεγχοι στα εισαγόμενα προϊόντα στην ευρωπαϊκή αγορά και θα πρέπει να αφιερωθούν περισσότεροι πόροι και έμψυχοι και οικονομικοί για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη σημαντική πρόκληση της νοθείας. Πάντως, αλλαγές νομοθετικές δεν προβλέπονται προς το παρόν. Καλύτερα να βελτιώσουμε τα υπάρχοντα νομοθετικά μέσα και ζητούμε από τα κράτη-μέλη να το κάνουν. Τώρα για την ξυλέλα. Το θέμα της ξυλέλας είναι επικίνδυνο. Η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία είναι τρεις χώρες οι οποίες έχουν παρατηρηθεί κρούσματα ξυλέλας και σε κάποια θερμοκήπια της Γερμανίας. Πάντως η Ισπανία αντιμετωπίζει πολύ ε, αποτελεσματικά το, ε, τον ε, επιβλαβή, οργανισμό, αλλά πρόβλημα έχουμε στην Ιταλία που δεν εφαρμόζονται επαρκώς συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της ξυλέλας. Τώρα προσπαθούμε να συνεργαστούμε με την Ιταλία και να θεσπίσουμε και ένα εθνικό, όχι μόνο περιφερειακό σχέδιο αντιμετώπιση. Τώρα έχει αναλάβει νέα Ιταλική κυβέρνηση και ελπίζω να αντιμετωπίσει πιο αποτελεσματικά. Δεν υπάρχει προς το παρόν θεραπεία ε, του οργανισμού, μόνο ε, κοπή των ε, δέντρων που έχουν προσβληθεί. Και αυτό είναι δύσκολο για τους ε, ελαιοπαραγούς να το δεχτούν, ότι θα χάσουν τα δέντρα τους. Ε, Πάντω, η μόνη στρατηγική για την ε, εξουδετερώση τη ξυλέλα είναι η εκρίζωση προ το παρόν και ζητούμε από την Ιταλία να ενεργοποιηθεί περισσότερο στην αντιμετώπιση. Τώρα να απαντήσω στον άλλο συνάδελφο. Να, να απαντήσω για αυτό που ρωτήσατε για την Αφρικανική Πανόλη του Χείρου. E, και πώς θα εκριζωθεί ε, και θα εξαλειφθεί αυτή η νόσος. Ακούσαμε διάφορους επιστήμονες, και αυτό τον καιρό γίνονται έρευνες για να βρεθεί εμβόλιο κατά του ιού της Αφρικανικής Πανόλης, του χείρου. Αλλιώς μόνο βιοασφάλεια ε, δηλαδή να έχουμε μια στρατηγική ε, αντιμετώπιση της θύρας με ενημέρωση των κυνηγών, κυνηγάν αγριούρουνα και να ε, σταματήσει η λαθροθυρία και το λαθρεμπόριο. Ε, δηλαδή είναι ανθρωπογενή τα προβλήματα. Μέχρι τώρα δεν έχουμε επιβάλει πιο περίπλοκα μέτρα, γι' αυτό είναι δύσκολο να αντιμετωπίσουμε αυτή την ασθένεια. Και είναι αρνητικό παράδειγμα. 40 χρόνια τώρα δεν έχει αντιμετωπιστεί, γιατί πριν από 40 χρόνια εμφανίστηκε στην Ευρώπη η Αφρικανική Πανόλη του χείρου και δεν αφορά ε, μόνο τα, τους αγριόχειρους, ε, αλλά και 20 τους χείρους που ε, κυκλοφορούν αδέσποτοι γιατί έχουν φύγει από τα σπίτια ή από τις εκτροφές και μεταδίδουν την νόσο και δεν κάνει κανείς ε, τίποτα στη διοίκηση, δεν κυνηγάνε τα ζώα αυτά, δεν τα θανατώνουν, δεν εφαρμόζονται τα μέτρα. Στην Ισπανία επίσης υπήρξε κρούσμα, αλλά αντιμετωπίστηκε με τρόπο πολύ αποτελεσματικό. Ήταν ένα πρόβλημα που χρόνιζε, αλλά τελικά λήφθησαν μέτρα για να περιοριστεί αυτό το κρούσμα. Δυνατότητες υπάρχουν, αν κανείς εφαρμόζει βέβαια πάντα σωστά τα μέτρα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ε, ε, όλη την Ήπειρο συνεχίζεται και προς Ανατολάς. Από το Καλίνιγκρατ μέχρι το Ιρκούτσκ δεν μπορούμε 100% να εξασφαλιστούμε γιατί δεν υπάρχει εμβόλιο. Άρα εκ των ενόντων θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με τα ε, κείμενα μέτρα και αυτό δεν μπορώ να σας δώσω και καμία πρόγνωση για ε, την κρίζωση της Αφρικανικής Πανόλης του χείρου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιτύχει κάποια πράγματα στον έλεγχο αλλά έχουμε και 10.000 χιλιόμετρα σύνορα χερσαία με τη Ρωσία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μπορούμε να ελέγξουμε τα σύνορα γιατί είναι μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα ε, αλλά εκτό τη Ένωσης και ε, αφήστε δε που μπλέκονται και διάφορα υπουργεία για τις προδιαγραφές και δεν είναι μόνο το Υπουργείο Γεωργίας. Σας διαβεβαιώ λοιπόν ότι υπάρχουν μέτρα, αλλά υπάρχουν και οι τρίτες χώρες. Αν έχουν ε, δικαίωμα τώρα οι τρίτες χώρες εισάγουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορούν να το κάνουν μόνο εφόσον έχουν πιστοποίηση, έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό το πιστοποιητικό περιλαμβάνει όλες τις απαιτήσεις που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορούν τη χώρα αυτή και όλες τις εταιρείες. Βραζιλία, Ινδία, και κάθε τρίτη χώρα. Και γίνονται και έλεγχοι σε τακτά χρονικά διαστήματα, χορηγείται το πιστοποιητικό και σε περίπτωση παράβασης ε, αφαιρείται. Δηλαδή, όταν έχουμε συμφωνίες με τρίτες χώρες, αυτό δεν σημαίνει ασυδοσία για τον κάθε εξαγωγέα. Ε, υπάρχουν κανόνες. Και γι' αυτό δεν είναι και απλή η υπόθεση για ε, τους παραγωγούς και για τους εμπόρους και τους εξαγωγείς. Έχουν πολύ αυστηρές προδιαγραφές. Το ίδιο ισχύει κατά κάποιο τρόπο και για την ερώτηση που έκανε η κυρία από την Κροατία, η κυρία Πέτυρ, για τους ελέγχους. Για τα απορροκυπευτικά. Θέλω να σας διαβεβαιώσω κι εγώ ότι είναι υπό έλεγχο η κατάσταση. ακούστηκαν κάποια μέτρα, τα οποία δεν ήταν καθόλου εύκολο να εγκριθούν. Θα το ελέγξω και θα σας απαντήσω γραπτός, αν θέλετε. Για τις γενικές τώρα προδιαγραφές και τα πρότυπα, ιδιαίτερα ε, αυτά που ισχύουν στα σφαγεία εφαρμόζονται. Υπάρχουν πάρα πολλοί σαφείς κατευθυντήρες γραμμές υποχρεωτικής ε, τήρησης για όλες τις εταιρείες που έχουν σφαγεία και υπάρχουν και αρμόδιες ελεγκτικές αρχές που κάνουν καλά τη δουλειά τους. Δεν μπορείς να ανοίξει σφαγείο ως επιχείρηση έτσι χωρίς να πάρεις άδεια και άδεια παίρνει μόνο εφόσον τηρείς κάποιες προϋποθέσεις και προδιαγραφές. Σε περίπτωση που υπάρξει ένα περιστατικό είναι επεισόδιο και καταγγέλλεται, ε, επεμβαίνουν οι ελεγκτές και αφαιρούν την άδεια λειτουργίας από το σφαγείο. Ε, όλα αυτά λοιπόν δεν είναι έτσι ανεξέλεγκτα και ασίδωτα. Ε, ε ρώτησε κάτι ένας ε, βουλευτής από την Εστονία, ο κύριος Πάντα, για το αν υπάρχουν φάρμακα κατά της πανόλης, της αφρικανικής πανόλης του χείρου. Εμβόλιο δεν υπάρχει ακόμα. 16 εκατομμύρια ευρώ ε, δόθηκαν σε επιστήμονες για να απτύξουν το εμβόλιο. Δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έχει στεφθεί αυτό με επιτυχία. Δεν μπορώ να σας δώσω οριστική απάντηση. Σε περίπτωση που υπήρχε εμβόλιο, φυσικά θα το είχαμε χρησιμοποιήσει ευρύτατα. Άλλη ερώτηση από τον κύριο Χόισλινγκ για τη λεγόμενη έγκριση για περιπτώσεις εκτάκτης ανάγκης, emergency authorization. Έχετε δίκιο. Σε 7 χώρες ε, κάναμε ελέγχου που ακολουθούν την πρακτική αυτή. Υπάρχουν ε, διαδικασίες έτσι ταχείας έγκρισης ε, επιπλέον μέτρων. Ο Οργανισμός Ασφάλειας Τροφίμων ΕΦΣΑ κάνει αυτό τον καιρό κάποιες μελέτες και ελέγχου. Έχουμε ζητήσει από τις χώρες αυτές ενημέρωση και τεκμηρίωση γιατί θα πρέπει να αποδείξουν εάν έχουν συμμορφωθεί με την νομοθεσία. Να το τεκμηριώσουν και να το αιτιολογήσουν ε, πρέπει οι χώρες και εξακολουθούν οι έλεγχοι. Και οι κανόνες στο μέλλον θα γίνουν ακόμα πιο αυστηροί, έτσι ώστε οι χώρες που θέλουν να χορηγήσουν άδεια για έκτακτες λεγόμενες περιστάσεις να τηρούν ε, την υποχρέωση κοινοποίηση. Δηλαδή πρώτα να διαβιβάζουν τα στοιχεία και μετά να λαμβάνουν την απόφαση. Αλλιώς υπάρχει η δυνατότητα και ακόμα και η πιθανότητα κατάχρησης ιδιαίτερα αυξημένη. Εφτά χώρες ήταν αυτές, είμαστε παρόντες εκεί σε αυτές τις εφτά χώρες και απαιτούμε και απάντηση. Ε, πώς ελήφθη αυτή η απόφαση και είναι, αν είναι αρκετά δικαιολογημένη και τεκμηριωμένη και ανάλογα με το αποτέλεσμα θα δούμε τι θα κάνουμε. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε την ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο Άντριο Κάιτες, ο οποίος διεξοδικά απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις των Ευρωβουλευτών. Επαναλαμβάνει ο Πρόεδρος. Ολοκληρώσαμε τη σύντηση μετά από διεξοδική απάντηση των ερωτήσεων των Ευρωβουλευτών. Έγκυψαμε σε μία σειρά θεμάτων και διεκπαιρεώσαμε αυτό το σημείο της ημερήση διάταξης. Ευχαριστούμε θερμά τον Επίτροπο για την πολύ χρήσιμη αυτή και επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων. Μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ενήμεροι για τα τρέχοντα θέματα. Σας ευχαριστούμε θερμά και πάλι κύριε Επίτροπε. Περνάμε τώρα με κάποια καθυστέρηση στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, ευχαριστώντας και αποχαιρετώντας τον Επίτροπο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης είναι το σημείο 10 που προβλέπει ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Άντριο Μακντάουελ, αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, με θέμα τις επενδύσεις στη γεωργία και την βιοοικονομία. Καλωσορίζω θερμότατα τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Θα μας μιλήσει για τις επενδύσεις ε, στη γεωργία και τη βιοοικονομία. Καλώς ήρθατε κύριε Αντιπρόεδρε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 Τράπεζα Επενδύσεων. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στηρίζει την αγροτική οικονομία και εξασφαλίζει παροχή τεχνικών συμβολών και αρρωγής. Ε, Συμβάλλοντας σε μια νέα προσέγγιση ε, και στα θέματα της γεωργίας και των τροφίμων. Περιμένουμε λοιπόν πληροφορίες από τον Αντιπρόεδρο της ΕΤΕΠ. Πληροφορίες που θα μας βοηθήσουν στην περαιτέρω συζήτηση για τη μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής και μετά το 2020. Θα σας δώσω το λόγο λοιπόν κύριε Πρόεδρε. Εκφράζοντας την ικανοποίησή μου εκ των προτέρων για την καρποφόρα συζήτηση που θα έχουμε. Thank you very much, Chairman, for the um, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για την πρόσκληση που μου απευθύνατε να έρθω στην Επιτροπή σας και ευχαριστώ πολύ και για τα πολύ καλά σας λόγια. Επιτρέψτε μου όμως να ξανασυστηθώ. Λέγομαι Άντρου Μακτιλέν και είμαι αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και είχα την τιμή να ασχολούμαι με τα γεωργικά θέματα από τον Δεκέμβριο όπου αποσύρθηκε ο προκάτοχός μου από την τράπεζα και επίσης ασχολούμαι και με θέματα ενέργειας μεταξύ άλλων, μεταξύ κάποιων άλλων θεμάτων με τα οποία ασχολούνται η τράπεζα. Έχω κοντά μου τον κύριο Μπέρνερ Σπιτ, τον παρακαθήμενο, είναι διευθυντή για θέματα περιβάλλοντος και βιώσιμη ε, ανάπτυξης, ενταφικής ανάπτυξης. Ε, είναι αρμόδιος επίσης για την πολιτική χορηγήσεων για γεωργικά δάνεια. Ε, χαιρόμαστε που είμαστε εδώ και για μένα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία εκ μέρου της διαχείρισης, της διεύθυνση να σας εξηγήσω ε, τη δική μας την ε, δέσμευση απέναντι στην στήριξη και την ευημερία του γεωργικού τομέα. Ο προκάτοχός μου, ο κ. Πέλεκαν, είχε έρθει πριν από τρία χρόνια περίπου στην Επιτροπή σας και έχει έρθει και στιγμή να σας ενημερώσω για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στον τομέα αυτό. Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να πω κάποια λόγια γενικά για τον οργανισμό μας. Ε, δεν θα ε, διαβάσω, θα πω μόνο μερικά πράγματα και μετά θα δεχτώ ερωτήσεις. 60η φέτος, εφέτος, ε, για την τραπεζά μας προβλεφθήκαμε από την συνθήκη της Ρώμης, από τα κράτη-μέλη. Ανήκουμε στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκπροσωπούνται στην τράπεζα τη δική μας. Ε, πριν από 60 χρόνια είχαμε έδρα στις Βρυξέλλες, 10 χρόνια μείναμε στις Βρυξέλλες, μετά μετακινηθήκαμε στο Λουξεμβούργο. 4 δις ε, πριν από 60 χρόνια ήταν η πρικοδότησή μας. Ε, ήταν ε, ένα πολύ σημαντικό δώρο από τα έξι ιδρυτικά μέλη. Αυτό το αρχικό κεφάλαιο, τα τέσσερα δις, ε, με την βοήθεια του γεγονότος ότι δεν καταβάλουμε μέρισμα στα κράτη-μέλη και δεν φορολογούμε τα, πρέπει να είμαι απόλυτα φορολογής επ' αυτού, τα τέσσερα δις ευρώ μέσα από αρκετές χορηγήσεις τα τελευταία χρόνια, τα φτάσει στα 600 δις, έκτοτε μόνο το 12 δεχτήκαμε μία χρηματοδοτική ένεση, περίπου 12 ε, δις ε, που επενδύθηκαν στην ε, τραπεζά μας. Δεν έχουμε καμία χρηματοδότηση από τον προϋπολισμό μόνο όταν πρόκειται για συγκεκριμένα θέματα και θα επανέλθω επ' αυτού. Γίναμε λοιπόν ο μεγαλύτερος δανειοδότης του κόσμου. Αυτό δεν αναφέρεται συχνά, αλλά αυτή η Τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο μεγαλύτερος χορηγός δανείων ανά τον κόσμο δάνεια που ανέρχονται σε 78 δις ε, και αν θέλετε σε σχέση με την Παγκόσμια Τράπεζα μιλάμε για διπλάσιο όγκο χορηγήσεων. Το 90% παραμένει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα 10% χορηγείται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με βάση τις συνθήκες, το καθήκον μας είναι να προσφέρουμε την χρηματοδότηση και την εμπειρογνωμοσύνη μας ε, σε βιώσιμα προγράμματα, τα οποία στηρίζουν τους στόχους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρία θέματα συγκεκριμένα. Έχουμε τις χορηγήσεις δανείων, που τώρα έχει επεκταθεί αυτό, ε, δεν επενδύουμε μόνο παραδοσιακά, αλλά και σε μετοχικό κεφάλαιο και έχουμε και εγγυήσει προσφέρουμε εγγύησει. Κατ' ουσίαν εκεί αναλαμβάνουμε κάποιους κινδύνους και αυτό το κάνουμε και μέσα από την τραπεζά μας και μέσα από την θηγατρική μας, ε, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Η δεύτερη ευθύνη μας είναι ένα είδος μείγματος. Δηλαδή, ξε, διπλώνουμε, ξεκλειδώνουμε κάποια χρήματα, κάποια κονδύλια, τα συνδυάζουμε και με άλλα κονδύλια, τα οποία λαμβάνουμε από οργανισμούς εκτός Ευρωπαϊκή Ένωσης. Ο τρίτο τομέα με τον οποίο ασχολούμεθα είναι η παροχή συμβουλών. Είναι το τρίτο εργαλείο που χρησιμοποιούμε για να στηρίζουμε τις επενδύσεις. Προσφέρουμε τεχνική αρρωγή και άλλες συμβουλευτικές υπηρεσίες ε, για να μπορούμε να ξεπεράσουμε τους φραγμούς στι ε, επενδύσει. Αυτό για πολύ καιρό ήταν η ευθύνη μα ε, και τώρα έχουμε αναλάβει και την ευθύνη για το European Advisory Hub υπό το Εκεί ε, συγκεντρώνονται όλοι οι επενδυτές και προσπαθούμε να τους κατευθύνουμε στους ε, σωστούς ε, τομείς. Σαφώς και είμαστε εμπορική τράπεζα πρέπει να έχουμε κέρδος στις επενδύσεις μας γιατί δεν χρηματοδοτούμεθα από τον προϋπολογισμό. Τα χρήματά μας τα αντλούμε από την ε, κεφαλαγορά και από τις τράπεζες αλλά οι δικές μας επενδύσεις πρέπει κατά κύριο λόγο να έχουν νόημα οικονομικό, να μην απαραίτητα 100% κερδοφόρες, να είναι επενδύσεις σε πολιτικές που είναι συμβατές με αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς χρηματοδοτούμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις παραμένει μια μεγάλη πρόκληση στην Ευρώπη. Παρεπιπτόντως, αυτό περιλαμβάνει και γεωργικούς συνεταιρισμού μέχρι 3.000 ε, υπαλλήλους. Στηρίζουμε την οικονομική και την κοινωνική συνοχή, την περιφερειακή ανάπτυξη και προφανώς ε, στηρίζουμε ε, την κλιματική αλλαγή, συγκεκριμένες δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, ε, θέματα που έχουν σχέση με την καινοτομία. Βεβαίως η αξιολόγηση για μας είναι 3α, χορηγούμε δάνεια μακροπρόθεσμα με χαμηλά επιτόκια για μεγάλο χρονικό διάστημα Άρα δηλαδή αυτό είναι καθαρά το δικό μας το επιχειρηματικό μοντέλο. Το δικό μας το όφελος το μετατρέπουμε στους, το μεταφέρουμε μάλλον, το μετακυλίουμε στους δικαιούχους. Δεν θέλουμε βεβαίως να εκτοπίσουμε τον ιδιωτικό τομέα, γιατί είναι σαφές. Εμείς είμαστε συμπληρωματικοί προς τον ιδιωτικό τομέα. Δεν θέλουμε να εκτοπίσουμε τον ιδιωτικό τομέα, αλλά να λειτουργούμε παράλληλα, να αναλαμβάνουμε κινδύνους που ξεκλειδώνουν κάποιες επενδύσεις. Ε, χρησιμοποιούμε τα δικά μας κεφάλαια, έχουμε αποθέματα τα οποία έχουμε συγκεντρώσει τα τελευταία 60 χρόνια μέσω των δραστηριοτήτων μας, αλλά περίπου όλο και περισσότερο ένα τρίτο των χορηγήσεών μας στηρίζονται από αυτό που αποκαλούμε mandates, εντολές αν θέλετε, που λαμβάνουμε κυρίως από τον ενωσιακό προϋπολογισμό. Χρησιμοποιούμε το ε, κεφάλαιο κινδύνου ένα πρόγραμμα που είναι πολύ σωστό που μας στηρίζει είναι το ΕΦΣΙ, το πρόγραμμα για στρατηγικές επενδύσεις. Αυτό είναι μια κεντρική εντολή, αλλά παίρνουμε εντολές και από άλλες διαχειριστικές αρχές για να δανειδετούμε ε, στις δικές τους αρμοδιότητες. Όσον αφορά τις εντολές που δεχόμεθα, όταν πρόκειται για χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είμαστε υπόλογοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Όταν ε, χρηματοδοτούμε απαιτούμε δράσεις ε, όπου λαμβάνουμε χρήματα από τα κράτη-μέλη, τότε ο μηχανισμός λογοδοσίας είναι τελείως διαφορετικός. Θα ήθελα λιγάκι να μιλήσω για την τράπεζά μας και τη Γεωργία. Πρέπει να πούμε ότι η δική μας η τράπεζα δεν συνδεόταν με την Γεωργία στον ίδιο βαθμό όπως συνδεόμαστε με όλους τους τομείς, όπως με τις υποδομές ή την μεταποίηση ή την ενέργεια. Αυτό τα τελευταία 60 χρόνια. Και υπάρχει και συγκεκριμένος λόγος γιατί. Παραδοσιακά λοιπόν τα δικά μας ε, τα μέλη, τα κράτη-μέλη μέσα από το Διοικητικό Συμβούλιο και το Προεδρείο ε, θεωρούσαν ότι στηρίζεται η Γεωργία μέσα από την κοινή γεωργική πολιτική και ότι δεν χρειάζεται η Γεωργία τη δική μας τη χρηματοδότηση. Και λόγω της φύσης της κοινή γεωργικής πολιτικής οι περισσότερες επενδύσεις ε, χρηματοδοτούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς όμως να είναι οικονομικές όπως στις τις χαρακτηρίζουμε εμείς. Δηλαδή είναι επενδύσεις οι οποίες δεν είναι οικονομικές με τη στενή έννοια του όρου. Ως εκ τούτου δεν ε, κάλυπταν τις δικές μας, τις, τα δικά μας τα προαπαιτούμενα. Τέλειωσαν, μάλλον με συγχωρείτε, άλλαξαν όλα αυτά την τελευταία δεκαετία υπάρχουν αλλαγέ και μεταρρυθμίσει που έλαβαν χώρα στον τομέα της γεωργίας. Τώρα πλέον πολλές από τις επενδύσει που προάγονται τώρα ε, καλύπτουν τα δικά μας τα κρατήρια επιλεξιμότητας και γι' αυτό το λόγο πλέον η τράπεζα εμπλέκεται με τον τομέα της γεωργίας. Και είναι και προφανές, έχουμε αναγνωρίσει ότι η γεωργία, η, τα τρόφιμα είναι ένα μεγάλο κομμάτι της Ευρώπης με πάρα πολλές θέσεις απασχόλησης, ε, το 9% νομίζω των θέσεων εργασία που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν και η Τράπεζα αποφάσισε να στηρίξει αυτόν τον τομέα. Αποφασίσαμε επίσης ότι σε γεωργικές περιοχές ζουν νομίζω περίπου 55% των πολιτών. Ως εκ τούτου μια άλλη υποχρέωση της ε, τράπεζας, όπως είπα προηγουμένως, είναι και η κλιματική αλλαγή. Αναγνωρίζουμε τον ειδικό ρόλο που παίζει η γεωργία και η βιοοικονομία και θα παίξει στο να ε, επιτευθούν οι πολύ φιλόδοξοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία του κλίματος και του περιβάλλοντος. Αλλάζουμε λοιπόν. Μας ενδιαφέρει περισσότερο η γεωργία. Το τι κάνουμε. Ξεκινήσαμε με ένα μνημόνιο συναντήληψης ε, το 2014 μετά από αίτημα τότε του Επιτρόπου Φιλ Χόγκαν. Και εκεί καθορίστηκαν οι τομεί όπου θα συνεργαζόμασταν περισσότερο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καθορίστηκαν επίση τα εργαλεία που θα χρησιμοποιούσαμε. Και εσωτερικά την τράπεζα, αναδιοργανωθήκαμε, ο Βέρνερ είναι με αυτό. Ε, υπάρχουν τομείς ε, που έχουν σχέση με τη γεωργία και κλείτσαν όλοι αυτοί να έχουν μία ε, συγκεκριμένη πολιτική. Έχουμε πολλά εργαλεία για να στηρίξουμε τον τομέα. Βεβαίως έχουμε ένα μηχανισμό άμεσων διανδιωτήσεων για μεγάλα προγράμματα, corporates, και αυτά αφορούν επενδυτικά προγράμματα πάνω από 25 εκατομμύρια. Εμείς ε, χρηματοδοτούμε τα μέλη ε, άμεσα, αναλαμβάνουμε άμεσα τον κίνδυνο. Πρόσφατα δώσαμε 55 εκατομμύρια σε ένα συνεταιρισμό γαλακτοπαραγωγικό για να ε, έχει παστεριωμένο γάλα υψηλής θερμοκρασίας. Είναι μια καινοτόμα διαδικασία ε, επίσης, 150 ε, εκατομμύρια δώσαμε σε μια εταιρεία σουηδική ε, στον δασοκομικό τομέα για να ξυγχρονιστεί και αυτή στην επεξεργασία του ξύλου. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ένα από τα πιο σημαντικά, τις πιο σημαντικές επιπτώσεις του ΕΦΣΙ ήταν ναι, και στη χρηματοδότηση. Πολλές αγροτικές δραστηριότητες για μας είναι κρίνονται επικίνδυνες, δεν είναι παραδοσιακέ. Το έψι όμως πλέον μας επιτρέπει να αναλαμβάνουμε επιχειρηματικό κίνδυνο. 22 οι άμεσε επενδύσει μας, με πολλά μείγματα, τρία δις το σύνολο των επενδύσεων, κυρίως ε, σε μεγάλα προγράμματα ε, και υπάρχουν και άλλες 15 ε, δράσεις που εξετάζονται. Για μικρότερες δραστηριότητες, γιατί μιλάμε για ένα τομέα όπου κυριαρχούν κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εκεί έχουμε ένα πλεονέκτημα ε, συνεργαζόμαστε με τοπικές τράπεζες ε, και άλλους ενδιάμεσους. Δηλαδή, εμείς χρηματοδοτούμε τους ενδιάμεσους και αυτοί δίνουν περαιτέρω τα δάνεια με πολύ χαμηλά επιτόκια μέχρι τον τελικό δικαιούχο. Επίσης, ε, αυτό που κάνουμε είναι ότι όλο και περισσότερο επιμερίζουμε τον κίνδυνο των ε, δανείων. Αν θέλετε μπορούμε να επανέλθουμε αυτό στη συζήτηση. Και όλο και περισσότερο προσφέρουμε με το κεφάλαιο. Με το κεφάλαιο μέσα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων το οποίο ε, προσφέρει ε, χρηματοδότηση σε επιχειρηματικό κεφάλαιο δεν το κάνουμε αυτό μόνο μέσα από τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, χρηματοδοτούμε και κυβερνήσεις στα ε, διάφορα προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης και της γεωργίας. Δηλαδή τα κράτη-μέλη προφανώς ε, έχουν τη δική τους συγχρηματοδότηση και το ποσοστό τους και εμείς βοηθούμε με δάνεια τις κυβερνήσεις να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. 1,35 δις ας πούμε στην Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, Ρουμανία, πιο πρόσφατα στην Πορτογαλία. Επίσης, ε, δώσαμε δάνειο στη χώρα για αρδευτικά έργα και καταπολέμηση της απερίμωσης. Και όλο και περισσότερο συνεργαζόμαστε με διαχειριστικές αρχές, με μικροδάνεια και άλλα χρηματοδοτικά μέσα. Από τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ε, από εκεί έχουν επιδοτήσεις, αλλά εμείς χορηγούμε δάνεια. Έχουμε και συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχουμε ε, και σε τράπεζες και σε διαχειριστικές αρχές για να αναβαθμίσουν τη δυνατότητά τους να δανειοδοτούνται, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον αγροτικό τομέα. Όλα αυτά τα μέσα έχουν αρχίσει να λειτουργούν από το 2012 μέχρι το 2017. Χρηματοδοτούμε δάνεια και με της τάξης των 33 δις μαζί με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων ε, το θηγατρικό μας και αυτή η χρηματοδότηση ε, κινητοποίησε περίπου 100 δισεκατομμύρια επενδύσεων σε όσους υποστηρίζουμε στη βιοοικονομία. Το 2016 ήταν στο Ζενίθ με ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό Πολύ Το 2012 ε, ήταν 3 ε, εκατομμύρια και το 2016 ε, διπλασιάστηκε. Δεν ξέρω τι θα προκύψει από τη συζήτηση για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτό είναι δική σας δουλειά, δικά, δικά σας χωράφια. Εμείς με βάση τους προηγούμενους ε, προϋπολογισμούς και τις προγραμματικές περιόδους έχουμε μάθει να επιτυχάνουμε περισσότερο με πόρους που συνεχώς φθήνουν. Η χρήση των χρηματοδοτικών μέσων στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυξηθεί πάρα πολύ από το 2007, όχι μόνο στη Γεωργία και στις μικρομεσαίες. Στην αρχή της προηγούμενης δεκαετίας ε, έχει είχε αντικατασταθεί αυτό το σύστημα που είχαν επιδοτήσεις οι εταιρείε και περάσαμε σε ένα σύστημα δανείων που πρέπει να αποπληρώνονται. Εμείς ήμασταν ο πρώτος ε, φορέας που διαχειρίστηκε αυτά ήταν πολύ αποτελεσματικά και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ήπεθρο και στην ενέργεια. Ο Επίτροπος Φιλ Χόγκαν μας ζήτησε να αξιοποιήσουμε αυτή την εμπειρία μας από μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να τη μεταφέρουμε και αλλού και στη Γεωργία. Δηλαδή, να χρησιμοποιήσουμε τα κονδύλια που έχουμε και από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και ε, να υπάρχει βιώσιμη δανειοδότηση και επένδυση εκεί. Δεν λέω ότι προσφέρεται αυτό για όλες ε, τις χρηματοδοτήσεις και ε, την γεωργία. Όταν είναι καλά σχεδιασμένα όμως, επιτρέπουν μια μόχλευση και κινητοποιείται και ιδιωτική επένδυση. Δηλαδή, Και κάθε ευρώ από το ΦΕΟΓΑ, το Γεωργικό Ταμείο, ε, πιάνει τόπο. Αυτό το 1 ευρώ δηλαδή ε, πολλαπλασιάζεται και επανέρχεται στην ε, διαχειριστική αρχή ανάλογα με το πώς αποδίδουν τα δάνεια. Αυτό το βλέπουμε και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την ε, αστική ανάπτυξη ε, βλέπουμε να επιστρέφουν αυτά τα κονδύλια, ε, revolving δηλαδή είναι όρος, στην διαχειριστική αρχή. Και αυτό μπορεί να επαναλαμβάνεται και να επανέρχεται είναι σημαντικό να συμμετέχουν και αυτοί οι φορεί για την, να επιλέγονται τα σωστά σχεδιασμένα προγράμματα. Κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνεργαζόμαστε και στη Γεωργία με τις διαχειριστικέ αρχές και θα έλεγα ότι έχει επιτευχθεί κάποια συγκρατημένη πρόοδος, πάντως υπάρχει πρόοδος. 200 εκατομμύρια περίπου έχουμε από ανάληψη υποχρεώσεων από εννέα ε, διαχειριστικές αρχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό θα οδηγήσει αναμένεται σε ένα δις εκατομμύριο δανείων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις γεωργικές. Ακόμα είναι στα σπάργανα αυτή η προσπάθεια στη γεωργία, δεν είναι τόσο προηγμένη όπως σε άλλους τομείς, αλλά βλέπουμε μεγάλο ενδιαφέρον να συγκεντρώνεται από όλο και περισσότερες διαχειριστικές αρχές που διαπιστώνουν ότι δεν έχουν αρκετούς πόρους για να κάνουν τη δουλειά τους. Με βάση τη νέα πρόταση για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, η νομική βάση και το νομικό πλαίσιο θα απλουστευτεί ε, έτσι ώστε ε, να ενισχυθεί η προσπάθεια αυτή χορήγησης ε, κεφαλαίου. Τώρα σκεφτόμαστε να δίνουμε δάνεια όχι μόνο σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και σε φορείς υποδομών και με τρόπο πιο ε, ευέλικτο που θα, ε, θα συνδέεται με την τιμή των πρώτων υλών και των εμπορευμάτων. Αυτό είναι ευαίσθητο ε, τομέα για τι γεωργικέ εκμεταλλεύσει. Ε, Ω ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο με αυξημένη παρουσία σε αυτό το κλάδο, θα πρέπει να εντείνουμε και να συσφίξουμε τους δεσμούς μας και τη συνεργασία μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να ακούμε και τις δικές σας προτάσεις, αλλά μπορώ να σας μιλήσω εξ ονόματος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και να σας πω ότι είμαστε απόλυτα προσιλωμένοι σε αυτή την προσπάθεια για να βοηθήσουμε τον κλάδο να ανταποκριθεί σε δύσκολους καιρούς. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Μακντάουελ. Στι ερωτήσει και παρατηρήσει των Ευρωβουλευτών. 1,5 λεπτό καθένα. παρακαλώ. Ο κύριο Καπούτο πρώτο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να σας πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ για τη σημερινή συνάντηση, διότι ε, δεν συναντά κανεί κάθε μέρα εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η Γεωργία χρειάζεται περισσότερε επενδύσει, έτσι ώστε να παραμείνει σε ανταγωνιστικό επίπεδο, σε παγκόσμια κλίμακα. Βέβαια, πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο, αν λάβει κανεί υπόψη του την ιδιαίτερη δομή που έχουν οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ευρώπη. Πάντως θα πρέπει να υπάρξουν περισσότερες ε, δράσεις, παραδείγματος χάρη στη γεωργία ακριβίας, ε, στην καινοτομία και θα ήθελα να ρωτήσω εσάς να μας πείτε κατά πόσον ενδεχομένως αυτή είναι μία από τις προτεραιότητές σας που λαμβάνετε υπόψη. Όσον αφορά στο μηχανισμό του, της μικροχρηματοδότησης και της δράσης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πρέπει να πω ότι λειτουργείται κυρίως μέσα από ε, ενδιάμεσους. Μην ξεχνάτε ότι τα δάνεια θα πρέπει να χορηγούνται κυρίως ε, για τους νέους και για τις αποκαλούμενες μειονεκτούσες περιοχές. Θέλω να ρωτήσω, αυτός ο μηχανισμός με τους ενδιάμεσους, σε τι ακριβώς βοηθάει και θέλω επίσης να ρωτήσω, θεωρείτε ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλεονέκτημα που προκύπτει από αυτή τη μορφή συνεργασίας. Υπάρχουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις ε, για συγκεκριμένες προτεραιότητες όπως για τους νέους. Αν θυμάμαι, είπατε στην αρχή της ομιλίας σας ότι αντί να εξετάζει κανείς την επιλεξιμότητα των προγραμμάτων, αυτό που εξετάζουν περισσότερο είναι κατά πόσο μια επένδυση είναι οικονομική, εισαγωγικά, αν έχει οικονομική βιωσιμότητα. Θέλω όμως να πω το εξής, ε, ότι αν δεν υπάρχουν ε, οι απαραίτητε εγγύησει, ε, καταλαβαίνετε ότι και οι επενδυτέ δεν θα δείξουν ενδιαφέρον. Άρα δηλαδή είναι πολύ σημαντικό και σε επίπεδο υποδομών κατά κάποιον τρόπο να παρεμβαίνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Μωγά. Σα ευχαριστούμε κύριε Αντιπρόεδρε που μας παρουσιάσετε τους λόγους για τους οποίους η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, έχει την πρόθεση σήμερα πια να πλησιάσει το γεωργικό κλάδο. Γνωρίζετε ότι κατά παράδοση η γεωργία συνήθως ε, ε, λειτουργεί με επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις και όχι τόσο με χρηματοδοτικά μέσα που πρέπει να αποπληρωθούν, να επιστραφούν. Αυτή είναι μεγάλη διαφορά ε, στην προσέγγιση. Γιατί ξαφνικά στρέφεται η ΕΤΕΠ και ενδιαφέρεται για τη Γεωργία και την Ήπεθρο. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, που είναι τράπεζα, θεωρεί ότι η Γεωργία και η Ήπεθρος ε, έχουν στρατηγική σημασία και είναι ε, χώροι καινοτομία και πειραματισμού για το μέλλον. Γι' αυτό στρέφει πια το ενδιαφέρον της και προς τα εκεί. Είπατε και στην παρουσίασή σας ότι τα έσοδα στις ζώνες αυτές είναι χαμηλότερα. Τα εισοδήματα είναι πιο χαμηλά από ό,τι σε άλλες περιοχές. Στις αγροτικές περιοχές είναι πολύ χαμηλότερα τα εισοδήματα. Και μάλιστα η μείωση κατά 25% του μελλοντικού προϋπολογισμού της ε, πολιτικής ε, περιφερειακής ανάπτυξης που είναι το επενδυτικό εργαλείο της ΚΑΠ θα αναγκάσουν και εσάς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βρουν άλλα, μέσα για να στηρίξουν τον κλάδο της γεωργίας γιατί θα χρειαστεί να αναλάβουν περισσότερες δράσεις με λιγότερα κονδύλια και με λιγότερους πόρους. Εν μέρει απαντήσατε στην απορία μου αυτή, αλλά σε ό,τι αφορά τα τοπικά και περιφερειακά σχέδια που θα στηρίξετε, για τι σχέδια και προγράμματα μιλάμε, τι κλίμακα έχουν, θα χορηγήσετε και μικροδάνεια σε τέτοιες περιπτώσεις. Όλα αυτά μας προβληματίζουν ε, με τη νέα στροφή της ΕΤΕ και προς την Ήπεθρο. Ε, κύριε Λοζό, έχουμε μείνει πολύ πίσω στο χρόνο. Παρακαλώ, χρόνου φίδου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε, αυτό το σχέδιο αρρωγής προς το γεωργικό κλάδο είναι ευπρόσδεκτο και το χαιρετίζουμε. Σίγουρα η γεωργία χρειάζεται εξυγχρονισμό, αλλά τώρα το να περάσει μέσα από μια χρηματοδοτική υποστήριξη των ιδιωτών για να ανανεωθεί η πέθρος. Είναι πολύ όμως ε, ε, πενιχρή η συμβολή της ΕΤΕ γιατί σίγουρα είναι καινοτόμα η Γεωργία και θα πρέπει να εξεχρονιστεί και να βοηθηθεί. Αλλά μην ξεχνούμε τους πραγματικούς λόγους που έφεραν σε δυσκολία όλο τον αγροτροφικό κλάδο και την αλυσίδα τη ευρωπαϊκή Ένωση και η υπαγωγή των γεωργικών ε, προϊόντων ε, στου κανόνε κανόνες της παγκόσμιας εμποδίζουν οποιαδήποτε προσπάθεια σταθεροποίηση του κλάδου και οποιαδήποτε προβλεψιμότητα του κεφαλαίου διαχείρισης. Οπότε οι δυσκολίες θα διονυστούν στο μέτρο που αυτές οι διαρθρωτικές αδυναμίες που έχουν διοργανωθεί και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα εξαλειφθούν. Ενώ η κοινωνία ζητά όλο και περισσότερες προσπάθειες από τους γεωργούς υπέρ του κλίματος. Κρίμα λοιπόν που δεν έχουμε περισσότερες επενδύσεις στην έρευνα για πιο βιώσιμα και λιγότερο δαπανηρά φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Ευχαριστώ κύριος Άγνιου. Σας ευχαριστώ κύριε Μακτάουλ πολύ ενδιαφέρουσα η επισκόπηση των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, αλλά δεν mm. αναφερθήκατε καθόλου στο Brexit. Είπατε ότι όταν ε, υπογράφει η συνθήκη της Ρώμης ε, ε, οι χώρες με χρηματοδότησαν την ΕΤΕ και το 2012 πρόσθεσαν νέα κονδύλια. Οπότε υπάρχουν και βρετανικά χρήματα στην ΕΤΕ. Βέβαια δεν επιστρέφεται μερίσματα στο Ηνωμένο Βασίλειο, οπότε θα είναι αχρησιμοποιητό κεφάλαιο, νεκρό κεφάλαιο για το Ηνωμένο Βασίλειο τα χρήματα που έχει δώσει στην ΕΤΕ. Πολλό δε μάλλον που θα χρησιμοποιηθεί για την ε, χρηματοδότηση γεωργικών εκμεταλλεύσεων των 27 χωρών που θα έχουν ανταγωνιστική θέση απέναντι ε, στου στους Βρετανούς παραγωγούς. Δηλαδή ουσιαστικά ο Βρετανός φορολογούμενος ε, χρηματοδοτεί δραστηριότητες εις βάρος των Βρετανών γεωργών. Φαντάζομαι ότι δεν είναι διόλου αμεληταίο το ποσό και σίγουρα το έχετε φροντίσει και το έχετε αξιοποιήσει. Αλλά τι θα γίνει τώρα μετά τον Brexit. 27 δευτερόλεπτα μου έχουν απομείνει, οπότε σας Θέλω παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε και στους υπόλοιπους συναδέλφους να κλείτε το μικρόφωνο τη στιγμή που θα ολοκληρώνουν το 1,5 λεπτό τους. Ευχαριστώ κύριε Σαντρία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και για την παρουσίασή σας. Και εγώ προβληματιζόμουν πολύ. Τι δουλειά έχει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στη Γεωργία. Ε, ε αλλά κατάλαβα όταν αναφερθήκατε ε, ε, σε, περί τίνος πρόκειται πάνω από 25 εκατομμύρια ευρώ ότι είναι οι μεγάλες επιχειρήσεις αυτές. Είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Στο εξή δηλαδή, και εδώ δεν συμφωνούμε όλοι, άλλοι μιλούν για οικογενειακή γεωργία και άλλοι για agro-business. Από το 1992 έχει απελευθερωθεί η Γεωργία και έχει γίνει πιο συγκεντρωτική. Γι' αυτό καταλαβαίνω τώρα που πάει να ε, εμπλακεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και είναι και πολιτική ευθύνη. Αύριο θα έχουμε επιδοτήσεις για την κοινή γεωργική πολιτική που θα πηγαίνουν στην οικογενειακή γεωργία και η Τράπεζα Επενδύσεων θα δανείζει τις μεγάλες επιχειρήσεις, τις αγροδιατροφικές. Όχι, εσείς δεν συνοδεύετε τη γεωργία, αλλά ένα είδος γεωργικής παραγωγής. Για να είμαστε ειλικρινείς, για να ξέρουμε ποια είναι η πραγματικότητα. Από 50 χρόνια μετά την ΚΑΠ, από το 1992, ε, έχουμε επικεντρωθεί στις μεγάλες μονάδες και εσείς εκεί επικεντρώνεστε, μέχρι ποιο βαθμό. Θα στραγγαλίσατε τελείως την Ήπεθρο και δεν θα υπάρχει κάτοικος ε, στην ε, ε, Ήπεθρο, στις πλαγιές και στα βουνά. Δύο μοντέλα λοιπόν, ε, χρηματοπιστωτική ενίσχυση με δάνεια και από την άλλη από τα 500 εκατομμύρια παίρνουμε χρήματα από τους Ευρωπαίους για να δίνουμε λίγα λεφτά στην οικογενειακή γεωργία. Έχουμε διαφορετικούς λοιπόν τύπους γεωργίας και διαφορετικά μέσα ενίσχυσης κάθε φορά. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Κάρθη. Ευχαριστώ και καλώς ήρθατε κύριε Μακδάουελ. Έχω μια ερώτηση για κάτι που είχαμε συζητήσει και κατηδίαν προηγουμένως. Η ΕΤΕ ανήγγειλε ένα λόγο σύστημα για ιδιωτικούς επενδυτές ε, στο τομέα τη δασοκομείας στην Ιρλανδία. Σας εξήγησα τα προβλήματα που δημιουργεί για τους τοπικούς γεωργούς ε, που ε, υπονομεύονται από τις αλλοδαπές εταιρείες που επενδύουν στα δάση της Ιρλανδίας και υποσκάπτουν την βιοπικιλότητα αξιοποιώντας αυτά τα κονδύλια. Η βασική δυσκολία που έχω με το θέμα αυτό είναι ότι προσπάθησα να λάβω πληροφορίες για το ποιος διαχειρίζεται τα κονδύλια αυτά πού ε, γράφονται αυτοί οι επενδυτές κεφαλαίου, ποιο είναι το χαρτοφυλάκιό τους, τα χαρακτηριστικά των ε, κερδοσκόπων και ποιες περιοχές αφορούν. Δεν έλαβα όμως πληροφορίες αυτές παρόλο που σας αναζήτησα. Εδώ μιλούμε κυρίως για δημόσια κονδύλια. Οπότε σας ερωτώ, η ΕΤΕ θα δημοσιεύσει επιτέλους ε, ή θα γνωστοποιήσει αυτές τις πληροφορίες γιατί στην Ελλανδία το 2% της έκθεσης μας καλύπτεται από δάση. Και δεν νομίζω ότι ε, συνάδει τέτοιο με την εθνική δασονομική πολιτική. Και πολύ φοβάμαι ότι η υπόλοιψη της ΕΤΕ θα αμαυρωθεί από τις δράσεις των κερδοσκόπων. Ο κύριος Φλάναγκαν. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ομιλία σας ε, και θέλω να σας πω ότι συναντηθήκαμε συναντή με την Τζιν Φιντζιν που εργάζεται για την ε, τράπεζά σας ε, και σε αυτήν επίσης εκφράσαμε τις ανησυχίες μας. Ε, Διερωτώ με, μήπως μπορείτε σήμερα να μας πείτε Πώς αισθάνεστε, θεωρείτε ότι αυτές οι επενδύσεις ακολουθούν κατά γράμμα την ευρωπαϊκή πολιτική, δηλαδή είναι πράγματι βιώσιμες. Και ρωτάνε οι γεωργοί, αυτοί πώς μπορούν να έχουν πρόσβαση ε, σε αυτές τις επενδύσεις όπως ε, και άλλες εταιρείε. Και όσον αφορά ε, στις χορηγήσεις που ανακοινώθηκαν με τη Rubber Bank 2 εκατομμύρια για τον γεωργικό τομέα. Αυτό είναι καλό, πράγματι πρέπει να γίνουν πολλά για τους γεωργούς, γιατί θεωρούμε ότι πρέπει να τους δίνετε δάνεια, κάνουν πολλά και για το κλίμα, για την βιοπικιλότητα, για την ποιότητα των υδάτων και για την ε, σωστή, ε, σωστό καταμερισμό της ε, ΚΑΠ. Αυτά λοιπόν που προανέφερα είναι σημαντικά. βεβαίω ε, πολύ σωστά επισημάνατε στην αρχή ότι κάνετε επενδύσεις και ότι κάπως τα χρήματα πρέπει να επιστρέφουν σε εσάς. Αλλά αυτή τη στιγμή αν δεν υπήρχαν όλα αυτά που προανέφερα για τους γεωργούς, οι γεωργοί ξέρετε πολύ καλά ότι χάνουν χρήματα. Και ερωτώ, πώς περιμένετε εσείς να σας πληρώσουν ε, αν δεν αλλάξουν οι προϋποθέσεις. Δεν είμαστε πλέον σε μια κατάσταση όπου οι γεωργοί καλούνται να αποπληρώνουν πλήρω τα δάνεια με την έννοια ότι χρησιμοποιείται η μόχλευση, παρεμβαίνει η μόχλευση. Εγώ θέλω να ρωτήσω πώς περιμένετε από τους γεωργούς να αποπληρώσουν τα δάνειά τους. Ευχαριστώ πολύ. Ε, κοιτάξτε, αυτά που άκουσα τώρα μου μοιασαν ότι επενδύεται σε μεγάλη τεχνολογία. Δίνεται τόσα εκατομμύρια σε μια μονάδα για την ε, παστεριοποίηση, ε, σε κάποια άλλη μονάδα επεξεργασία ξύλου. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω τι γίνεται με τους μικρούς που έχουν πρόβλημα πρόσβαση στο κεφάλαιο. Δηλαδή δεν βρίσκουν οι μικροί αυτοί οι γεωργοί τράπεζε για να του βοηθήσουν και δεν αναφέρεται κανένα παράδειγμα. Πού είναι το κατώτατο όριο, ε, από ποιο σημείο και μετά μπορεί κανεί να απευθυνθεί στην Τράπεζα Επενδύσεων. Είπατε ότι ε, δαπανάτε κονδύλια για τη βιοοικονομία. Τι είναι αυτό, τι ακριβώ προάγεται. Η βιοοικονομία είναι τα πάντα. Ε, Μήπω μπορείτε συγκεκριμένα να μα πείτε τι ακριβώ προάγεται και προς, μια κατέ, προς ποια κατεύθυνση εξελίσσονται όλα αυτά. Θα ήθελα να έχω μια εικόνα κατά πόσον πραγματικά επιμερίζετε σωστά τα δάνειά σας ή μήπως σας ενδιαφέρει μόνο να στηρίξετε την τεχνολογία. Γιατί υπάρχουν πολλοί τομείς που δεν έχουν σχέση με την τεχνολογία και χρειάζονται και αυτές δάνεια. Εσείς τι κάνετε, στηρίζετε μόνο την τεχνολογία. Ευχαριστώ κυρία Μαγκίνα, σας ευχαριστώ και ευχαριστώ Άντριο για την παρουσίαση. Ο καθένα κοιτάει τη χώρα του. Και εγώ βλέπω την Ιρλανδία και βλέπω ένα δισεκατομμύριο πέρυσι ε, ε, επενδύθηκε από την τράπεζα σε υγεία, παιδεία, ε, ε, μαζικές μεταφορές, ε, ε κοινωνικές κατοικίες, ε, ΑΠΕ. Και μάλιστα στην ιστοσελίδα της ΕΤΕ αναφέρεται στο ιδίλιο της Ιρλανδίας με το Σέκερς που σαν να μας ενδιαφέρει υπερβολικά αυτό πώς εξασφαλίζεται ε, τη δανειοδοσία στον δοσοκομικό τομέα. Αν μία ομάδα γεωργών ε, ε, ζητήσει ως ομάδα να συνάψει δάνειο, θα μπορέσετε να τη θεωρήσετε μεγάλη κλίμακο επαδίτη, θα πρέπει να περάσει από το κράτο μέλο, τι μηχανισμό θα πρέπει να, να ακολουθήσει και πόσο ε, ευρεία ε, να είναι η ομάδα. Γιατί σίγουρα ο δανεισμό είναι πρόβλημα και όσο χαμηλότερο είναι το κόστο, τόσο καλύτερο. Μπορείτε να μα πείτε πώ θα εξασφαλιστεί τέτοιο χαμηλό δανεισμό. Ευχαριστώ και τώρα θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον κύριο Πίλκε, να σχολιάσει. Γίνεται εν συντομία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μια σύντομη παρατήρηση για τα χρηματοδοτικά μέσα και την ανάπτυξη της υπαίθρου. Αυτό το μέσο έρχεται να συμπληρώσει τις επιδοτήσεις, γιατί χρειάζονται πολλές επενδύσεις και στη γεωργία και γενικότερα στην Ήπεθρο και στις αγροτικές περιοχές και δεν μπορούμε να τα καλύψουμε αυτά μόνο από τις επιδοτήσεις που διαθέτουμε. Γι' αυτό χρειάζονται στοχευμένα, καλά σχεδιασμένα χρηματοδοτικά μέσα για μικρούς και μεγάλους αγρότες. Για να δούμε και την κατάσταση και την πρόσβαση στις, στα κεφάλαια, στα κράτη-μέλη και στις περιφέρειες. Είναι τόσο διαφορετική η κατάσταση κάθε φορά, οπότε χρειάζεται να σχεδιάσουμε καλά τα μέσα για να πετύχουμε τους στόχους πολιτικής. Αυτά που κάνει η ΕΤΕΠ λοιπόν έρχονται να συμπληρώσουν τη δική μας πολιτική. Έχουμε και άλλους εταίρους όπως είναι εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ε, για να έχουμε περισσότερα έργα καλής ποιότητας στην Ήπεθρο. Σας ευχαριστώ. Μάλιστα, Οπότε θα ξαναδώσω το λόγο στον καλεσμένο μας, τον κύριο Μακτάουελ, για να απαντήσει. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Θα προσπαθήσω να απαντήσω όσες περισσότερες μπορώ στο λίγο χρόνο που έχω και θα ζητήσω από τον συνάδελφο τον κύριο Βέρνερ Σμιτ να με συμπληρώσει Καινοτομία και γεωργία. Σίγουρα πολύ σημαντικό ο στόχο τη καινοτομία και στη γεωργία. Και μάλιστα όταν χρηματοδοτούμε μεγάλα επίβολα σχέδια ε, που δεν προωθούνται από, δηλαδή από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα πρέπει να συμβάλλουν και σε άλλου στόχου πολιτική, στι κλιματικέ αλλαγέ ε, και πολύ συχνά και στην καινοτομία. Οπότε δεν χρηματοδοτούμε μόνο ε, ε, μια σημαντική εταιρεία ε, βιοοικονομίας ή σημαντική επιχείρηση τροφίμων, αν δεν ε, παρουσιάσει ένα καινοτόμο σχέδιο με νέες τεχνολογίες ε, και σε ό,τι αφορά την τεχνολογία προϊόντων και την ε, τεχνολογία επεξεργασίας, είτε απορροφώντας τεχνολογία για πρώτη φορά στην Ευρώπη που έχει αναπτυχθεί αλλού ή ε, προτείνοντας μια ρηξικέλευθη τεχνολογία. Το στοιχείο καινοτομία είναι πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να υπάρχει μια συνιστόσα καινοτομία στο σχέδιο που λαμβάνει τη δανειοδότηση. Και αυτό λαμβάνεται, η καινοτομία λαμβάνεται υπόψη και σε επίπεδο χορήγηση κονδυλίων. Θα, θέλουμε να δούμε τι είδου καινοτομίε θα γίνονται στη γεωργία, ώστε να, να ληφθούν υπόψη οι παγκόσμιε προκλήσει. Η ψηφιοποίηση, για παράδειγμα, των γεωργικών εκμεταλλεύσεων είναι τεράστια πρόκληση και σημαντική ευκαιρία. Και δεν μιλάω για την σύνδεση της γεωργικής εκμετάλλευσης με την ευρυζωνικότητα, αλλά κατά μέτρηση της ποιότητας του ε, εδάφους, ε, τη σύνθεση του εδάφους, ε, την παροχή μέσω της ψηφιοποίησης και όλο και μεγαλύτερη αυτοματοποίηση της διαχείρισης της γεωργικής εκμετάλλευσης. Τέτοιου είδους καινοτομίες ε, αναζητούμε ε, και προσπαθούμε με νέες προσεγγίσεις να στηρίξουμε την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Καινοτομία λοιπόν σημαντικό θέμα. Μικροδανισμός επίσης ε, Σημαντικό θέμα. Ο Βέρναρ θα σα μιλήσει για κάποια σχέδια μακρο, μικροδανισμού. Δεν σας εξήγησα και πολύ καλά πώ. ε, ε, χρησιμοποιούμε αυτά τα μικρότερα σχέδια. Μέσω άμεσου δανεισμού, και σας ανέφερα τα 75 εκατομμύρια που είναι το, το κατόφλι, 25, ε, 25 εκατομμύρια. Και όταν περνάμε μέσω από τραπεζικούς μεσάζοντες, ε, φτάνουμε, ε, έχουμε και μέχρι 45.000 ευρώ, που είναι πολύ πιο προσιτό ποσό σε σχέση με τη μέση αγροτική εκμετάλλευση. Και αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε άμεσα, γιατί είμαστε μια τράπεζα σχετικά μικρή, αλλά μόνο με 3.000 προσωπικό, μέτρα το Λουξεμβούργο και δεν μπορούμε να δίνουμε τόσο μικρά δάνεια. Δεν θα ήταν ευχαριστώ πρακτικό ούτε αποτελεσματικό. Οπότε είμαστε αναγκασμένοι να περάσουμε από μεσάζοντες για να παράγουν ε, και να μπορέσουν να χορηγούν μέσω της δικής μας χρηματοδότησης ε, φτηνά δάνεια ή μέσω των εγγύησεών μας. Οπότε έχουμε εταιρικέ σχέσεις με τοπικούς μεσάζοντες και περιφερειακούς μεσάζοντες για να φτάνουν και στα μικρά σχέδια τα πλεονεκτήματα της ΕΤΕ. Τώρα, η συντριπτική πλειοψηφία το, της χρηματοδότησης ε, στη Γεωργία περνάει μέσα από μικρά, ε, περνάει, φτάνει σε μικρούς καλλιεργητές μέσω των μεσαζόντων. Είπαμε το 75% της χρηματοδότησης πάει σε μικρά σχέδια. Λυπάμαι που δεν το διευκρίνησα προηγουμένως. Επίσης έχουμε συγκεκριμένα ειδικά προγράμματα και συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων για τους νέους αγρότες. Έχουμε ειδικά δάνεια για νέους αγρότες μέσω τραπεζικών μεσοζώντων, μέσω της Rubber Bank αλλά και μέσω της Credit Agricole έχουμε ειδικά δάνεια για νέους αγρότες με ιδιαίτερα ελκυστικούς και ευνοϊκούς όρους και τα κριτήρια επιλεξιμότητας ε, ακριβώς ε, ε, λαμβάνουν υπόψη το νερό της ηλικία των αγροτών ή την νέα ε, ε, ενασχόληση με την γεωργική εκμετάλλευση, τη γεωργική δραστηριότητα. Μιλήσατε για την οικονομική ελκυστικότητα και τις μεγάλες τράπεζες. Έχουμε ένα καλό ιταλικό παράδειγμα. Έχουμε συνεργασία με 10 περιφερειακές αρχές στην Ιταλία που χρησιμοποιούν διαρθρωτικά ταμεία από το διαρθρωτικά κονδύλια από το Γεωργικό Ταμείο και τα συγκεντρώνουν σε ένα πουλ ώστε να μπορέσουν 500 εκατομμύρια να ε, δανείσουν σε ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έτσι ε, κατάφεραν να ελαχιστοποιήσουν το κόστος, να έχουν μεγαλύτερη οικονομική αποδοτικότητα και να επιτρέψουν στις τράπεζες να δώσουν μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια δανεισμού, να δίνουν δάνεια με πολύ πιο ευνοϊκού όρου και είναι πολύ καινοτόμο ο τρόπο που συνεργάστηκαν διάφορες Ιταλικέ περιφέρειες για να δώσουν αυτή την εντολή στην ΕΤΕ. Και μάλιστα το επόμενο εξάμεινο θα ολοκληρωθούν οι υπογραφέ ε, με, τις, με του χρηματοπιστωτικού φορεί. Και είναι παράδειγμα προ μίμηση αυτή η Ιταλική συνεργασία των περιφερειών. Ε, με ρωτήσατε πολλά για την πολιτική και τι προτινόμενες μεταρρυθμίσεις ε, στην κοινή γεωρική πολιτική και το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Ε, θα μου επιτρέψετε να αποφύγω τέτοιε απαντήσει ε, σε θέματα πολιτική για την αρμοδιότητα του Κοινοβουλίου και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμεί, ω Ευρωπαϊκή Τράπεζα δεν έχουμε τέτοια αρμοδιότητα. Εμεί εφαρμόζουμε την πολιτική, δεν σχεδιάζουμε την πολιτική. Οπότε σας ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να απαντήσω σε ερωτήματα πολιτικής. Επίσης με ρωτήσατε γιατί κάποιοι γεωργικοί κλάδοι αντιμετωπίζουν δυσκολίε, τι πιέσει υφίστανται από τις παγκόσμιες τιμέ. και προσπαθούμε να στηρίξουμε επιμέρους γεωργικούς κλάδους για να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα μέσω της χρηματοδότησης και να αυξήσουμε την παραγωγικότητα του γεωργικού τομέα για να ανταποκριθεί στις παγκόσμιες προκλήσεις και στις αυξανόμενες παγκόσμιες πιέσεις στις αγορές ε, τέθηκε και μια ερώτηση για το Brexit. Στη συμφωνία αποχώρησης, στο σχέδιο συμφωνίας αποχώρησης που δημοσιεύθηκε το Δεκέμβριο υπήρχε ένα εκτενές κεφάλαιο για την ΕΤΕ με τους όρους της αποχώρησης ε, του Ηνωμένου Βασιλείου από την Τράπεζα Επενδύσεων. Και εκεί αναφέρεται πώς θα επιστραφεί το κεφάλαιο που έχει ε, συμβάλει το Ηνωμένο Βασίλειο, που είναι 3,5 δις και σε ποιο χρόνο θα επιστραφεί. Πάντως είχε ήδη συμφωνηθεί αυτό το κεφάλαιο. Βέβαια, μέχρι την συνολική συμφωνία τίποτα δεν έχει ήδη εκπαιδευτεί, αλλά υπάρχει συγκεκριμένο κεφάλαιο για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την επιστροφή του κεφαλαίου που έχει συνεισφέρει. Για τα διάφορα γεωρικά μοντέλα, σίγουρα ένα από τα νέα στοιχεία της Τράπεζας Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, είναι να εξασφαλιστεί διακριτική ευχαίρεια στον τρόπο που υλοποιούν τους στόχους γεωργικής πολιτικής στα κράτη-μέλη. Εμείς συνεχίζουμε να χρηματοδοτούμε τις πολιτικές των κρατών μελών και τις ε, απαιτούμενε συνεισφορέ του στα επιχειρησιακά προγράμματα. Δεν χρηματοδοτούμε ένα γεωργικό μοντέλο ή ένα γεωργικό σύστημα. Μέσω τη της συγχρηματοδότηση ε, των εθνικών προγραμμάτων πολιτική χρηματοδοτούμε τι εθνικέ επιλογέ ανάλογα με τι εθνικέ γεωργικέ προτεραιότητε σε ό,τι αφορά την ερώτηση για τη δασοκομεία των κυρίων Κάρθη και Φλάναγκαν. Εμείς εφαρμόζουμε την πολιτική, δεν την χαράζουμε ούτε τη σχεδιάζουμε. Η Ιρλανδική κυβέρνηση έχει θεσπίσει τις προτεραιότητες και τις φιλοδοξίες της για το, τους στόχους δασοκάλυψης της Ιρλανδίας και μάλιστα συνάδει με την ευρωπαϊκή πολιτική και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ό,τι κάνουμε σε οποιαδήποτε χώρα και στην Ιρλανδία φυσικά θα πρέπει να λάβει την έγκριση του κράτους μέλους. Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε σε καμία χώρα αν δεν έχουμε την έγκριση της ενδιαφερόμενης χώρας. Και όταν χρηματοδοτούμε μια δοσοκομική ε, επιχείρηση, ε, ρωτούμε τις ε, Ιρλανδικές αρχές που θα εγκρίνουν ή θα απορρίψουν τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Και φυσικά Θέλουμε οι αγροδασοκομικές δραστηριότητες να έχουν μια πιο βιώσιμη προσέγγιση. Και έχουμε ένα ε, ταμείο που βρίσκεται, ένα, χρηματοδοτικό, ένα χρηματοδοτικό, χρηματοπιστωτικό ταμείο που βρίσκεται στην, στο Ηνωμένο Βασίλειο και ε, επενδύει στη δασοκομεία στην Ιρλανδία και έχουμε περάσει από μια προσέγγιση μόνο καλλιέργεια που ίσχυε μέχρι τώρα σε άλλα μοντέλα που ισχύουν περισσότερο σε κεντροευρωπαϊκέ χώρε ή τη Δανία, για να έχουμε μια συνεχή κάλυψη με διαφορετικά είδη ε, ώστε να μην έχουμε ε, ένα τριακοτατή κύκλο που να πρέπει να καθαρίσει πρώτο το δάσος για να ξαναφυτευτεί. Εμείς θεωρούμε ότι και οικονομικά και εμπορικά είναι πιο βιώσιμο αυτό το μοντέλο και τέτοιου είδους ε, δάση με μεγαλύτερη ποικιλία φυτών είναι πιο βιώσιμα και πιο ανθεκτικά. Οπότε λαμβάνουμε υπόψη και περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα όταν χρηματοδοτούμε δασοκομικές ενέργειες και σίγουρα αν πιστεύουμε πιστεύετε ότι η ΕΤΕ χρηματοδοτεί επενδυτές που καταστρατηγούν ε, περιβαλλοντικές ε, ε, διατάξεις οποιαδήποτε άλλη νομοθετική διάταξη Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε μηχανισμό προσφυγών και αν υπάρχουν τέτοιες υπόνοιες παρακαλώ να τις επισημαίνετε υπάρχουν δυνατότητες να διαμαρτυρηθείτε ναι αλλά πού να ενημερωθούμε για τα για τη χρηματοδότηση, μα στην ιστοσελίδα μας έχουμε στοιχεία για όλα τα σχέδια που χρηματοδοτούμε. Όταν επενδύουμε σε ένα ταμείο, έχουμε υποχρέωση διαφάνειας και να αποκαλύψουμε πόσο έχουμε επενδύσει στο συγκεκριμένο ταμείο, ποιον στηρίζουμε και τι προδιαγραφές στηρούνται αυτό το ταμείο. Τώρα, που θα επενδύσει το ταμείο είναι δική του ευθύνη. Πάντως εμείς εξακολουθούμε να είμαστε ε, υπεύθυνοι για την τήρηση των περιβαλλοντικών ε, προτύπων και προδιαγραφών από τους δικαιούχους της επένδυσης. Αυτή την ε, ευθύνη δεν την αποποιούμαστε. Για να απαντήσω τώρα στην ερώτηση της κυρίας Μακίνες σχετικά Σχετικά με τους συνεταιρισμούς, ε, θέλω να πω ότι βεβαίως και συζητάμε πάρα πολλές δράσεις, όχι μόνο στην Ιρλανδία, αλλά και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, σχετικά με τη χρηματοδότηση των ε, συνεταιρισμών και τις επενδύσεις τους. Εμείς έχουμε ήδη χρηματοδοτήσει μία, ένας δύο συνεταιρισμούς στην Ιρλανδία ε, και υπάρχουν και κάποιες άλλες, αιτήσει που τις εξετάζουμε. Πρωτοβουλία Κόσμε. Έχουμε χρηματοδοτήσει κάποιες μικρές επιχειρήσεις στην Ιρλανδία ε, με την θηγατρική μας πέρυσι 330 ε, εκατομμύρια χορηγήσαμε σε γεωργούς μεμονωμένα μέσα από το τραπεζικό σύστημα. Αυτή ήταν η πρωτοβουλία πέρυσι. Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να δώσω και το λόγο στον συνάδελφό μου, τον κύριο Βέρνερ Σμιτ, για να θέσει κάποιες, να απαντήσει κυρίως όσον αφορά την μικροχρηματοδότηση και την ε, καινοτομία. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους σας. Είναι μεγάλη χαρά για μένα που βρίσκομαι εδώ και επιτρέψτε μου ε, να κάνω κάποιες ε, συμπληρωματικές παρατηρήσεις σε αυτά που ήδη καλύφθηκαν πάρα πολύ καλά. Να επενθυμίσω σε όλα τα μέλη της Επιτροπής. Εμείς είμαστε ένας ε, οργανισμός που υπάρχει επειδή υπάρχει ζήτηση. Αν δεν υπάρχει ζήτηση δεν θα μπορούμε και εμείς να επενδύσουμε. Και αν οι όροι που προσφέρουμε δεν είναι καλοί δεν θα μας χρησιμοποιείτε. Ε, απαντώ στη γερμανική ερώτηση. Τα τελευταία χρόνια είδαμε με απόλυτη σαφήνεια μία τάση προς όλο και μεγαλύτερη συμμετοχή μας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αν δηλαδή έχετε την εντύπωση ότι, ότι χρηματοδοτούμε μόνο μεγάλες δράσεις, μεγάλα έργα και τεχνολογία, δεν ισχύει αυτό. Όπως είπε ο συνάδελφός μου, 40.000 ευρώ είναι το κατόφλι και το 2017 το 18% των χορηγήσεών μας ε, διοχετεύτηκε σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 20%, 80% ήταν το ποσοστό και 20% σε μεγάλα έργα. Όλα αυτά τα προγράμματα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας και έχουμε και ένα ειδικό κομμάτι που αφορά τη γεωργία. Όσον αφορά τώρα τη, τα μικροδάνεια, ε, νομίζω ότι αναφέρθηκε ήδη το Ταμείο, το αδελφό μας ε, όργανο και εκεί ε, αυτό το ταμείο χρηματοδοτεί ε, σε μεγάλο βαθμό το γεωργικό τομέα. Αν σας ενδιαφέρει και οι εκλογείς σας να έχουν ε, πρόσβαση σε αυτό το ταμείο προφανώς και υπάρχει μία σειρά ενδιάμεσων αναφέρονται αυτοί στην ιστοσελίδα μας υπάρχουν σε όλα τα κράτη αυτό ήθελα κατ' ουσία να προσθέσω. Αυτά είχα να πω και σας ευχαριστώ πολύ. Για μισό λεπτό παρακαλώ μπορείτε να επανέλθετε. Εάν κάποιος ε, ψηφοφόρος θέλει να έρθει σε επαφή μαζί μου για το ενδεχόμενο παραβίασης ε, του περιβαλλοντικού δικαίου. Για το ότι υπάρχει, παραδείγματο χάρη, μία μονάδα επεξεργασία δασοπονική πολύ κοντά σε ένα ποτάμι. Εσεί πώ το ελέγχετε αυτό. Δηλαδή να επανέλθω εγώ σε εσά να σας το πω και να παρέμβετε εσείς ε, εκ των υστέρων ή μετά ε, με τον τρόπο με τον οποίο αναφέρατε προηγουμένως. Πώς γίνεται, πώς ακολουθείτε όλη αυτή η διαδικασία. Κοιτάξτε, το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι να απευθυνθεί κανείς στον άμεσο χρηματοδότη και να ζητήσει λεπτομέρειες ε, παραδείγματος χάρη όσον αφορά σε αυτή τη συγκεκριμένη δασοκομική μονάδα. Αν όμως υπάρχει μια συγκεκριμένη προσφυγή που ε, αναφέρει ότι έχουμε παρεκκλίνει από τις προδιαγραφές που ισχύουν για μας, αν μας το επισημάνετε αυτό και εμείς ε, θα προσπαθήσουμε να διαπιστώσουμε κατά πόσον πράγματι αυτή η μονάδα είναι ο τελικός αποδέκτης ε, χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Θα το ερευνήσουμε θα τα δημοσιεύσουμε όλα αυτά και αυτή η έρευνα είναι ανεξάρτητη από την τράπεζα. Δηλαδή ισχύει μέσα στην τράπεζα ένας ανεξάρτητος μηχανισμός προσφυγών και μετά, όπως σας είπα, η προσφυγή αυτή δημοσιοποιείται. Άρα δηλαδή μπορούμε να παρακολουθούμε προσφυγές και με μεγάλη μας χαρά το πράττουμε αυτό οποτεδήποτε μας ε, επισημαίνεται συγκεκριμένες ε, παρατυπίες. Σας ευχαριστώ. Οπότε εξαντλήσαμε το θέμα. Έγινε διεξοδική συζήτηση με τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους. Όπως είπα και στην αρχή, ήταν πολύ ανέμενα πολύ καρποφόρα συζήτηση. Αυτό και έγινε και πραγματικά λάβαμε πολύ εμπεριστατωμένες πληροφορίες. Ολοκληρώνουμε λοιπόν το σημείο αυτό της της διάταξης, ευχαριστώντας και πάλι θερμά τους καλεσμένους μας. Και περνάμε με αρκετή καθυστέρηση στο επόμενο σημείο. Περνάμε τώρα στο θέμα της αστικής και περιαστικής γεωργίας. Θα ακούσουμε την παρουσίαση μιας μελέτης ε, την οποία έθεσε το τμήμα πολιτικής Β. Την παρουσίαση θα μας κάνουν η δόκτωρ Ανέτ Πιόρ και ο δόκτωρ Ίγκο Ζασάντα από το Κέντρο Έρευνας Γεωργικού Τοπίου του Κέντρου Λάιμπνιτς. Τις χλιψίες δηλαδή. Επαναλαμβάνω την μελέτη τη ζήτησε το Τμήμα Πολιτικής Β. Η μελέτη θα μας παρουσιάσει την αστική και περιαστική γεωργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, θα γίνει μια ανάλυση της ε, πολυμορφίας του φαινομένου, των χαρακτηριστικών, ε, των πλεονεκτημάτων και των περιορισμών της ε, αστικής και περιαστικής γεωργίας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Εξαρτάται από το πλαίσιο της κάθε χώρας. Και φυσικά εξαρτάται και από τις δυνατότητες που προσφέρει η αγορά. Περιμένουμε την ανάλυση αυτών των πληροφοριών από τους εμπειρογνώμονές μας και τους παρακαλώ να μην ξεπεράσουν τα 20 λεπτά. Παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτέ. Σας ευχαριστούμε για την εισαγωγή κύριε Πρόεδρε. Ονομάζομαι Ίγκο Ζασάντα από το Κέντρο της Λειψίας για την έρευνα γεωργικού τοπίου και η κυρία Ανέτ Πιόρ είναι μαζί μου. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για την ευκαιρία που μας δίνετε να σας παρουσιάσουμε τη μελέτη μας για την αστική και περιαστική γεωργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μας ανέθεσε η Επιτροπή Γεωργίας και που σας έχουμε στείλει. Η παρουσίαση μας θα πραγματευτεί 10 ζητήματα που συνοψίζονται σε τέσσερα θέματα. Γεωργία και αστικό περιβάλλον, κίνητρα, στόχοι και δυναμικό είναι το δεύτερο σκέλος στη αστική περιοχή. Το πολιτικό και θεσμικό περιβάλλον είναι το τρίτο σκέλος και το τέταρτο σκέλος είναι οι συστάσεις για δράση πολιτικής. Πριν περάσουμε στο θέμα της ε, γεωργίας στην αστική και περιαστική ε, περιοχή, να δούμε καταρχήν την χωρική διάσταση αυτού του φαινομένου της αστικής και περιαστικής γεωργίας. Συνήθως ε, πρόκειται για μια γεωργία που ασκεί στις παρυφές μιας πόλης, δηλαδή μιας πόλης που βρίσκεται στο σημείο επαφής μεταξύ της υπαίθρου και της πόλεως του αστικού κέντρου. Αυτή η περιαστική ζώνη χαρακτηρίζεται από πολύ δυναμικά στοιχεία. Υπάρχει μια ισχυρή διαδικασία αστικοποίησης, αύξηση του πληθυσμού, αστιφιλία, αλλά επίσης χαρακτηρίζεται και από μια κατακαιρματισμένη διοικητική κατάσταση. που οδηγεί σε πιέσεις ε, στα αστικά κέντρα, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί και ευκαιρίε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το έχουμε υπόψη όταν μιλούμε για την αστική και περιαστική γεωργία. Δηλαδή, από τη μια έχουμε του γεωργού αυτές αυτέ τι παρυφέ των πόλων που αντιμετωπίζουν ε, σημαντικές πιέσεις γιατί έχουν, ε, ανταγωνίζονται άλλους γεωργούς σε ό,τι αφορά την γη, τη διαχείριση της γεωρικής γης, αλλά και της αγοράς εργασίας και μερικές φορές αντιμετωπίζονται ως ενόχληση, αλλά και δεδομένης της εγκύτητας τους προς τις αγορές καταναλωτή, τις αστικές αγορές, έχουν συγκεκριμένα πλεονεκτήματα. Αυτή η εγκύτητα προς τις αστικές αγορές κατανάλωσης οδηγεί στην ε, δημιουργία και νέων ε, αστικών κοινοτήτων που δημιουργούν μια νέα όθηση προς τη γεωργία. Η γεωργία στις περιοχές αυτές, στις ζώνες αυτές, έχει εφαρμόσει πολλές στρατηγικές προσαρμογής και επιχειρηματικά μοντέλα που θα θέλαμε να σας αναπτύξουμε στη συνέχεια. Καταρχήν, ας ξεκινήσουμε από την γεωργία που γίνεται σε αστικό πλαίσιο. Έχουμε πολύ συγκεκριμένες ε, τεχνολογικές λύσεις, ε, ιδιαίτερες, αλλά και ε, γεωργία που έχουν μια δημοτική ή κοινοτική κατεύθυνση και προσανατολισμό. Γενικώ προσπαθούμε να βρούμε κάποια κοινά χαρακτηριστικά αυτών των γεωργικών πρακτικών που γίνονται συνήθως σε περιορισμένο χώρο, στο αστικό πλαίσιο. Συνήθως οι γεωργοί αυτοί είναι ουσιαστικά κυπουροί, έχουν λαχανόκηπους, δεν έχουν κάποια παιδεία γεωργική, γεωπονική ε, και δεν είναι ιδιαίτερα επικεντρωμένοι στο κέρδος. Χρησιμοποιούν ό,τι χώρους είναι διαθέσιμοι και έτσι έχουν αναπτύξει, ανάλογα με τους περιορισμούς, πολλές καινοτόμες τεχνικές και λύσεις. Γενικώ κάνουμε διάκριση μεταξύ των διαφόρων γεωργικών επιχειρήσεων, ανάλογα με την κλίμακά του. Συνήθω η κλίμακα είναι μικρή. Έχουμε διάφορους ε, παράγοντες και φορεί γιατί δεν έχουμε πάντα κανονικούς γεωργού, κλασικούς γεωργού. Συνήθω έχουμε απλού πολίτε που ασχολούνται με την καλλιέργεια οποροκυπευτικών. Και φυσικά τα κίνητρά τους είναι διαφορετικά και τα ενδιαφέροντά τους είναι διαφορετικά. Έχουμε διακρίνει λοιπόν τρεις τύπους αστικής γεωργίας που είτε επικεντρώνεται στην επιβίωση, είναι γεωργία επιβίωσης, όπως ε, έχει κανείς ένα λαχανόκηπο στον κήπο του. Ε, έχουμε και κοινοτικού λαχανόκηπους με τέτοιες δραστηριότητες καλλιεργητικές, με ένα έντονο κοινωνικό πολιτιστικό προσανατολισμό, έχουμε σχολικούς λαχανόκηπους, διαπολιτισμικούς λαχανόκηπους, αλλά και ε, κάποιες εμπορικές ε, κερδοφόρες λύσεις. Μερικές φορές έχουμε ε, λαχανόκηπους ε, σκεπές ή ε, μανιταροκαλλιέργεια σε υπόγεια. Τώρα, περνάμε από την αστική ζώνη στην περιαστική ζώνη. Βλέπουμε ότι η περιαστική ζώνη έχει περισσότερα κοινά σημεία με τη συνήθη γεωργική πρακτική ή με άλλες ε, αγροτικές δραστηριότητες στην Ήπεθρο. Μια και όμως η περιαστική γεωργία επηρεάζεται από την εγκύτητα με την πόλη, μια και ασκείται στις παρυφές ε, μιας πόλεως, διαπιστώνουμε ότι η περιεστική γεωργία περιλαμβάνει και κάποιες διαφορετικές δραστηριότητες από την κλασική γεωργία στην Ήπεθρο. Γενικώ, και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το έχουμε υπόψη, είναι ότι η προοπτική της γεωργίας σε αυτές τις περιαστικές ζώνες, στις παρυφές των πόλων, έχει αλλάξει πολύ τις τελευταίες δεκαετίες. Στη δεκαετία του 70, για παράδειγμα, όταν ο ΣΑ αναφερόταν στην γεωργία, εμ, την περιαστική που ήταν είχε επηρεαστεί αρνητικά, σήμερα αναγνωρίζει το αναπτυξιακό δυναμικό τέτοιου είδους περιαστικής γεωργίας. Εδώ βλέπουμε τέσσερα διαφορετικά είδη ε, στρατηγικών προσαρμογής που έχουν υιοθετήσει οι, λαχανο, οι, παραγωγοί, οι λαχανόκηποι. Έχουμε ειδικευμένη παραγωγή, σχετικά εντατική παραγωγή οπωροκυπευτικών με καλλιέργειες υψηλής αξίας ή ειδίκευση των υπηρεσιών που απαιτούνται από τους καταναλωτές των πόλων. Όπως έχουμε κάποιες δραστηριότητε υποδρομίας. Ε, επίσης, άλλες τακτικές είναι το, η άμεση διάθεση στην αγορά με τόσο βραχίες αλυσίδες, ε, τροφικές αλυσίδες. Για πολλά χρόνια είχαμε, για πολύ καιρό είχαμε τέτοια φαινόμενα, αλλά βλέπουμε όλο και περισσότερο τους γεωργούς να χρησιμοποιούν ψηφιακές λύσεις για να διαφημίζουν τα προϊόντα τους στους καταναλωτές. Υπάρχει και το θέμα της διαφοροποίησης του γεωργικού εισοδήματος. Είναι το τρίτο είδος περιαστικής γεωργίας. Πολύ δημοφιλές μοντέλο περιαστικής γεωργίας. Εδώ έχουμε τον αγροτουρισμό που ενισχύει κάπως το γεωργικό εισόδημα και η τελευταία μορφή περιαστικής γεωργίας μοιάζει με αυτή της αστικής γεωργίας με έντονο χαρακτήρα κοινότητας, κοινοτικό προσανατολισμό. κάποιοι λαχανόκηποι, ε, συγκομιδή για ίδια κατανάλωση και ούτω καθεξής. Υπάρχει μεγάλη πολυμορφία των είδων γεωργικών δραστηριοτήτων αλλά και των φορέων άσκησης τέτοιων γεωργικών δραστηριοτήτων, των, παρα, των παραγόντων άσκησης τέτοιων δραστηριοτήτων. Και βλέπουμε ε, πόσο διαφορετικά είναι και τα πλεονεκτήματα και τα ωφέλη τέτοιων δραστηριοτήτων. Μερικές τέτοιες δραστηριότητες συμβάλλουν περισσότερο στην δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στην δημιουργία εισοδήματος. Από τη μια, από την άλλη όμως, η αστική και περιαστική γεωργία συμβάλλει και την βελτίωση του περιβάλλοντος, την προστασία του περιβάλλοντος, ε, ε, συμβάλλει στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του κοινού στις περιαστικές περιοχές. Και έτσι συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας ε, φιλο... περιβαλλοντικής υποδομής. Αλλά υπάρχουν και κοινωνικά ωφέλη τέτοιου είδους γεωργίας. Ενισχύει την αποκτήση γνώσεων, την κοινωνικοποίηση, συμμετοχή στα κοινά. Ε, υπάρχουν διαπολιτισμικοί κήποι, ας πούμε, και, και λαχανόκηποι και κοινωνική ε, γεωργία είναι κάτι που πρέπει να τονιστεί, που βλέπουμε συχνά στις πόλεις. Θα σταματήσω εδώ και θα αφήσω τη συνάδελφο. Πρέπει να τονίσω ότι στις αστικές και περιαστικές περιοχές έχουμε ένα είδος γεωργίας διαφορετικό. Έχει έρθει πιο κοντά ε, στα αιτήματα και στη ζήτηση μιας αστικής κοινωνίας η γεωργία και μπορεί να παρέχει πληθώρα ευεργετημάτων και προϊόντων. Και είναι και μια βιτρίνα για το τι ε, μπορεί να γίνει στο μέλλον ε, στην αστική και περιαστική γεωργία. Και θα δώσω το λόγο στη συναδελφό μου. Ε, ε, πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής, με χαρά ε, θα μιλήσω και εγώ τώρα με τη σειρά μου, λέει η δόκτωρ Άνετ Πιόρ. Η πρόσβαση στις ΓΕΣ είναι ένας από τους μεγαλύτερους περιορισμούς, όπως ακούσαμε. Είναι κατακαιρματισμένο ε, το έδαφος, αυξάνονται οι τιμές των ε, αγροτεμαχίων. Έχουμε και νέους φορείς ε, στην Ήπεθρο που δραστηριοποιούνται και εντείνονται οι πιέσει, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οικογένειες. Ε, μπαίνουν νέοι γεωργοί ε, στην εκμετάλλευση, νέα μοντέλα εκμετάλλευσης υιοθετούνται Υπάρχουν κάποιες τεχνολογικές ε, λύσεις που δεν έχουν πλήρως ακόμα αναπτυχθεί. Είναι πολλά ε, πιλωτικά προγράμματα με νεοφυείς επιχειρήσεις, αλλά αυτό έχει μεγάλο επενδυτικό κόστος, ε, το οποίο δεν έχει ακόμα αναπτυχθεί. Επίσης, υπάρχουν περιορισμοί αλλά και απειλές για την αστική και περιαστική γεωργία ακριβώ, διότι δεν έχουμε πολλές γνώσεις για τη Γεωργία και υπάρχουν πολλές γκρίζες ζώνες. Δεν ξέρουμε κατά πόσο συμμορφώνονται απολύτως προς όλες τις ε, διατάξεις για ε, τα λοιπάσματα, για την επεξεργασία των γεών, για την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, τι γίνεται με τους ποιοτικού ελέγχους, ασφάλεια στην εργασία. Ε, φόροι, τέλη, όλα αυτά είναι σε γκρίζε ζώνες, γιατί τα συστήματα είναι άτυπα και όχι επίσημα. Αλλά ακριβώς λόγω αυτού του άτυπου χαρακτήρα και του ανεπίσημου υπάρχει και μεγάλη ευκαιρία. Και έχουμε πολλά παραδείγματα για το πώς ε, βλέπουμε να συμβαίνουν διάφορες αλλαγές και μετασχηματισμοί. Ακριβώς ε, λόγω αυτών των αποκρίσεων στις παγκόσμιες προκλήσεις. Όλο και περισσότερο είναι νέοι αγρότες ε, στην ε, ε, πόλη και πολλές γυναίκες και έχουμε πολύ επιτυχημένα μοντέλα όπως εντάσσονται σε αυτές τις δράσεις οι πρόσφυγες. Η οικονομική ανάπτυξη επίσης έχει μεγάλη επίπτωση. Ας πούμε έχουμε ένα δίκτυο ε, περιαστικών περιοχών ε. Επίσης, ε, είναι οι περιορισμοί, αλλά έχουμε και ευκαιρίες για τα νέα φαινόμενα αστικής και περιαστικής γεωργίας. Από την άλλη βλέπουμε πολλούς φορείς και παράγοντες που έχουν διαφορετικά οικονομικά μοντέλα, πρότυπα παραγωγής και δεν έχουν πάντα ε, ε, σκοπό το κέρδος. Ο κυρίως δεν έχουν το κέρδος. Ε, για ποιο λόγο ακολουθούν αυτό το τύπο γεωργίας και τι στόχους έχουν. Θα πρέπει να το δούμε από την προοπτική του αγρότη αυτό, από τη μια ότι είναι διαφορετικό επιχειρηματικό μοντέλο, νέοι αγρότες, νέοι φορείς και οι αγρότες συνεργάζονται στενά με τους καταναλωτές και οι καταναλωτές τους αναγνωρίζουν ως παραγωγούς, ενώ στην ύπεθρο αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Από την προοπτική ε, των καταναλωτών, οι καταναλωτές είναι δυσαρεστημένοι από το παγκοσμιοποιημένο εμπόριο τροφίμων και θέλουν να έχουν επαφή με τους παραγωγούς, να υπάρχει ίχνηλασιμότητα, εμπιστοσύνη, να, να αλλάζουν επίσης διατροφικές συνήθειες. Επίσης, ε, ο τρόπος με τον οποίο αυτή η γεωργία συνεισφέρει στην ασφάλεια των τροφίμων δεν μπορεί να απαντηθεί, γιατί έχουμε λίγα στοιχεία και όχι αποδείξεις. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι ε, παρακολούθησης και συλλογής στατιστικών στοιχείων, αλλά δεν μας βοηθούν να καταλήξουμε σε ε, συμπεράσματα. Επίσης, σε ό,τι αφορά την επιστήμη δεν είναι το θέμα επιστημιστική ασφάλεια, αλλά επιστημιστική κυριαρχία. Πρόσβαση στην τροφή, ποιότητα της τροφής, ποικιλία ε, των τροφίμων. Ε, υπάρχουν διάφορα ερωτήματα. Ε, υπάρχουν και επίσης ε, οπορώνες σε αστικές και περιφερειακές και περιαστικές περιοχές ή ακόμα και ε, καλλιέργεια οποροκυπευτικών σε ταράτσες και σε στέγες. Ε, κυρίως πρόκειται για τη βιολογική ε, γεωργία. Υπάρχει μεγάλη κοινωνική αποδοχή αλλά υπάρχουν και αντιστάσεις απέναντι σε κάποια συστήματα υψηλής τεχνολογίας τεχνητά. σε ένα θεσμικό πλαίσιο ποιος κάνει τι και πού. Στη μελέτη μας θα βρείτε πολλά στοιχεία περιστατωμένα. Υπάρχουν διάφορα δίκτυα όπως η, πλατφόρμα, MOV πλατφόρμα για τις περιαστικές περιοχές στην Ευρώπη. Είναι το ο Ίδρυμα Ρούαφ από την ε, βιώσιμη αστική γεωργία και συστήματα τροφίμων. Όλα αυτά είναι διασυνδεδεμένοι φορείς και το βλέπουν και από τη σκοπιά των προ, αλλά και της γενικότερης ε, παραγωγής. χρηματοδότηση της έρευνας στα προηγούμενα προγράμματα πλαίσιο και στον ορίζοντα 2020 έχουμε μεγαλύτερη συνειδητοποίηση του φαινομένου και βλέπετε εδώ ότι υπάρχει ευρία γκάμα ε, Ε, ωφελών και πρόσβασης. Και αυτό το ανακλάτε και στην έρευνα. Έρχομαι τώρα ε, σε ε, βασικά επιχειρήματα και διάδραση για την επέμβαση της άσκης πολιτικής. Βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει γεωργική πολιτική και πολιτική αγροτικής ανάπτυξης. Μέχρι τώρα δεν υπάρχουν ειδικά μέτρα για την ενίσχυση αστικής και περιαστικής γεωργίας και εκμεταλλεύσεων υπάρχουν πολύ διαφορετικοί φορείς και επίσης δεν, δεν έχει απασχολήσει μέχρι σήμερα αυτό το θέμα. Ε, έχουν, υπάρχουν διάφορα μέτρα για την γεωργία, την ε, βιολογική γεωργία, υποστήριξη επενδύσεων. Υπάρχει και το θέμα ε, του, του προγράμματος Leader. Έχουν γίνει κάποιες αλλαγές σε σχέση με το παρελθόν ως προς την εξισορρόπηση της ανάπτυξης ε, της υπαίθρου και της αστικής ανάπτυξης. Και τώρα γίνεται και μια δημόσια διαβούλευση για την κοινή γεωργική πολιτική μετά το 2020. Θα πρέπει να σπάσει αυτή η διάκριση ε, αστικών περιοχών και υπαίθρου. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, θα τα βρείτε στην έκθεση, αν θέλετε να το συζητήσουμε στη συνέχεια. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι υπάρχουν πολλοί σημαντικά και πολύ δυναμικά νέα δίκτυα για την παραγωγή τροφίμων στις πόλεις σε τοπικό επίπεδο, σε περιφερειακό επίπεδο. Υπάρχουν ε, δραστηριότητες από την κοινωνία των πολιτών που συνενώνονται ο καθένας από διαφορετική προοπτική, πρόσβαση στην τροφή ή ε, λαϊκές αγορές παραγωγών, σχολικά γεύματα και δημιουργούνται και νέες θεσμικές δομές. Ας πούμε, ε, ε, ε, δίκτυα που συνεργάζονται στα πλαίσια της πρωτοβολίας του Μιλάνου συμμετέχουν πάνω από 160 πόλεις, 80 είναι στην Ευρώπη. Είναι ένα σύμφωνο λοιπόν για την παραγωγή τροφίμων στις πόλεις που έκυψε στο Μιλάνο. Θα πρέπει να προστατεύονται οι γέες αυτές, να είναι αποκλειστικά αφιερωμένες για την παραγωγή ε, τροφίμων. Υπάρχουν και πολλά εμπόδια και φραγμοί. Λείπει η ολοκλήρωση ανάμεσα στα διάφορα θέματα και ανάμεσα στις διάφορες υπηρεσίες ε, των Δήμων. Ε, δεν είναι ξεκαθαρισμένες οι αρμοδιότητες αν είναι εθνικές, τοπικές ή περιφερειακές. Δεν υπάρχει αρκετή ε, συνοχή ανάμεσα στις διάφορες πολυεπίπεδες πολιτικές. Και έρχομαι τώρα στις συστάσεις. Τι βλέπουμε ουσιαστικά. Ότι αστική και περιαστική η γεωργία δεν προσφέρεται για να υπάρξει ξεχωριστή πολιτική ή ένας κλάδος της κοινή γεωργικής πολιτικής. Αλλά εμείς το βλέπουμε ως μοχλό για να επιτευχθεί ένας ευρύτερος σκοπός, μια, να υπάρξει μια ευρύτερη στρατηγική για το μέλλον. Και θα πρέπει ε, διάφορα θέματα να ενσωματωθούν και να, σε μια ολοκληρωμένη προοπτική για όλες αυτές τις περιοχές. Θα πρέπει να ξεπεραστεί ε, αυτό το χάσμα, αυτή η διάκριση ανάμεσα σε αστικές και υπαίθριες περιοχές οι και αγροτικές. Θα πρέπει να υπάρχει μια νέα πολιτική, να συνδεθούν οι πόλεις με την Ήπεθρο. Να ε, υπάρχει και συνεργασία ε, δημοσίου ιδιωτικού τομέα και ε, να δουν οι θύνοντε πώς μπορεί να συνεννοηθεί το κάθε επίπεδο διακυβέρνησης. Αυτό έχει να κάνει και μια, με μια τομεακή ολοκλήρωση και μπορεί να αποτελέσει το δρόμο προς ε, απάντηση στις απαιτήσει κοινωνία, στη ζήτηση. Όλο λέμε στις διάφορες ε, ομιλίες ότι ε, θέλουμε να στραφούμε προς ε, τις επιθυμίες των καταναλωτών και τη ζήτηση των ε, τοπικών κοινωνιών. Αυτά όμως θα πρέπει να αντανακλώνται και ε, στις πολιτικές που ασκούνται και αποφασίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και πρέπει να έχει χαρίσει και μια στρατηγική θεώρηση. Take place. Access to one issue. Η πρόσβαση στη γη είναι ένα θέμα, ένα άλλο θέμα είναι η πρόσβαση στην αγορά. Θα πρέπει να βρεθούν ε, λύσεις ε, και σε ό,τι φορά την κτηματαγορά, την περιαστική. Είναι όλο και πιο σημαντική λοιπόν αυτή η γεωργία και έχει και θετική απόκριση, προσφέρεται πολύ ε, για να διδαχθούμε, για να αλλάξουμε την πολιτική μας. Είναι ένα οικονομικό, δυναμικό φαινόμενο. Ε, είναι πολύ διαφορετικές ε, οι μορφές της γεωργίας, της αστικής και της περιαστικής, αλλά πάντα είναι προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας αλλά βλέπουμε και διάφορους τομείς πολιτικής που πρέπει να συνενωθούν για να έχουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για καλύτερη στόχευση και καλύτερη απόδοση των ε, στόχων της πολιτικής. Um, ε, θα πρέπει λοιπόν όλες αυτές οι στρατηγικές και όλα αυτά τα μοντέλα να συνδυαστούν, να συνενωθούν για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε και πώς θα φτάσουμε στους βιώσιμους στόχους. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μεγαλύτερο σχεδιασμό, συντονισμό των διαφορών τομέων πολιτικής, διάφορα έργα και ε, ε, μέσα και εργαλεία. Αλλά εμεί δεν ζητούμε ειδικού στόχου ή να θεωρηθεί αυτό ένα ξεχωριστό ειδικό κλάδο τη Γεωργία. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ. Και τώρα στρέφουμε στην Ομιγυρή. Πρώτα ζήτησε το λόγο η κυρία Εράνς Καρσία, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι λέγομαι Εράνς. Αυτό είναι το επιθετό μου. Γιατί λέτε Γκαρθία και εγώ θυμάμαι την Ιράτσε Γκαρθία. Μια και είμαστε λίγοι, καλύτερα να, με προφέρετε, να προφέρετε το επιθετό μου το πρώτο, το ΕΡΑΝΣ, για να καταλαβαίνω σε ποιον απευθύνεστε. Ευχαριστώ α, τους δύο εμπειρογνώμονες για την παρουσίαση. Ε, εγώ είμαι γεωγράφος και γνωρίζω πως η μεγάλη σημασία έχει η σύνδεση των αστικών περιοχών με την Ήπεθρο, με τις αγροτικές περιοχές που ίσχυε στο παρελθόν και έχει χαθεί τώρα, καλό θα ήταν να αποκατασταθεί. Εγώ κατάγομαι από μια μικρή περιφέρεια ε, ε, με την πρωτεύουσα της Ριόχα, του Λογρόνιο, που κρατάει ισχυρή περιαστική γεωργία. Και μάλιστα και στη συνοικία μου ε, έχουμε τέτοιες δραστηριότητες που όμως χρησιμοποιούνται όλο και λιγότερο και είναι κρίμα γιατί είναι τόσα τα κοινωνικά, τα πολιτιστικά ωφέλη της αστικής και περιαστικής γεωργίας που είναι κρίμα να μην τα εκμεταλλευτούμε. Όταν όμως μας προτείνετε κάποιες συστάσεις λύσει και το συνδέετε με την κοινή γεωρική πολιτική και το πηγαίνετε προς το πρόγραμμα Leader, αυτό κατά τη γνώμη μου είναι λάθος. Ναι, μεν η εδαφική ε, διάκριση που έχουμε είναι λαθασμένη, θα πρέπει να έχουμε καλύτερη ε, ολοκλήρωση των ε, χώρων των περιφερειών και το ξέρω αυτό ο γεωγράφος, αλλά η Μερικές φορές ε, συνδέουμε την ιδέα της ε, αγροτικής ανάπτυξης ε, μόνο με την Ήπεθρο και την περιορίζουμε στην Ήπεθρο. Τη διαχωρίζουμε από τα αστικά κέντρα για τις αστικές περιοχές. Έχουμε πρωτοβουλία σαν το Urban, που κατά τη γνώμη μου ήταν πολύ σημαντικό μηχανισμός και εργαλείο γιατί εκεί μιλούμε για την αρχιτεκτονική, τον πολιτισμό, την τέχνη. Γιατί να με συμπεριλάβουμε και την περιαστική γεωργία στην εμβέλεια του Urban, του προγράμματος αυτού. Και δεν έχει ίσως, ε, α, δεν δίνει τη δέουσα σημασία σε αυτό το αστικό σκέλος, γιατί συνδέουμε το Urban με πάρκα ή κήπους, αλλά όχι με λαχανόκηπους, ε, με περιαστική γεωργία και τέτοιου είδους ε, δραστηριότητες σαν αυτές που μας παρουσιάσατε δεν, έχετε, δεν είστε και στις γνώμες γνώμης ότι προγράμματα σαν το Urban και γενικώ εργαλεία που είναι πιο προσανατολισμένα προς τις πόλεις θα ήταν πιο ενδιαφέροντες μηχανισμοί για την προώθηση της περιαστικής και αστικής γεωργίας. Συζητούμε τη μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Αν όμως πούμε ότι από την αγροτική ανάπτυξη και από τα σχέδια αγροτικής ανάπτυξης θα πρέπει να προβλεφθούν κονδύλια για την αστική και περιαστική γεωργία, να πω, δεν βλέπω πώς θα μπορέσουμε να το εφαρμόσουμε. Γιατί στοχεύω στην αγροτική ανάπτυξη. Στην Ήπεθρο η Βαρκελόνη δεν έχει πρόσβαση στην αγροτική ανάπτυξη, αλλά στην αστική ανάπτυξη. Και νομίζω ότι θα έχουμε τέτοιε μεγάλε διαφορέ που θα χαθούμε στην πορεία. Καλό θα ήταν να βρούμε άλλους μηχανισμούς για την πρόθεση τέτοιων σχεδίων. Ο κύριο Αντρουέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω για τη μελέτη που μας παρουσιάσατε, που ήταν σαφέστατη και που έθεσαν ένα ζήτημα που δεν είναι καθόλου ίσονος σημασίας. Φυσικά είναι ένα καινούριο φαινόμενο και παίρνει διαστάσεις. Θα πρέπει να οριμάσει κάπως ε, και στο μυαλό μας αυτή η κατάσταση. Αλλά υπάρχει κάποιο στοιχείο της κοινή γεωρικής πολιτικής. Αλλά ίσως ε, είναι απόδειξη και της αποτυχίας της κοινή γεωργικής πολιτικής. Είναι μια πολιτική που εφαρμόζουμε εδώ και 54 χρόνια βέβαια, εντάξει. Ε, πάρτε με κάποιο μέτρο αυτά που λέω, με επιφύλαξη. Δεν υπάρχουν τεράστια, τεράστιες ανησυχίες, αλλά υπάρχει μια απώλεια εμπιστοσύνης ε, ανάμεσα στον καταναλωτή και στο τρόφιμο. Αρχίζει και χάνει ο καταναλωτής την πίστη του, την εμπιστοσύνη του στα τρόφιμα. Γιατί εμείς ε, συμβάλαμε και ενισχύσαμε την αστιφιλία και την αστικοποίηση, γιατί θε... νομίζαμε ότι αυτό ήταν το ιδεώδε σύγχρονο μοντέλο, αλλά προσκρούσαμε σε κάποια εμπόδια, όπως είναι κάποια περιθωριοποίηση ορισμένων συνοικιών και το θέμα το διατροφικό δεν είναι άσχετο με τα προβλήματα της αστικοποίησης. Οπότε σήμερα ο καταναλωτής, κάτοικος των πολλών, που αυτός ε, κανονίζει περισσότερο και είναι πιο απαιτητικό ε, για τα τρόφιμα που αγοράζει. Γιατί αντιλαμβάνεται όλο και περισσότερο ότι τα τρόφιμα επηρεάζουν την υγεία του. Οπότε θέλει εγγύησει ότι τα τρόφιμα που αγοράζει είναι ασφαλή. Και ίσως γι' αυτό αναπτύχθηκε τόσο η αστική και περιαστική γεωργία, γιατί εξασφαλίζει μια εγκύτητα της παραγωγής του τροφίμου με την κατανάλωση. Ξέρει ο καταναλωτής που καλλιεργήθηκαν τα λαχανικά που καταναλώνει και στην ε, μελέτη σας ε, μιλάτε για μια όλο και μεγαλύτερη άνθηση αυτού του μοντέλου. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στι κρατικέ πολιτικέ που εφαρμόσουμε, στι δημόσιε πολιτικέ. Γιατί αν δεν υπήρχε αυτή η ρήξη τη εμπιστοσύνη προ το τρόφιμο, ε, δεν θα είχαμε τόσο αναπτυγμένη αστική και περιαστική γεωργία. Ακριβώ αναπτύχθηκε η αστική και περιαστική γεωργία λόγω τη έλλειψη εμπιστοσύνη του καταναλωτή προ τα γεωργικά προϊόντα. Και εγώ προβληματίζομαι αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον από την άλλη πλευρά αυτό το φαινόμενο, γιατί όπως είπατε και εσείς, μας αναγκάζει στο μέλλον να ε, αντιμετωπίσουμε πιο ολιστικά σφαιρικά την εδαφικότητα, γιατί υπάρχει η αστική διάσταση, η περιαστική και η υπαίθρια, η αγροτική. Γιατί έχουμε όλο και πιο πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές και σίγουρα η περιαστική γεωργία έχει και μια οικολογική αξία και περιβαλλοντική. Θα δούμε πώ θα αποκτασίσουμε την ισορροπία μεταξύ του αστικού ε, πλαισίου και του αγροτικού. Ε, γιατί θα ήταν καταστροφικό να αναπτυχθεί ε, υπερβολικά η αστική και περιεστική γεωργία και να οδηγήσει στην εξαφάνιση της ε, γεωργίας στην Ήπεθρο. Γιατί σε 15-20 χρόνια μπορούμε να έχουμε πιο σαφείς παρατηρήσεις ε. Επίσης, άλλο σημαντικό στοιχείο που επισημάνατε είναι ο κοινωνικός σύνδεσμος, το κοινωνικό στοιχείο. Γιατί βλέπουμε ότι στα αστικά κέντρα υπάρχει ρήξη του κοινωνικού ιστού, του κοινωνικού δεσμού. Οπότε, αν το τρώ, τα τρόφιμα και η παραγωγή με τέτοιο τρόπο αποκαταστήσει, επουλώσει αυτή τον λαβωμένο κοινωνικό σύνδεσμο, είναι πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Σε ό,τι αφορά τις προοπτικές, δεν νομίζω ότι έχουμε κατάλληλε ε, σήμερα δημόσιες πολιτικές για το φαινόμενο αυτό. Θα πρέπει να προσέξουμε γιατί το κίνημα θα επιταχυνθεί και καλό θα ήταν στι μελλοντικέ μας δημόσιες πολιτικές να, λάβουμε, να το λάβουμε υπόψη. Ευχαριστώ. Α, δεν ξέρω αν, ε, αν συνειδητοποίησες πόσο μίλησες. <laughs> Τέσσερα λεπτά, Ερικ. Ενώ κανονικά δύο λεπτά έχει ο καθένας. Κύριε Χόισλινγκ, παρακαλώ, δύο λεπτά. Ε, αφού μιλήσει τέσσερα λεπτά, ε, τώρα νομίζω ότι αυτό μπορεί να ισχύει και για τους επόμενους. Ε, έκανε, άνοιξε τον δρόμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη μελέτη. Αυτή η ενία είναι πολύ σημαντική του πώς όλα αυτά μπορούμε να τα συνδέσουμε με την κοινή ορική πολιτική. Αυτό δεν γίνεται, δεν χρειάζεται κιόλα. Εγώ θα έλεγα ότι κάτι άλλο χρειάζεται για αυτά τα προγράμματα, αλλά όχι η κονδύλια από την ε, κοινή γεωργική πολιτική. Και ξέρετε αυτό που συζητάμε έχει και πολιτιστικό χαρακτήρα γιατί ξέρω στη Γερμανία υπάρχουν ε, πολλές ε, περιοχές οι οποίες θρέφονται από περιεστική γεωργία και αυτό είναι πάρα πολύ καλό γιατί είναι ακριβώς η αντίθετη τάση προς την παγκοσμιοποίηση. Ως εκ τούτου πρέπει να το στηρίξουμε. Γνωρίζω πολλές πρωτοβουλίες ε, που αντιμετωπίζουν προβλήματα και να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Ε, παράδειγμα από τη Φραγκφούρτη. Εκεί το εκτάριο κοστίζει 1,5 εκατομμύριο στη Φραγκφούρτη και τέτοιου είδου προγράμματα κινδυνεύουν διότι τους λένε συνεχώ, ξέρετε η χώρα, με συγχωρείτε, η πόλη επεκτείνεται διαρκώς και γι' αυτό τίθεται θέμα επιβίωσης. Το θέμα είναι πώς ε, αυτή η γεωργία θα ενταχθεί μέσα σε προγράμματα για να μπορεί κανείς και να επενδύσει σε αυτή. Ένα άλλο δευτερεύον πρόβλημα έχει σχέση με τι ε, αστικές ε, πρωτοβουλίε. Εγώ πρέπει να σα πω ότι δεν έχω πάρα πολύ, ε, δεν το βρίσκω πολύ σημαντικό και δεν την έχω σε εκτίμηση αυτή την αντάρτικη γεωργία. Εγώ δεν θα τρεφόμουν από αυτήν. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα σχετικά με τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Και υπάρχει και κάτι άλλο, υπάρχουν προγράμματα παραδείγματος χάρη στις πολυκατοικίες, στην ταράτσα. Ε, αυτά πώς μπορούμε να τα συμπεριλάβουμε στον αστικό σχεδιασμό. Θα βοηθούσε πάρα πολύ. Και τέλος, η χρηματοδότηση αυτών των προγραμμάτων γίνονται γίνεται με ίδια πρωτοβουλία, αλλά τέτοιου είδου προγράμματα έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Και αν όχι, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Εγώ, ξέρετε, καμιά φορά συμφωνώ με το πράσινο λόμπι, κύριε Πρόεδρε. Τυχαίνει και αυτό. Κυρίως όταν μιλάμε για την κατασπατάληση τροφίμων, υπάρχει αυτό στις αστικές περιοχές και μιλάμε ότι ε, είναι πάρα πολύ καλές ε, οι τροφές αυτές και πάνε στα, στα γουρούνια, στους χείρους. Αυτό ε, παλαιότερα γινόταν ε, και ήταν κρίμα. Πάρα πολλοί άνθρωποι άρχισαν να δείχνουν ενδιαφέρον για το τελικά ε, περί τίνος πρόκειται ακριβώς στην Γεωργία. Το θέμα είναι ότι είναι πολύ λογικό να προχωρήσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση, γιατί για δέτε λιγάκι τα ποντίκια που ξέρετε γιατί υπάρχουν, υπάρχουν γιατί πετάνε άλλοι τα τρόφιμα. Αν λοιπόν τα τρόφιμα τα δίναμε στα γουρούνια θα λυνόταν το πρόβλημα και έχω διαπιστώσει το εξή. Όσον αφορά την ε, περιαστική γεωργία, εγώ δεν χρησιμοποιώ συνήθω αυτό τον όρο, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν θέλουμε να κάνουμε κάτι για την περιεστική γεωργία και για την ενεργό γεωργία, ξέρετε φοβάμαι ότι μπορεί να καταλήξουμε και στον ε, βανδαλισμό. Γιατί ε, πολλοί πιστεύουν ότι είναι αστείο το να σκοτώνει κανείς ένα ζώο. Ε, υπάρχει αυτός ο κίνδυνος και παρόλα αυτά ε, παρότι υπάρχει κάποια επιτυχία όπως μας είπατε σε κάποιες διαφάνειες ε, δεν νομίζω ότι ήταν περιεστική η περιοχή ήταν καθαρά γεωργική πάνω σε αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε αυτά που περισσεύουν Ευχαριστώ πολύ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση που μας κάνατε. Το πρώτο που έρχεται στο μυαλό μου με την αστική γεωργία και νομίζω το έπηξαν οι δύο προηγούμενοι ομιλητές είναι το ενδεχόμενο της ε, ρήπανσης. Εγώ ε, δύο χρόνια πέρασα εδώ με τα τρία μου παιδιά και τη γυναίκα μου. Ε, σχεδόν δεν βγαίναμε καθόλου έξω γιατί σε εμά στη δική μας περιοχή τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Και διερωτώ με, έχει γίνει ίσως κάποια μελέτη για δυνάμει ρήπους όπως τα βαρέα μέταλλα παραδείγματος χάρη. Ίσως ε, μπορούμε τους ανθρώπους ε, να τους επαναφέρουμε σε αυτό που τους λείπει από την ικανοποίηση, από ικανοποίηση από την επαγγελματική απασχόληση. Ε, εγώ αυτό που με απασχολεί είναι, σας είπα, η δυνάμη ρήπη. Όσον αφορά τώρα το πότε μπορούν όλα αυτά να γίνουν, ξέρετε, στον Καναδά έχει νομοποιηθεί η κάναβη και η αστική γεωργία δεν είναι κάτι το καινούριο, σίγουρα όχι στον Καναδά. Σήμερα η αστική γεωργία θα, έχει, θα νομοποιηθεί και ελπίζω να νομοποιηθεί η δική μου κυρίως η αστική γεωργία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ και τους καλεσμένους μας για τη μελέτη τους. Ε, πραγματικά όλο και περισσότεροι συμπολίτες μας συνειδητοποιούν ότι μπορούν να παράγουν τρόφιμα όχι μόνο σε κλασικούς αγρούς, ε, στα χωράφια στην Ήπεθρο, αλλά και σε αστικές και περιαστικές ε, ζώνες. Και η μελέτη σας περιλαμβάνει πολλά παραδείγματα και από τη δική μου την πατρίδα, τη Σλοβενία. Και μάλιστα αρχικά ως δήμαρχος και κατόπιν ως υπουργός συμμετείχα στη, σε ένα πρόγραμμα δημιουργίας λαχανόκηπων σε σχολεία. Και μάλιστα φτιάξαμε και πολλούς περιαστικούς λαχανόκηπους με τους πολίτες να παράγουν τα λαχανικά που κατανάλωναν. Είναι σημαντικό να έχουμε υγιεινά τρόφιμα τοπικής παραγωγής, αυξάνοντας έτσι την ε, επάρκειά μας ε, σε τρόφιμα, την επιστημιστική και δημιουργεί διαφορετικούς τρόπους ε, διαβίωσης, ε, Πειράζει τη γαστρονομία, την παρασκευή τροφίμων, τον τρόπο μαγειρέματος, όλη αυτή η συνειδητοποίηση και η επαφή με τα τρόφιμα. Και έτσι μπορούμε να διαπαιδαγωγήσουμε καλύτερα τους νέους που βλέπουν ε, πώς παράγεται ένα τρόφιμο. Γιατί λίγοι έχουν, ε, κατάγονται από χωριό και γνωρίζουν πραγματικά τι μορφή έχουν τα τρόφιμα όταν καλλιεργούνται. Με την περιαστική και αστική γεωργία μπορούμε να αλλάξουμε αυτή την ε, άγνοια και να ε, κάνουμε τους νέους να εξοικειωθούν με τον τρόπο καλλιέργειας. Έχουμε πολλές, ε, πολλά θετικά παραδείγματα όπως την αστική μελισσοκομεία και εγώ έχω ένα παράδειγμα που μία φάρμα σε, περιαστική ζώνη, σε, σε προαστιακή ζώνη απασχολούσε άτομα με αναπηρίες. Τέτοιου είδους ε, παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων σε μια εκμετάλλευση ή παραγωγή λαχανικών σε σχολικούς λαχανόκηπους, σε κοινοτικούς λαχανόκηπους, ε, έχει πολλά πλονεκτήματα γιατί και παράγει λαχανικά τοπικά και δίνει θέση, δίνει δουλειά σε άτομα με αναπηρίες. Δεν νομίζω ότι είναι απειλή για την ύπεθρο τέτοιου είδους φαινόμενα αστικής ε, και περιαστικής γεωργίας, αλλά έχει και πολλά κοινωνικά ωφέλη. Ευχαριστώ. Δεν ζητά άλλο το λόγο. Οπότε θα ακούσουμε τον εκπρόσωπο της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Πίλκε. Παρακαλώ. Thank you, Chairman. Ευχαριστώ για αυτή την ενδιαφέρουσα μελέτη που δείχνει την ποικιλία και την ποικιλομορφία ε, της αστικής και περιαστικής γεωργίας και πόσο συνεισφέρει ιδιαίτερα για την αστική ανάπτυξη. Η μελέτη επίσης δείχνει με πολύ ωραίο τρόπο ότι αυτό το είδος γεωργίας μπορεί να συνεισφέρει στην επαναφορά των δεσμών ε, ε, πόλεων με την Ήπεθρο. Τώρα, όταν πρόκειται για τα απαραίτητα μέσα και εργαλεία που θα προωθήσουν αυτές τις ενέργειες, η μελέτη ήδη ε, αναφέρει τα υφιστάμενα, ας πούμε, η κοινή γεωργική πολιτική, οι επενδύσεις Ε, στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις δεν περιορίζονται μόνο σε αγροτικές περιοχές. Είναι επιλέξιμες και εκμεταλλεύσεις σε περιαστικό περιβάλλον. Υπάρχουν μέσα και εργαλεία. Και επίσης πολύ ωραία μας δείχνει η μελέτη ότι υπάρχει μια στρατηγική ε, που πρέπει να συνενώσει όλα αυτά τα ε, μέσα. Αναφέρετε το πρόγραμμα Leader στη μελέτη σας. Δεν είναι μόνο το Leader. Είναι η όλη έννοια της τοπικής ανάπτυξης που θα προέρθει από την τοπική κοινωνία. Και αντί να τα συζητάμε αυτά σε ένα υψηλό επίπεδο, τα μέσα αυτά θα πρέπει να εξετάζονται ε, σε τοπικό επίπεδο και πώς μπορεί να συνεργαστεί η τοπική κοινωνία. Παράδειγμα, η χωροταξία και ε, η χρήση ε, των γεών και η πολεοδομία είναι κάτι σημαντικό και σε σχέση με αυτό. Προτείνεται να δίνεται ένα πριμ για την εγκατάσταση νέων ε, γεωργών. Δηλαδή ένας νέος αγρότης που θα εγκατασταθεί κοντά σε μια πόλη ε, θα ε, προτιμηθεί από κάποιο νέο αγρότη που θα εγκατασταθεί στην Ήπεθρο. Δεν ξέρω. αν είναι αυτός ε, σε μειονεκτική θέση και δεν είναι ένας αγρότης που ζει σε μια πολύ απομακρυσμένη περιφέρεια που είναι μακριά και από τις αγορές. Πάντως υπάρχει μεγάλο όφελος και για την κοινή γνώμη και θα μπορούσαν θαυμάσια να συνδυαστούν υφιστάμενα μέσα και εργαλεία. Ευχαριστώ. Να πω και εγώ δύο λόγια. Η ανάπτυξη των πόλεων ε, μερικές φορές ε, ε, έγινε σε πολύ, προ, ε, πολύ γόνιμα εδάφη, στα καλύτερα ε, εδάφη. Έτσι χάθηκαν γόνιμα εδάφη για τη Γεωργία. Και είναι μεγάλος ο αριθμός αυτών των κτημάτων. Έχουμε 38 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή ε, εκτάρια που έχουν ε, εξαφανιστεί από τη Γεωργία ε, για να κατοικήσουν 250 εκατομμύρια άνθρωποι. Και μερικές φορές οι περιφερειακές αρχές έκαναν τα στραβά μάτια και έτσι χαρακτηρίστηκαν ως ε, κτήματα ε, για πολεοδόμηση, περιοχές που ήταν είτε γεωργικές είτε δασοκομικές, είτε δάση. Και έτσι θα πρέπει να λάβουμε και την ιστορική αυτή διάσταση. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αστική γεωργία, εφαρμόζεται ένας ιδιαίτερος το... τρόπος παραγωγής. Αλλά αν είναι διαφορετικός τρόπος παραγωγής αυτός της κλασικής γεωργίας, μήπως δημιουργηθεί πρόβλημα ανταγωνιστικότητας. Τι τιμές θα έχουν ε, τα προϊόντα της αστικής γεωργίας, μήπως θα είναι ανταγωνιστικά με τα προϊόντα της κλασικής, της συμβατικής γεωργίας. Επίσης, μιλήσατε για τον παιδαγωγικό χαρακτήρα της γεωργίας ή την ε, άσκηση γεωργικής δραστηριότητας από άτομα με αναπηρία από πιο ηλικιωμένους ε, συμπολίτες. Οπότε εκτός από την ε, παιδαγωγική λειτουργία της αστικής και περιαστικής γεωργίας έχουμε και μια κοινωνική, ψυχαγωγική διάσταση. Αλλά τι άλλη διέξοδο μπορούν να έχουν αυτά τα προϊόντα. Δημιουργούνται σημαντικά ερωτήματα. Σίγουρα από πολλές χώρες όπως η Σλοβενία είχαμε πολύ καλές εμπειρίες, αλλά πολλά εξαρτώνται από την προσέγγιση των τοπικών και περιφερειακών αρχών και την θέση της κοινωνίας των πολιτών. Βέβαια η πλειοψηφία είναι υπέρ ε, είχα πάει στη Ζηρίχη σε ένα Ινστιτούτο που μελετούσε τις ε, κτηνοτροφικές δραστηριότητες και εκεί είχαμε παρατηρήσει τέτοια φαινόμενα. Ενώ στην Βαρσοβία έγιναν πολύ αρνητικά σχόλια για το ότι κυκλοφορούσαν ελεύθερα ζώα σε μια αστική περιοχή. Γιατί μερικέ φορέ εμεί έχουμε την ιδέα ότι οι αγελάδε πρέπει να είναι στην ύπεθρο, όχι να κυκλοφορούν ελεύθερα και γύρω, γύρω από τι πόλει. Οπότε ανακύπτουν και τέτοιε ερωτήσει και εξαρτάται πολλά εξαρτώνται από την ανάγκη που έχει ο τοπικό πληθυσμό, από τα εδάφη που έχουμε διαθέσιμα για την καλλιέργεια. Και το Σάββατο είχα πάει σε ένα φίλο μου που χρησιμοποιεί ένα ιδιαίτερα περίεργο σύστημα με μια κάθετη δομή και σε αυτή την κάθετη δομή που έκανε δημιούργησε το μπαλκόνι του για το πότισμα έβαλε γλάστρες με νερό, με ε, χώμα στην ένα έβαλε ε, μαϊδανό, στην άλλη διάφορα άλλα βότανα. Και σίγουρα τα βότανα είναι πολύ σημαντικά, τα μυρωδικά μάλλον, στη δική του παραγωγή. Και πολύ συχνά έχουμε τέτοιου είδους καλλιέργειες μέσα στις πόλεις. Θα σας δώσω τώρα το λόγο για να απαντήσετε δεν έχουμε πολύ χρόνο γιατί στις 6.30 ακριβώς πρέπει να ολοκληρώσουμε. Um, thank uh, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ε, ερωτήσεις. Ε, πρώτα απ' όλα ε, θα ήθελα να απαντήσω στον βουλευτή κύριο Άντριου. Κοιτάξτε, πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι υπάρχει το φαινόμενο της παραγωγής ε, τροφίμων στις αστικές ε, περιοχές. Εδώ δεν μιλάμε για ποσότητες οι οποίες ε, να μπορούν με οποιονδήποτε τρόπο να αντικαταστήσουν παραγωγή τροφίμων για αστικές περιοχές. Δηλαδή το θέμα δεν είναι να αντικαταστήσουμε κάτι, ούτε να υπάρξει ανταγωνισμός ανάμεσα στις αστικές και τις γεωργικές περιοχές. Θέλω επίσης να υπογραμμίσω αυτά που είπε ο κύριος Πίκ από την Επιτροπή. Δηλαδή η γεωργία στις αστικές και τις περιεστικές περιοχές μπορεί να χρησιμοποιήσει ως γέφυρα ανάμεσα στους καταναλωτές και τις γεωργικές περιοχές. Μπορεί να δείξει το τι μπορεί να προσφέρει η γεωργία ε, σε μια αστική περιοχή και πέρα ε, μόνο από την προσφορά τροφίμων. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Και αυτό που ενδιαφέρει είναι να αποκτήσει κανείς γνώσεις ε, για την παραγωγή τροφίμων σε αστικές περιοχές και να συμβάλλει στην ε, εξέλιξη μιας περιοχής, να δώσει τη δυνατότητα σε άτομα που δεν μπορούν να βρουν απαντήσεις σε μια αστική κοινωνία. Το θέμα δεν είναι θέμα ποσότητας, ε, ούτε θέμα ποιότητας, είναι οι άνθρωποι να έχουν την επιλογή, να είναι περισσότερο αυτάρκης, ε, να μπορούν μόνοι να αποφασίσουν ε, πώς θα τρέφονται, πώς θα τρώνε, περί αυτού πρόκειται. Θα ήθελα να απαντήσω στον κύριο Χόισλινγκ. Αναφερθήκατε στο ρόλο των ε, συμβουλίων Διατροφή ή τροφίμων στις αστικές περιοχές. Ότι έρχεται αυτό ω εξέλιξη. Αν δείτε λιγάκι την κοινωνία των πολιτών, το ρόλο που παίζουν οι κοινωνίε των πολιτών στις αστικές περιοχές, κάτι που δεν υπήρχε στο παρελθόν ε, και τώρα προσπαθούν να καλύψουν τις ανάγκες ε, της αστικής κοινωνίας και αυτό επεκτείνεται και στον πολιτικό τομέα. Αυτό λοιπόν είναι αναμφίβολα κάτι που πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Λέμε ότι θα πρέπει να εξτάσουμε παράλληλα και τις γεωργικές και τις αστικές περιοχές παρότι ο ρόλος αυτών των συμβουλίων δεν περιορίζεται μόνο στην ε, παραγωγή τροφίμων και στη γεωργία. Αναφέρατε το παράδειγμα του πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται οι τεχνικές λύσεις, ε, ε, να αντιμετωπίζονται η παραγωγή τροφίμων σε αστικές περιοχές, όπως παραδείγματο χάρη σε πολυκατοικίες. Στην Ολλανδία γίνονται διάφορα πειράματα και αν το θέμα τίθεται πώς ακριβώς εντασσόμεθα σε ένα αστικό πλαίσιο, διαπιστώνουμε ότι πρέπει και να σκεφτούμε τι μπορεί να είναι η γεωργία. Αυτή τη στιγμή οι πολεοδόμοι στις αστικές περιοχές δεν λαμβάνουν καθόλου υπόψη τους τη γεωργία. Ως εκ τούτου θα πρέπει να υπάρξει ενδεχομένω κάποια αναθεώρηση όλης αυτής της κατάστασης. Και ήθελα επίση και να αναφερθώ ε, σε αυτό που είπε η Ισπανίδα κυρία βουλευτή, η οποία έφυγε το μεταξύ και η οποία αναφέρθηκε στην Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία. Είναι ένα εργαλείο, αλλά είναι και μια ευκαιρία για να ενισχυθούν ε, μειονεκτούσες περιοχές ε, σε αστικές ζώνες. Είναι μια δυνατότητα αυτές να ε, ενσωματωθούν σε γεωργικές περιοχές. Με το leader υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να εξελιχθεί περαιτέρω να χρησιμοποιηθεί ως άλλο ένα εργαλείο για να αντιμετωπιστούν ε, οι ανάγκες ε, της σε κάτω από το αστικό ή το περιεστικό πρίσμα. Mm. εγώ να κάνω λίγα σχόλια στο τέλος και να απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις που άφησες ναι. εσύ. Καταρχήν, ο ε, πρώτος ευρωβουλευτής έθεξε το ειδικό πρόβλημα ότι στα παραδοσιακά συστήματα πολλές δραστηριότητες γίνονται σε μερική απασχόληση γεωργική. Τα απογεύματα, για παράδειγμα, ως παράπλευρη δραστηριότητα. Αυτό θα εξαφανιστεί μάλλον την επόμενη 20 γιατί είναι μάλλον ζήτημα γενιάς. Και τώρα, αν χάσουμε στο μέλλον της γεωργίας, μήπως είναι απειλή η περιεστική και αστική γεωργία. Ναι, αλλά ε, πραγματικά άνθρωποι των πόλεων που δεν έχουν καμία σχέση με τη γεωργία, που έχουν την ευκαιρία να βιώσουν τη γεωργική δραστηριότητα και να δουν πώς ε, λειτουργεί η γεωργία και πώς συνδέεται με τη φύση, είναι θετικό. Και αυτό σχετίζεται με αυτό που επισημάνατε και εσείς. Υπάρχει ένα παιδαγωγικό στοιχείο ε, που ίσως οφείλεται στην έλλειψη εμπιστοσύνη που έχουν οι καταναλωτέ, στην εμπιστοσύνη που έχασαν οι καταναλωτέ στα τρόφιμα επίση ε, ιδιαίτερε γνώσεις που χρειάζονται μερικέ φορέ για τι δραστηριότητε. Αυτέ ή πώς θα μαθαίνει ο κόσμο πώ παράγονται τα προϊόντα, όλη τη διαδικασία για να αντιληφθεί ο καταναλωτή πόσο περίπλοκες διαδικασίε ε, ε, θα πρέπει να, να εφαρμόσει ο γεωργός για να παράγει ένα προϊόν. Όλες αυτές είναι καινούριε γνώσεις που θα βοηθήσουν τον απλό πολίτη να αντιληφθεί τι σημαίνει η γεωργία και να αναγνωρίσει τι αξία έχει και δικαιολογημένα απορροφά ένα μεγάλο τιμά των, ε, του γεωργικού προπολογισμού. Τώρα, για τα, την γεωργία στα κτίρια, σε πολυκατοικίες ή στις ταράτσες στα υπόγεια. Σήμερα ε, δεν λαμβάνονται υπόψη στην οικοδόμηση, στην κατασκευή κτηρίων αυτά τα στοιχεία. Γι' αυτό στο μέλλον θα πρέπει και η μηχανικοί ε, αρχιτέκτονες ε, να καταλήξουν σε τέτοιες λύσεις που μπορεί να μην καλύπτουν όλο το σύνολο της πόλης, αλλά να περιλάβουν και κάποια νέα στοιχεία για την δυνατότητα άσκησης τέτοιας αστικής γεωργίας. Σε ό,τι αφορά τη σπατάλη τροφίμων και τους ε, κύκλους, το θέμα των υπολοιμάτων τροφίμων των οικοκυριών είναι ένα ζήτημα, αλλά σε μερικές προσωμιώσεις που κάναμε ε, βλέπω ότι υπάρχουν απώλειες και στη συγκομιδή και μετά τη συγκομιδή και αυτό πολλές φορές ε, οφείλεται στην συμπεριφορά που έχουμε και στον ορισμό της ποιότητας και στη συνεργασία που έχουμε με γεωργούς ε, βλέπουμε ότι δέχονται ως ποιοτικά κάποια προϊόντα που δεν μπορούν να διαθέσουν στην αγορά, δεν έχουν αγοραία αξία. Και εκεί θα μπορούσαμε να προσδιορίσουμε διαφορετικά τους κύκλους ε, ε, της διάρκειας ε, του τροφίμου και να έχουμε διάφορες φάσεις της αλυσίδας της τροφικής για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα τα υπολείμματα και να μην σπαταληθούν ή να τα χρησιμοποιήσουμε για την παραγωγή βιοενέργειας για παράδειγμα. Επίσης το ζήτημα της μόλης, της ρήπασης του περιβάλλοντος. Μίλησατε για τα βαρέα μέταλλα, κυρίως πρόκειται για μια κατακάθιση από τον αέρα και το θέμα είναι αν βρίσκεται κοντά σε δρόμο κυκλοφορίας ή όχι. Αυτό και αν μπορούμε να το αποφύγουμε, αν μπορούμε να αποφύγουμε αυτού του είδους την ατμοσφαιρική ρήπανση. Δεν έχουμε ακόμη τις απαραίτητες γνώσεις, οι πολίτες που ασχολούνται με αυτά τα θέματα ή χρησιμοποιούν πολλές φορές κομπόστα ή οργανικό λίπασμα σε μεγάλες ποσότητες που δεν ευθυγραμμίζονται με το νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της έλλειψης ειδικών γεωπονικών γνώσεων γιατί ο νομικός ορισμός προβλέπει ότι το οργανικό λίπασμα εφαρμόζεται συμπληρωματικά, ενώ μερικές φορές ε, ε, χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο του, του χώματος από μερικούς ερασιτέχνες τέτοιους γεωργούς. Οπότε έχουμε μεγάλες ποσότητες αζότου. Αλλά μπορούμε να κάνουμε ένα καλύτερο εξορθολογισμό. Γίνεται με καλύτερη ενημέρωση. Τώρα για τους σχολικούς λαχανόκηπους στη Σλοβενία. Ε, συνάδελφοι από τη Λιουμπλιάνα εντόπισαν και ένα άλλο πλονέκτημα. Σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες όπως είναι οι σχολικοί λαχανόκηποι ε, έχουμε μεγάλο ενθουσιασμό και συμβολή του κοινού. Και όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε τώρα λόγω έλλειψης δεδομένων για την ε, σύγκομιδή, για τις καιρικέ συνθήκες, αν αξιοποιήσουμε αυτή την, την επιθυμία, την προθυμία και τον ενθουσιασμό των πολιτών να συμμετέχουν και να συγκεντρώνουν στοιχεία, θα είναι πολύ α, θετικό. Και από τη Σλοβενία είχαμε ήδη ένα καλό παράδειγμα. Ε, μία άλλη ερώτηση έγινε για τα διάφορα εργαλεία και από πού θα πρέπει να προέλθουν τα κονδύλια για να υποστηριχθεί. Ίσως κάποια πριμ για την συνεργασία. Αυτό συζητήθηκε για τη συνεργασία με γεωργούς, με, με συνεταιρισμούς, για να έχουμε συνεργασία μεταξύ γεωργών και καταναλωτών ή άλλων φορέων ε, παραγόντων της αλυσίδας. Υπάρχει δυνατότητα ε, χορήγησης ε, πρημοδότησης. Ένα άλλο θέμα είναι τα αποτελέσματα, τα θετικά αποτελέσματα, τα πλεονεκτήματα της παροχής δημοσίων αγαθών. Και μια τέτοια εργασία, γεωργού και καταναλωτή, μπορεί να έχει και νέες διεξόδους. Αντισταθμίσεις εδαφικού χαρακτήρα για να έχουμε προστασία κάποιων φυσικών χώρων, να έχουμε εξοικονόμηση του εδάφους και αυτό θα μπορούσε να γίνει χάρη στη Γεωργία, στη συνεργασία μάλλον. Και τέλος, η μη επιλεξιμότητα, άλλα δύο λεπτά έχετε λέει ο πρόεδρος, η αστική γεωργία πολύ συχνά λαμβάνει η χώρα σε δημόσια κτήματα. Ε, βέβαια η διαπραγμάτευση γίνεται υπό όρους, αλλά η δημόσ, τα δημόσια κτήματα δεν είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από τον πρώτο και δεύτερο πυλώνα. Επίσης είπατε ότι επειδή οι πόλεις αναπτύχθηκαν σε έφορα εδάφη μπορούν ε, να παράγουν ποιοτικά προϊόντα. Όντως, ε, η περιαστική γεωργία έχει τετραπλάσια διαθέσιμη γη από ό,τι στις αστικές περιοχές και σίγουρα εδώ επηρεάζονται τα πιο έφορα εδάφη. Πάντως η ιδέα που χρησιμοποιείται είναι να στηρίζεται στη φύση. Και εδώ έχουμε πολλές στρατηγικές για παραγωγικές ε, ζώνες σε αστικές ε, περιοχές. Σε συνδυασμό με την προστασία του περιβάλλοντος, προκειμένου να μειωθεί η θερμοκρασία και των πόλεων. Το θέμα είναι πού βρίσκεται όμως, αν είναι καλλιέργεια κοντά σε δρόμο, αν βρίσκεται σε υψηλή επιφάνεια και φυσικά αν είναι η καλλιέργεια δίπλα σε έναν δρόμο υψηλής κυκλοφορίας, σίγουρα τα προϊόντα θα, δεν θα ήταν κατάλληλα προς κατανάλωση. Και έχουμε πολύ γνωστά παραδείγματα μελισσοκομείας στις πόλεις και το τελευταίο παράδειγμα που μας είπατε με την καλλιέργεια στα μπαλκόνια. Έχουμε πολλά ενδιαφέροντα παραδείγματα. Πάντως σας ευχαριστούμε που μας τα παρουσιάσατε. Ευχαριστούμε τους καλεσμένους μας εμπειρογνώμονες. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η μελέτη. Θα μας εμπνεύσει και τις περαιτέρω εργασίες. Είχαμε αρκετό καιρό και για τη συζήτηση μετά και τις ερωτήσεις. Σπάνια έχουμε τέτοια πολυτέλεια χρόνου να μην περιορίζουμε τους αγορητές μας. Ευχαριστώ θερμά τους εμπειρογνώμονες μας και τον συνάδελφο που προετοίμασε και διοργάνωσε την ακρόαση αυτή. Νομίζω ήταν πολύ χρήσιμες πληροφορίες που συγκεντρώσαμε και νομίζω ότι εδώ μπορούμε να βάλουμε ένα τέρμα στην πολύ έντονη μέρα που είχαμε σήμερα με ένα πολύ βαστό πρόγραμμα. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που έμειναν μέχρι το τέλος και να σας ευχηθώ καλό βράδυ. Αύριο εγώ θα πρέπει να δώσω μια διάλεξη, οπότε θα με αντικαταστήσει ο συνάδελφος Δεκάστρο στην Προεδρία. Ευχαριστώ και τους Δερμηνείς Λεπρόεδρος. Καλό σας βράδυ και το επανειδήν.